Uh, good evening, Chairman. It's very good to see you. Um, my point of order, my simply. Ένα διαδικαστικό, Πρόεδρε. Πιστεύετε ότι μπορείτε να πείσετε τις αρχές ε, να χαμηλώσουν λίγο τη θέρμανση, γιατί έχουμε πολύ πολύ ζεστό αέρα, κενό αέρα. Τουλάχιστον να μην είναι τόσο ζεστή η ατμόσφαιρα εδώ πέρα, ο κύριος Μπροκ. Κύριε Τάνοκ, το πρώτο το διεκπαιρεώσαμε, το δεύτερο τώρα το σημείο. Κοιτάξτε, είσαστε συντριπτικό και εγώ είχα συναντηθεί και με άλλου συντριπτικού. Είχα μία αντιπροσωπή από τη Βόρεια Κορέα στο γραφείο μου πριν από λίγο. Και γι' αυτό καθυστέρησα λοιπόν λίγο. Θα το θέσω το θέμα. Οι Ιρανοί προχώρησαν κάπως εσείς. Δεν είναι και για αυτούς καιρός να προχωρήσουν λίγο. Νομίζω ότι και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα επιχείρημα σε ό,τι αφορά και τους ε, Βορειοκορεάτες και το πυρηνικό πρόγραμμα. Να πω ότι θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Άστον και την κυρία Σμίτη για την επιτυχία τους και θα πρέπει πάντα να πούμε ότι λέμε και κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν έχει αντίκτυπο στην εξωτερική πολιτική, αλλά χωρίς την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό δεν θα ήταν δυνατόν. Θα πρέπει να το τονίσουμε λοιπόν αυτό και κάποιες φορές να πούμε ότι έχει και κάποιο θετικό αντίκτυπο η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εξελίξεις. Ο κύριος Τάνοκ με πρόλαβε. Έχετε απόλυτο δίκιο τη ε, της δημοσιότητας ε, που είχε η Λέδη θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, συγγνώμη, ε, και η θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το έργο της και μιλώ ως πολιτικός αντίπαλος. Ο κύριος Μπρόκ, κοιτάξτε, ξέρω ότι είναι για έξι μήνες μόνο και όλο αυτό θα πρέπει να τεθεί υπό αναστολή σε ό,τι αφορά τον εμπλουτισμό πλειδονίου που είναι πολύ επικίνδυνο. Έχουμε λοιπόν μόνο μισό χρόνο να προχωρήσουμε με το όλο θέμα θεωρώ ότι αποτελεί πρόεδρο αυτό. Να προσπαθήσουμε τουλάχιστον αύριο μετά το μεσημεριανό πριν τη συνεδρίαση του διευρυμένου προεδρίου να μας ε, ενημερώσει η Γελίκα Σμίτ για τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει η ενημέρωση σε μια δημόσια ανοιχτή συνεδρίαση. Θα προσπαθήσουμε, εν πάση περιπτώσει, μέχρι αύριο το απόγευμα να μας ενημερώσουν για το θέμα αυτό, για την συμφωνία αυτή, αν συμφωνείτε και εσείς ασφαλώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ενημερώσουμε ότι ο πρόεδρος της Αγκόλα αναγκάστηκε να ακυρώσει το ταξίδι του, άρα και μπορούμε να το διαγράψουμε από την ημερησία διάταξη. Ανταυτού θα ακούσουμε, θα συζητήσουμε την έκθεση της, της κυρίας Ντουρά. Γιατί την συμμετοχή στην ε, αντιπροσωπεία στην ε, Μιανμάρ το Σεπτέμβριο και μια έκθεση του κυρίου Τσέκλε σε ό,τι αφορά την αποστολή για παρατηρήση των εκλογών στο Ταζικιστάν, αν συμφωνείτε. Για το Ιράν τα είπα τα πράγματα που είχα να πω σε ό,τι αφορά τη έγκριση των πρακτικών. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια αντίρρηση ή όχι. Και τώρα περνάμε στην έκθεση πρόοδου για την Αλβανία. Ο κ. Βουλιανίτς είναι εισηγητής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχει ετοιμαστεί το ψήφισμα, όπως έχετε δει, και έχει μοιραστεί. Το έχετε λάβει. Οι τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Οι συμβαστικές τροπολογίες επίσης έχουν κατατεθεί. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους ασκιώδεις εισηγητές και όλα τα μέλη που υπέβαλαν τις τροπολογίες τους και προσπάθησαν να βελτιώσουν το ψήφισμα και να το κάνουν πιο κατανοητό. Όλος ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Doris Πακ, τον κύριο Κούκαν και την κυρία Λίμπορ, που με βοήθησαν πολύ με τις ε, υποδείξεις τους και το προσωπικό της Γραμματείας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις προτάσεις της Επιτροπής. Ευχαριστώ το προσωπικό της ομάδας μου και τους βοηθούς μου που έκαναν την περισσότερη δουλειά και έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να ετοιμαστεί αυτό το ψήφισμα. Το ψήφισμα περιλαμβάνει και κάποιες προτάσεις από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τις ευχαριστώ για αυτές, καθώς και τα αποτελέσματα των προσωπικών μου επαφών που είχα στην Αλβανία, με τις αλβανικές αρχές, με πολιτικούς, με πολιτικούς αντιπολίτευση, με δημοσιογράφους, με μη κυβερνητικέ οργανώσει στην Αλβανία και με Αλβανούς πολίτες που προσπάθησαν να έρθουν ιδιωτικά σε επαφή μαζί τους. Είδατε όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για το ψήφισμα και σας καλώ εσάς όλη την Επιτροπή και τις πολιτικές ομάδες να δεχτείτε την πρόταση ότι το ψήφισμα πρέπει να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα, αλλά και για το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάρει θέση το Κοινοβούλιο πριν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Όποια και αν είναι απόφαση του Συμβουλίου, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει δική τον εξάρτητη και αυτόνομη θέση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώ γι' αυτό θα προτιμούσα και θα σας πρότεινα η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας να γίνει αύριο, εάν είναι δυνατόν. Και αν όχι, στις 5 Δεκεμβρίου. Τόσο ώστε να έχουμε έτοιμη την έκθεση στην Ολομέλεια και μάλιστα στις 9 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Και τα δύο ψηφίσματα είναι καλά. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε το Δεκέμβριο. Όσο πλήρες και αν είναι ένα τέτοιο έγγραφο, δεν μπορεί να τα περιλαμβάνει όλα προφανώς. Έχει δύο στόχους κατά την άποψή μου. Καταρχήν, να βοηθήσει τη χώρα υποστηρίζοντας την έκθεση προόδου της Κομισιόν και να προσφέρει επιπλέον λόγους για το Συμβούλιο, ούτως ώστε να δώσει στην Αλβανία το καθεστώς του υποψήφιου κράτους. Αλλά ο δεύτερος και εξίσου σημαντικός στόχος είναι να συνεισφέρει στη σταθερότητα της περιοχής και να ενισχύσει τη θέση και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, πρόοδοι θα πρέπει να γίνουν σεβαστές και να επιβραβεύονται σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι χώρες για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τις πρόοδους που έχει σημειώσει η χώρα. Η πολιτική οριμότητα που έχει επιτευχθεί είναι σαφής. Πριν από κάνα δύο εβδομάδες χώρα, η κυβέρνηση αρνήθηκε να λάβει ε, χημικά όπλα από τη Συρία προς διάθεση και καταστροφή στην Αλβανία. Δηλαδή, οι Αλβανοί ακούνε τις προτάσεις μας, τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μια τελείως νέα κατάσταση αυτή για τη χώρα. Φυσικά υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να επιληθούν. Μην ξεχνάμε όμως ότι και πολλά άλλα προβλήματα έχουν λυθεί ήδη. Και ότι η υποψηφιότητα, το καθεστώς της υποψήφιας χώρας είναι ένα βήμα ε, στην ενταξιακή διαδικασία και δεν είναι το τελευταίο βήμα προφανώς. Είναι όμως ένα σημαντικό βήμα. Γιατί η χώρα θα είναι με το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων πραγματικά στο μάτι όλων προς παρακολούθηση και θα μας προσφέρει και μηχανισμούς παρακολούθησης και διόρθωσης, ούτως ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλες μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκε η αλβανική κυβέρνηση. Τα ωφέλη θα είναι να ενισχυθούν οι μεταρρυθμίσεις, ε, πιο στενή παρακολούθηση της χώρας και μια επιρροή της χώρας προς τους, στους γειτονές της. Τα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν, κατά τη γνώμη μου, είναι πάνω απ' όλα ένα υψηλότερο επίπεδο πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου στην Αλβανία. Προσπαθούν, αλλά όχι με επαρκή επιτυχία. Η καταπολέμηση της διαφόρας, ένα άλλο πρόβλημα που είναι πολύ εξαρπλωμένη στην Αλβανία, αλλά όχι μόνο εκεί, όπως ξέρουμε, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών. Ε, η καταπολέμηση ε, της βεντέτας και πολλά άλλα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα. Αλλά Πιστεύω ότι με τη βοήθεια οι Αλβανοί, με τη βοήθεια τη δική μας, οι Αλβανοί θα μπορέσουν να επιλύσουν όλα αυτά τα προβλήματα και θα κάνουν τη χώρα τους πιο ευχάριστη. Γιατί όλος ο στόχος αυτής της κατάστασης αυτό είναι, να γίνει η χώρα πιο ευχάριστη, πιο όμορφη. Ε, δεν είναι ο στόχος η ένταξη αυτή καθεαυτή. Αυτός είναι ο στόχος που έχει μια χώρα όταν θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πρώτα θέλω να συγχαρώ τον κύριο Βουλιάνη για το σχέδιο έκθεσης. Είναι μια σωστή έκθεση προς τη σωστή κατεύθυνση. Να πω ότι ομιλώ εξ ονόματος της κυρίας Ντόρις Πακ που είναι σκιώδης εισηγήτρια του ΕΛΚ και δεν μπορεί να παραστεί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων απόψε. Η Αλβανία βρίσκεται σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι προσεκτικό στέλνοντας τα σωστά και δίκαια μηνύματα. Το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές ε, και αναμφίσιμο. Πιστεύω ότι η έκθεση δεν πρέπει να είναι αμφίσιμη. Κατά την τελευταία μας επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στα Τύρανα είχαμε κοινή συνένεση μεταξύ των μελών των διαφορετικών πολιτικών ομάδων υποστηρίζοντας την Αλβανία στην περαιτέρω προσέγγιση της στα βήματα της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης εκτιμούμε το ότι συμφώνησαν πρόσφατα οι σκιώδεις εισηγητές σε μια παρόμοια επικοδομητική προσέγγιση με την, τις συμβαστικές τροπολογίες που κατατέθηκαν για αυτή την έκθεση. Και σε σχέση με την συνάντηση των σχεδόν εισηγητών, ιδιαίτερα με το γεγονός ότι υπάρχει γενική συμφωνία να υποστηριχθούν οι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση πρόοδου. Ζητούμε λοιπόν από το Συμβούλιο να αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί από αυτή τη χώρα, από την Αλβανία και να δώσει στην Αλβανία το καθεστώ υποψήφια χώρα χωρί περαιτέρω καθυστέρηση. Θα πρέπει επίση παρόλα αυτά να γίνει κατανοητό ότι η έκθεση, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί πρέπει να παγιωθεί περαιτέρω και να ε, εμπεδοθεί περαιτέρω η η προώθηση μεταρρυθμίσεων πρέπει να ενταθεί. Διακομματική συνεργασία είναι το κλειδί για την πρόοδο και για την ε, ε, διαδικασία ολοκλήρωσης ε, και για τη δημιουργία ενός θετικού πολιτικού κλίματος που θα είναι επικοδομητικό για την προώθηση των αναγκαίων περαιτέρω μεταρρυθμίσεων. Έτσι λοιπόν, σε σχέση με τις πολιτικές δυνάμεις και την έναρξη της νέας κοινοβουλευτής, περίοδου, κατά την έναρξή της, οι συγκρούσεις και οι διαφορές μας ανησυχούν. Γι' αυτό πρέπει τα μείζωνα πολιτικά κόμματα να δεσμευτούν να βελτιωθεί το πολιτικό κλίμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία. Ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, της ανθρωποεμπορίας, των αρνητικών διακριτικών μεταχειρήσεων, καθώς επίσης και την ανεξαρτησία των κυριότερων θεσμικών οργάνων σε σχέση με την κρατική εξουσία. Όλα αυτά πρέπει να προωθούν. Πρέπει να σημειωθούν συγκεκριμένες πρόοδοι σε αυτό το πεδίο. Αν επιθυμεί η Αλβανία να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις για να προσεγγίσει περαιτέρω την Ευρώπη και υποστηρίζουμε τις τροπολογίες που αντανακλούν αυτό το μήνυμα. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βούλιανιτς για την πολύ καλή του έκθεση. Όσον αφορά την ψήφιση στην Επιτροπή Εξωτερικών, ΑΦΕΤ, η Ντόρις Πακ υποστηρίζει και λέει ότι πρέπει να ψηφίσουμε στην περίοδο συνόδου του Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια, όχι αργότερα. Όταν θέλει η ώρα να ψηφιστεί το θέμα στην Επιτροπή Εξωτερικών, πρέπει να είναι δυνατόν από πλευρά της γραμματείας ε, θεωρούμε να γίνει αυτό και θα το υποστηρίζαμε. Το πιο όμως σημαντικό είναι να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you, Chairman. Let me also first of... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να συγχαρώ και εγώ και να ευχαριστήσω τον Νίκολα Βουλιάνιτς για μια πολύ καλή έκθεση που συνέταξε. Αυτό το ανέφερε ο κύριος Κούκαν πιο πριν. Υπάρχει και είναι αναγκαία συνένεση και από πλευρά της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής μας Εξωτερικών Υποθέσεων και από πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες υπάρχει στεναρή συνένεση όπως εκφράζεται και και από τις συμβαστικές τροπολογίες στις οποίες καταλήξαμε. Όσον αφορά την Αλβανία θα ήθελα και εγώ να τονίσω αυτό το σημείο ώστε να, ε, για να επιτευχθούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαία συνεργασία μεταξύ των μεγαλύτερων κοινοβουλευτικών και πολιτικών ομάδων, ε, πολιτικών ομάδων στην Αλβανία για τις ε, μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προς την προσέγγιση της Ευρώπης από την Αλβανία και αυτό συμπεριλαμβάνει και άλλες εσωτερικές μεταρρυθμίσεις στην Αλβανία. Εγώ και η πολιτική μου ομάδα επίσης θεωρούμε ότι το καθεστώς υποψήφιας χώρας πρέπει να ε, εγκριθεί και να δοθεί στην Αλβανία χωρίς καθυστέρηση. Έκανε τεράστια πρόοδο η Αλβανία με νομοθετικό έργο το οποίο προωθήθηκε. Οι κοινοβουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Υπήρξε μετάθεση, μεταφορά εξουσίας που έγινε με πολύ όμαλο και σωστό τρόπο. Και τώρα πιστεύω ότι είναι η χρονική στιγμή για μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας, τις δεσμεύσεις μας έναντι της Αλβανίας. Να τηρηθεί η διαδικασία ένταξης ε, αξιόπιστη ως διαδικασία. Και όσον αφορά την Αλβανία, για τους πολίτες είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους ψηφοφόρους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, υπάρχουν βέβαια πολλά θέματα, τα οποία πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω, χωρίς καμιά αμφιβολία και στην ενδιάμεση έκθεση αναφέρονται αυτά, δεν θα τα επαναλάβω εγώ εδώ τώρα. Αυτό όμω που είναι σημαντικό είναι να εγκριθεί και να δοθεί το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρα στην Αλβανία. Θα υπάρξουν μήνε και χρόνια μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που θα μπορέσουν αυτέ οι μεταρρυθμίσει να υλοποιηθούν όχι μόνο στα χαρτιά αλλά χειροπιαστά. Όσον αφορά την έγκριση τη έκθεση από πλευρά Ευρωκοινοβουλίου θεωρώ το πιο σημαντικό είναι στην περίοδο συνόδου στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου να το εξετάσουμε και αν θα ψηφίσουμε σε αυτή την εβδομάδα ή όχι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είναι θέμα που πρέπει να αποφασιστεί από πλευρά τη Προεδρία όταν θα υπάρχει η ετοιμότητά μα και θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Το πιο σημαντικό όμω είναι να εγκριθεί στην περίοδο συνόδου στην Ολομέλεια του Στρασβούργου το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um... Κυρία Σχάκε. Ναι, κοιτάξτε. Ταξίδεψα στην Κωνσταντινούπολη για να μιλήσω και να εκφωνήσω μια ομιλία και η κυρία αυτή έκανε conference call, ε, ε διάσκεψη δηλαδή, τη διάσκεψη. Ναι, είσαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Θα μπορούσατε να έχετε γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Πολλά είπαμε για τους, από του συναδέλφου. Πολλά είπαν οι συνάδελφοι. Δεν θέλω να προσθέσω κι εγώ τίποτα από αυτά που είπαν. Να πω μόνο ότι στην παρούσα φάση μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά τις εξέλιξεις στην Αλβανία. Εκ παραλλήλου πιστεύω ότι θα πρέπει και στην Αλβανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκρατηθούμε σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες μας. Ακούμε ότι πολλοί σχολιάζουν ότι η Αλβανία δεν είναι έτοιμη για προσχώρηση. Είναι αλήθεια αυτό, κανείς δεν τον αμφισβητεί. Και πολλά θέματα είναι ακρέμη το οργανωμένο έγκλαμα, η διαφθορά, η διακριτική μεταχείριση, θέματα σε ό,τι αφορά το κράτος, δικαίου, το κράτος δικαίου και την ε, ελευθερία του τύπου και θα πρέπει λοιπόν να έχουμε συγκρατημένες προσδοκίες όπου σε διάφορες ε, περιπτώσεις ε, τα πολιτικά κόμματα λένε ότι ανοίγουν τα βήματα για την προσχώρηση. Φυσικά θέλουμε να κάνουμε κοινή προσπάθεια για τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες. Δεν θέλουμε να υπάρξει πόλωση στο πολιτικό και κοινωνικό τοπίο της χώρας. Του τουλεκτάτως θεωρώ ότι είναι σημαντικό να είμαστε σαφείς για το τι κάνουμε στην παρούσα φάση. Αποστέλουμε ένα μήνυμα. Δείχνουμε ότι περιμένουμε από την Αλβανία να συνεχίσει τις θετικές μεταρρυθμίσεις ως υποψήφια χώρα και ότι πολλά ακόμα θα πρέπει να γίνουν, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να παρέχει αρρωγή προς την Αλβανία σε ό,τι αφορά και την υιοθέτηση του κεκτημένου, το οποίο θα αποτελέσει μακρά διαδικασία, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Κόνολη. Η κυρία Κορνέλησεν, ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές με όλους τους. Θεωρώ ότι είναι η πιο θετική έκθεση που έχουμε ε, καταρτήσει για την Αλβανία σε αυτήν τη θητεία και δικαιολογημένα γιατί επιτέλους υπήρξε ανταλλαγή αν θέλετε της ηγεσία χωρίς μεγάλες τριβές. Άρα ε, υπάρχουν ε, λόγοι για τους οποίους μπορούμε να επενέσουμε τη χώρα αλλά να μην ε, το παρακάνουμε κιόλας. Γιατί η αλλαγή ε, της ηγεσία ε, χωρίς ε, τριβές, χωρίς απεργίες πείνας είναι κατά βάση κάτι το φυσιολογικό. Και οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες προγραμματίζουμε είναι επίσης κάτι το φυσιολογικό. Άρα να μην πλέξουμε και ένα τεράστιο εγκόμιο. Να θυμόμαστε τι έχει γίνει στο πρόσφατο παρελθόν, να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί για το μέλλον. Δεν ξεκίνησε το Κοινοβούλιο τόσο αρμονικά όσο φαίνεται και θα ήθελα πραγματικά η Αλβανία να μας δείξει ένα μητρό άμεμπτο σε ό,τι αφορά και την θετική συνεργασία μεταξύ των κομμάτων. Έχουμε πλέον συμβιβασμούς ισορροπημένους, οι οποίοι αφενός εγκομιάζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί και αφετέρου επικρίνουν, κάνουν συστάσεις για το μέλλον. Πιστεύω ότι τελικά θα είναι καλή η έκθεση και ελπίζω να υπερψηφιστεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Ο τελευταίο σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι θα καταθέσω μια προφορική τροπολογία. Ερευνήσαμε το θέμα, αυτό που με απασχολεί μετά την λήξη της προστασμίας Και τις το θέμα για τις βεντέτες. Το θέμα αυτό, ξέρετε, ότι είναι πολύ σημαντικό στην Αλβανία ο αριθμός των δολοφονιών που συνδέονται με τέτοιες υποθέσεις ε, βεντέτας είναι τουλάχιστον 150 και μιλάμε για τα αναγνωρισμένα περιστατικά πολλά παιδιά, ε, αγόρια δεν μπορούν να βγουν έξω να παίξουν να πάνε στο σχολείο λόγω της βεντέτας και υπάρχει σχετικός ε, μηχανισμός, υπάρχει, υπάρχουν κανόνες από το 2005 και μετά έχει περάσει ένα σχετικό νόμος, ε, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει δραστικά την κατάσταση. Το ΕΛΚ και οι Δημοκράτες θα υποστηρίξουν αυτή την ε, προφορική μου τροπολογία. Ελπίζω να μας υποστηρίξει και ο εισηγητής. Θα την καταθέσω λοιπόν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Uh, thank you, Mr. President. Well, I too... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ συγχαίρω από πλευρά CCR τον, τον εισηγητή για την ισορροπημένη αυτή έκθεση. Η Αλβανία πρόσφατα όντως ε, ήταν πολύ προβληματικό κράτος με πόλωση, όπως είπε και η πράσινη συνάδελφος, και με ε, βία που ξέσπασε πριν από δύο χρόνια. Από την άλλη πρέπει να συγχαρούμε την Αλβανία για την ειρηνική αλλαγή της εξουσίας, αλλά αυτό πρέπει να είναι συνηθισμένη κατάσταση σε, ένα, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η αρχή μιας μακρά διαδικασίας. Έχω υποβάλει δύο τροπολογίες. Ε, πρέπει να υπάρχει ανοχή προς τις σκέφτικες μειονότητες, ειδικά τους χριστιανού χριστιανούς και η ελευθερία προ προς τα διάφορα θρησκεύματα. τη συγχαίρω γι' αυτό. Είναι κάτι ασυνήθιστο στο, στα Βαλκάνια ε, δημιουργεί κάποια διλήμματα ε, εξωτερικής πολιτικής ε, αν ποτέ έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πολύ θετικό είναι ότι έχει μια πολύ μη θρησκευτική παράδοση η Αλβανία. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγους μήνες ε, ήρθε εδώ, ε, ανήκει στη δική μου πολιτική οικογένεια και έμαθε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις να μην προσβάλλει τους γείτονες όπως η Μακεδονία, ε, ζητώντας όπως είχε ζητήσει ο Μπερίσα μια, τη, μεγάλη, τη δημιουργία της μεγάλης Αλβανίας. Ε, αυτό το αναφέρει παράγραφος 17 της έκθεσης. Λυπάμαι που η τροπολογία με 116 για την, τα στοιχήματα δεν έγινε δεχτή από τον εισηγητή, γιατί α, αυτό συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα το οργανωμένο έγκλημα μπορεί να είναι επίσης και μια μη νόμιμη πηγή εισοδημάτων για την κυβέρνηση. Ε, θα πρέπει να το ξαναδούμε. Επίσης η ομάδα μου υποστηρίζει ότι αυτή η έκθεση θα πρέπει να περάσει από την Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαίρω. Ευχαριστώ τον εισηγητή προσωπικά. Γιατί ε, κάτι που δεν ε, είχαμε τα τελευταία χρόνια είναι ένα έτσι πολύ ενεργητικό εισηγητή για την Αλβανία. Η Αλβανία από μόνη της δεν μπορεί να ετοιμάσει μια έκθεση όσο το κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Και παρότι ήρθε καθυστερημένα αυτή η έκθεση, τελικά είναι πραγματικότητα και είναι μια σημαντική συνεισφορά για να κινητοποιήσει και να βοηθήσει την Αλβανία στις προσπάθειές της. Επίσης θέλω να τονίσω τη σημασία των θετικών εξελίξεων στην Αλβανία για την περιφερειακή σταθερότητα. Πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες να δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη δυναμική προς την ένταξη στην Αδριατική ακτή. Και αν στηρίξουμε την Αλβανία μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία, όχι μόνο στην Αδριατική ακτογραμμή, αλλά και η Μακεδονία μπορεί να βοηθηθεί. Χρειαζόμαστε περισσότερα καμπανάκια για τα Σκόπια και νομίζω ότι αυτή η έκθεση πρέπει να αναγνωριστεί ως τέτοια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή την εξαιρετική έκθεση του συναδέφου Βούλιανιτς. Θέλω μόνο δύο πράγματα να τονίσω. Το ένα <clears throat> για το τι ακριβώς ε, σημαίνει αυτή η ε, αλβανική έκθεση για τα, σκόπια, για τα Σκόπια. Δεν είναι κάτι απόλυτα κατανοητό αυτό για μένα. Γιατί και στη Μακεδονία υπάρχουν πρόοδοι. Και αυτά θα τα εξετάσουμε όταν ασχοληθούμε με την έκθεση για τη Μακεδονία που αυτή τη στιγμή δεν είναι στην ημερησία διάταξη. Αυτά που είπε ο συνάδελφος Κάσιν πραγματικά δεν τα κατανόησα, δεν τα κατάλαβα. Το δεύτερο τώρα επ' αυτών είναι ότι για τους συναδέλφους τους πρασίνων. Από τους πρασίνους τονίστηκε η κυβερνητική αλλαγή. Θα θέλω όμως να πω ότι πρόκειται για την έκθεση προόδου που το 2013 συντάχθηκε. Αν όμως δεν κάνω λάθος, αφορά ουσιαστικά μια και αυτό από την Επιτροπή κατά το θέρος ε, συντάχθηκε, ασχολείται με τις πρόοδους το 2012. Όλες αυτές οι πρόοδοι που επετεύχθησαν στην Αλβανία και που δίκαια επενέθηκαν, σε μεγάλο βαθμό το 2012 επετεύχθησαν, πριν λοιπόν από την κυβερνητική αλλαγή. Να μην το ξεχνάμε αυτό, μην δημιουργείται εδώ η εντύπωση σαν να εξαρτάται από το αν κάποια συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι στην εξουσία σε κάποια συγκεκριμένη χώρα και τότε έχουμε θετικότερες εκθέσεις για αυτή τη χώρα. Θέλω να το τονίσω, πρόκειται για μια έκθεση για μεγάλες πρόοδους που επετέλεσε και πέτυχε η Αλβανία το 2012, ήδη κατά την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το χαιρετίζω και εγώ, ότι η κυβερνητική αλλαγή σχετικά ομαλά λειτουργήσε. Εντάξει, ευχαριστώ. Δεν θέλω να συμμετάσχω, δεν θέλω να συμμετάσχω στη συζήτηση ποια είναι και ποιος είναι ο πιο όμορφος και η πιο όμορφη σε όλη τη χώρα. Αλλά σε ένα θέμα έχει ο κύριος Πόσελ φυσικά δίκαιο. Δεν είναι αυτόματο, με, με, δεν γίνονται αυτόματα όλα καλύτερα με μια κυβερνητική αλλαγή. Εντάξει, το πιο σημαντικό που μπορεί και πρέπει να καταδείξει αυτή η Επιτροπή, η Επιτροπή Εξωτερικών, και είναι καλό το ότι ομίλησαν Ολλανδοί και Γερμανοί συνάδελφοι, είναι να δοθεί ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση ότι τώρα έφτασε η ώρα και πρέπει να δοθεί το καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Αλβανία. Το αξίζουν αυτό οι Αλβανοί. Έχουν επιτεύγματα που έχουν επιτελέσει. Αν οπισθοδρομήσουμε πάλι κάνοντας ένα βήμα προς τα πίσω, τότε πάλι θα χάσουμε. Θα χάσουμε κάποτε και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων αυτών. Και πού οδηγεί μια τέτοια κατάσταση μπορούμε να το δούμε αλλού σε σχέση με κάποια άλλη χώρα. Είμαι πεισμένος ότι όλα πρέπει να τα κάνουμε όσα περνούν από το χέρι μας ώστε με τη δική μας κυβέρνηση όταν θα υπάρξει και να το συνηθίσουμε, να συνηθίσουμε για αυτή την κατάσταση να πάνε τα πράγματα καλά και να πάρει το καθεστώς υποψήφιας χώρας ε, η Αλβανία. Ευχαριστώ θερμά, ωραίο θα ήταν, αν και για την παλαιά κυβέρνηση να είναι σαφές λοιπόν ε, σε σχέση και με τους σοσιαλδημοκράτες το τι πρέπει να ε, γίνει και πώς πρέπει να προχωρήσουν. Ναι, εντάξει, γι' αυτό το ανέφερα. Γνωρίζετε καλά τι εννοώ, έτσι. Ήθελα απλά και μόνο να επισημάνω ότι αυτό ε, συναισθάνομαι. Θα έχει τον λόγο ο κύριος Μπέλντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συνάδελφος φεύγει, αλλά θα ήθελα να της πω ότι θα υποστηρίξω πλήρως την ε, ε, τροπολογία της και πριν από κάποια χρόνια είπα και μίλησα στον Επιτροπό σε ό,τι αφορά την ε, φρικτή κατάσταση για τις εκδικήσεις με αίμα στην Αλβανία και ελπίζουμε λοιπόν αυτό να επισέλθει εκ νέου στην έκθεση και να απευθυνθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα ε, επίσης να πω ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η έκθεση και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο οι αλβανικές αρχές σε συνεργασία με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν γιατί πρόκειται για παιδιά τα οποία διδάσκονται στο σπίτι, ζουν μια περιορισμένη ζωή. Πρόκειται λοιπόν για μια αδικία η οποία δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω δύο λόγια. Η Κομισιόν ευχαριστεί ακόμα μια φορά τον κύριο Βουλιάνιτς για την πολύ καλή και ισορροπημένη έκθεση που αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Αλβανία για τις μεταρρυθμίσεις και η Κομισιόν εμένει στη σύστασή της να δοθεί στην Αλβανία το καθεστώς υποψήφιας χώρας. Η Κομισιόν καλωσορίζει όλες τις τροπολογίες των Ευρωβουλευτών προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή υπέρ της, του καθεστώτος υποψηφιότητας. Και στην περίοδο Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο είχαμε, είδαμε την αυξημένη δραστηριότητα της κυβέρνησης ε, σε δράσεις ε, για το κράτος δικαίου. Ο Επίτροπος Φιούλε και ο Πρωθυπουργός Ράμα ε, πρόσφατα ξεκίνησαν ένα διάλογο υψηλού επίπεδου, τόσο ώστε η Αλβανία να παραμείνει έτσι, στοχοθετημένη στην ευρωπαϊκή ένταξη. Στην περασμένη, την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες έγινε η επίσκεψη τριών Αλβανών υπουργών που μίλησαν για το όραμά τους για το μέλλον της Αλβανίας. Και πριν λίγες μέρες, μία διάσκεψη κάτι διαφθοράς υψηλού επίπεδου έλαβε χώρα και μετά από τις συζητήσεις ε, θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα τα συμπεράσματα για τις διώξεις και την, ε, τις των εγκλημάτων έχουμε ειδικέ έρευνε και σε διάφορους πολύ ευαίσθητους τομείς, αστυνομία, εκπαίδευση, τοπική αυτοδιοίκηση, έως και τελωνιακές αρχές, εκεί υπάρχει μεγάλη αστριότητα. Από το Σεπτέμβριο τον, έως τον Νοέμβριο, οι διοκτικές αρχές της Αλβανίας έχουν τι δραστηριότητε τους για να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα. Και επίσης ε, έχουμε γίνει μάρτυρες ε, σαφών στοιχείων ένταξης σε ό,τι αφορά συμπερίληψη πολλών έτσι, ομάδων πληθυσμιακών σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Τους τελευταίους τρεις μήνες, δηλαδή, η Αλβανία ενίσχυσε περαιτέρω τις προσπάθειές τους και τους λόγους που υπάρχουν για να της δοθεί το, το καθεστώς της υποψήφιας χώρας, ο εισηγητής. Λίγες παρατηρήσεις ε, ως απάντηση στα σχόλια των συναδέλφων. Πουθενά δεν μίλησα για μια αλλαγή που προέρχεται από την αλλαγή της κυβέρνησης. Πουθενά δεν γίνεται αυτό και ούτε και στην Αλβανία έγινε. Αυτό που με ανησυχεί στη σχέση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι ότι δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ τους. Αυτός ο διάλογος θα πρέπει να δημιουργηθεί. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να προχωρήσει, να προχωρήσουν τα πράγματα. Η κατάσταση είναι αβίωτη. Για αυτή την προφορική τροπολογία, για τις βεντέτες, δεν την έχω συμπεριλάβει στην έκθεσή μου στο ψήφισμα, παρότι ξέρω το πρόβλημα, όλοι το ξέρουμε. Απλώς δεν ήθελα να βάλω πολλά επιμέρους θέματα σε μία και μόνο έκθεση. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να αναφερθεί σε ένα άλλο, μεταγενέστερο έγγραφο. Μπορούμε να συζητήσουμε αυτή την προφορική τροπολογία. Ανάλογα με τα όσα προβλέπει η διαδικασία πάντως. Επίσης για τη θρησκευτική ανοχή που ανέφερε ο κύριος Τάνοκ. Πριν πάω στην Αλβανία δεν το πίστευα. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση μου επιβεβαίωσαν ότι έτσι συμβαίνει. Είπαν ότι η θρησκεία τους ενδιαφέρει, ότι είναι προσωπική υπόθεση του καθενός και αυτό είναι θαυμάσιο. Πουθενά άλλου δεν το έχω δει στα Βαλκάνια, ούτε καν στην Κροατία. Για τα τυχερά παιχνίδια και το οργανωμένο έγκλημα. Έβαλα μείον στην τροπολογία, το πρόσημο, το αρνητικό στην τροπολογία, γιατί άκουσα ότι σταμάτησαν τα παράνομα τυχερά παιχνίδια, δηλαδή ναι μεν κατάφεραν να τα σταματήσουν, αλλά δεν έπιασαν κανένα εγκληματία, κανένα μαφιόζο, γιατί κάποιος αστυνομικός ενημέρωσε τους εγκληματίες ότι πρόκειται να γίνει αυτή η επιχείρηση της αστυνομίας. Και επομένω δεν θεωρώ ότι αυτό ήταν μια επιτυχία. Εντάξει, ήταν μια καλή προσπάθεια, αλλά δεν στέφθηκε από επιτυχία, γι' αυτό δεν την έβαλα στο ψήφισμα. Όλοι οι εκπρόσωποι όλων των πολιτικών ομάδων είπαν ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε το κείμενο το Δεκέμβριο Δεν επιμένω ότι αύριο πρέπει να ψηφίσουμε και καλά. Ας ψηφίσουμε στις 5 Δεκεμβρίου, εάν δεν μπορούμε αύριο. Δεν θα φέρω αντίρρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά συνάδελφε. Έχουμε και ομάδες που λένε ότι δεν είναι σε θέση αύριο να ψηφίσουν. Και γι' αυτό με τη διαδικασία που ακολουθούμε θα έλεγα θα ψηφίσουμε στις 5 Δεκεμβρίου, ώστε έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε σωστότερα. Ευχαριστώ. Συμφωνείτε με αυτό. Αυτό λοιπόν αποφασίζουμε και αυτό θα γίνει. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Είναι ένα σημαντικό σημείο αυτό. Είναι η έκθεση για τη Σερβία αυτή. Ο κύριος Κάτσιν, συνάδελφε Κάτσιν, έχει τον λόγο. Α, να κάνουμε όμως πρώτα το άλλο. Ναι, εντάξει πρώτα να πάρουμε σε σχέση με το 2006 ε, και μετά ε, το 6 με συγχωρείτε του συναδέφου Κούκαν και μετά θα δούμε τη συνάντηση ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Σερβίας σε σχέση με το Βελιγράδι το Νοέμβριο. Έχετε τον λόγο συνάδελφε να μας εξηγήσετε τα σχετικά. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Λοιπόν, για αυτή την έκθεση μπορώ προσωπικά να σας αναφέρω τη δική μου θέση. 15 Νοεμβρίου είχαμε την πρώτη συνάντηση της ε, Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής στο Βελιγράδι. <clears throat> Μετά άλλους ευρωβουλευτές ξεκινήσαμε <clears throat> αυτό το νέο επίπεδο ε, προσέγγισης ε, με τη Σερβία και το Κοινοβούλιο της Σερβίας ε, διμερώς ε, με βάση την ε, σταθεροποίηση και τη συμφωνία σταθεροποίηση και σταθερο, σταθεροποίησης και σύνδεσης. Συναντήσαμε και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών πέρα από κοινοβουλευτικούς. Πήγαμε στο Βελιγράδι πριν από τις ε, εκλογές στη Μήτροβιτσα, Κόσοβσκα Μήτροβιτσα, στις 17 Νοεμβρίου και δύο εβδομάδες πριν από την διακυβερνητική διάσκεψη που ουσιαστικά ε, είναι η διαπραγμάτευση για την το, ε, το καθεστώς υποψήφιας χώρας προς ένδειξη η Σερβία δεν είναι κάτι το οποίο υπόσχεται, είναι πρακτική εφαρμογή ήδη που έχει ξεκινήσει με μεταρρυθμίσεις που έχουν επιπτώσεις στις λήψεις αποφάσεων. Έχουμε στεναρή άποψη ότι κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που διαρκώς συνιστούμε στη Σερβία εδώ και δεκαετίες θα έχουν μια ευκαιρία τώρα να υλοποιηθούν και να λάβουν χώρα. Κάποιες παρατηρήσεις η οικονομία της Σερβίας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι εφημισμός αυτό. Και μάλιστα το δημόσιο χρέος ταχύτατα αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω και των επιδοτήσεων και ενισχύσεων από πλευρά τη κυβέρνηση. Υπάρχει τεράστια ανεργία στον δημόσιο τομέα. Μας ενημέρωσαν και μας είπαν ότι οι ριζοσπαστικές περικοπές όσον αφορά την πολιτική έχουν οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση και έχουμε την εντύπωση ότι είναι έτοιμη η ηγεσία να αντιμετωπίσει την δυσαρέσκεια αυτή από πλευρά των ψηφοφόρων των πολιτών μέσω αυτών των μεταρρυθμίσεων. Και εδώ πρέπει να το δούμε αυτό σε σχέση με τις ε, υποθέσεις και εικασίες ε, για πρώιμες εκλογές. Δεν υπάρχει καμία πίεση μεταξύ των ηγετών να γίνουν πρόορες εκλογές. Μια και έχουν συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική σταθερότητα στη Σερβία είναι μεγαλύτερη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα της περιοχής αυτής. Για το κοσυφοπέδιο που έτυχε ιδιαίτερης προσοχής ε, στη συζήτηση λόγω των εκφοβιστικών ε, εκστρατιών στην Μήτροβίσα επανελήφθησαν εκλογές ε, κατά την 17η Νοεμβρίου. Έγινε λοιπόν επανάληψη και έγινε προσπάθεια από πλευρά των σερβικών αρχών ε, να ηρεμήσουν τα πράγματα. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη όμως στο πρώτο γύρο των εκλογών. Και ακούσαμε και είπαμε και εμεί στους εταίρους μας ότι δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να δεχθούμε επισκέψεις αξιωματούχων της Σερβίας με παραστρατιωτικές ε, στολές ε, ε, στο κοσυφοπέδιο, διότι αυτό επιδεινώνει την κατάσταση. Σήμερα η κατάσταση φαίνεται να είναι καλύτερη, καλύτερη. και εγώ <clears throat> κρίνω σχετικά θετικά την στάση των σερβικών αρχών όσον αφορά την εξομάλυση των σχέσεων με την Πρίστινα. Η καταπολέμηση της διαφθαράς και του οργανωμένου εγκλήματος εντείνεται <clears throat> και είναι κάτι το οποίο ε, εκτιμούμε. Δεν θέλω να υπησέφθω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα μόνο μια κρίσιμη παρατήρηση να κάνω. Η διαδικασία αυτή έχει τύχη προτεραιοτήτων και ιεραρχήσεων που είναι δεδομένες. Ωστόσο, η μάχη δεν διεξάγεται μέσα στα υφιστάμενα θεσμικά όργανα και στο νομικό πλαίσιο. Έχει μια εκ των χαρακτήρα και μια ε, έντονη πολιτική χρειά. Αυτό μπορεί ίσως αρχικά να υπαρκούσε ή να υπαρκεί. Μακροπρόθεσμα όμως ε, υπονομεύει την έννοια του κράτους δικαίου και το πώς οι πολίτες θα ήθελαν να προχωρήσει και βλέπουν τα πράγματα πώς θα ήθελαν να προχωρήσουν. Και σε σχέση με την παρακολούθηση σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ε, για ένταξη της Σερβίας πρέπει να εκπαιδευτούν ε, οι πολίτες της Σερβίας και να γνωρίσουν τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορέσουμε ε, με επιδέξιο τρόπο να το κάνουμε αυτό σε σχέση με τα δικαιώματα της αρχής επικουρικότητας και των εθνοτικών δικαιωμάτων. Εθνοτικών δικαιωμάτων έναντι ενός κρατικού κεντρικού σχεδιασμού ή κράτους. Και σε σχέση με τις αντιπροσωπείες του Ευρωκοινοβουλίου προς τη Σερβία υπό Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Επιτροπή Περιβάλλοντος που θα μεταβούν στη Σερβία. Σαν συνέπεια τούτου η δική μας ε, ε, Επιτροπή προσπάθησε να μην ε, δημιουργήσει επικαλύψεις σε σχέση με θέματα άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βελιγράδι καθώς επίσης και την υποστήριξη και συνδρομή που μας παρήχαν. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Okay, I have not finished. I uh, uh, δεν ολοκλήρωσα. Θα σας πω κάποια ανέκδοτα για να γεμίσουμε το χρόνο μέχρι να επιστρέψει. Λοιπόν, πολύ καλά. Νομίζω ότι λογικό είναι ο επόμενος αγορητής να είναι ο Γιώργο Κάτσιν. Και έτσι λοιπόν έτσι θα προχωρήσουμε. Παρακαλώ. Thank you, ευχαριστώ κύριε Κούκαν. Θα συνεργαστούμε και συνεργαζόμαστε διαρκώς. Από την αρχική εξέταση της εκθεσής μου για τη Σερβία, η πρώτη χώρα, οι πρώτες εκλογές, ε, εθνικές ε, εκλογές έλαβαν χώρα στη Σερβία και η προσέλευση ήταν ε, αναπάντεχα υψηλή στα περίκλειστους περιοχές στους στήλακες Στη Μητροβίτσα στις 7 Νοεμβρίου δεν παρουσιάστηκαν ευτυχώς επεισόδια. Αυτές οι εκλογές ήταν πάρα πολύ σημαντικές για να θεωρηθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια που έθεσε το Συμβούλιο στην διακυβερνητική διάσκεψη. Και έτσι λοιπόν Πιστεύω ότι η διακυβερνητική θα πρέπει να λάβει χώρα το Δεκέμβριο φέτος και θα καταδείξει τη δέσμευση έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διαδικασία της προσχώρησης. Ε, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να πραγματοποιηθεί αυτή η διακυβερνητική Πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν για να ομολοποιηθεί η σχέση μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου, αλλά τώρα οι Σέρβοι ηγέτες φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν το διάλογο με την Πρίστινα και να γυρίσουν σελίδα στα σφάλματα του παρελθόντος. Η εφαρμογή της συμφωνίας του Απριλίου και οι μετέπειτα συμφωνίες θα πρέπει να παρακολουθούνται με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον στις πρώτες φάσεις των συζητήσεων προσχώρησης. Η δικαστική μεταρρύθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά παραμένει ένα δύσκολο εγχείρημα. Οι εισαγγελείς εργάζονται υπό μεγάλη πίεση και εξακολουθούν να αποτελούν από τους πιο αδύναμους ε, κρίκους στην καταπολέμηση της συστημικής διαφθοράς. Ε, η προσφυγή και οι καταγγελίες σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα θα πρέπει να αυξηθούν. 23-24 τα άρθρα αυτά ελέγχονται πλέον. Ελπίζω οι αρχές να δείξουν και να ανοίξουν οικονομικούς και λοιπούς πόρους για το δικαστικό σώμα. Τέλος, σε ό,τι αφορά περιπτώσεις και υποθέσεις ε, διαφθοράς με μεγάλη προβολή, ε, είναι σπάνιες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά είναι σημαντικές. Ε, και θα πρέπει να καταπολεμηθούν. Επίσης το κράτος δικαίου στη Σερβία δεν θα μπορέσει να θεωρηθεί καθιερωμένο όσο δεν ε, ερευνηθεί πλήρως και εξονεχιστικά η δολοφονία του Πρωθυπουργού Ζένσιτς ε, και δεν προσαχθούν τα υπέτη. Επίσης η δολοφονία δημοσιογράφων κατά το κράτος του Μιλόσεβιτς. Η Σερβία λοιπόν πηρεί κάποια πολιτικά κριτήρια. Παρ' όλα αυτά οι ηγέτες της Σερβίας θα πρέπει να οικοδομήσουν ένα καθεστώς εμπιστοσύνης και καλύτερες σχέσεις με τον συνασπισμό και με την αντιπολίτευση. Επίσης τίθεται το θέμα της καθαίρεσης του Δημάρχου του Πελεγραδίου που ήταν αντίπαλου πολιτικού κόμματος. Δεν υπάρχει λοιπόν ουσιαστική αντιπολίτευση δεδομένου του ποσοστού ανεργίας στη χώρα και του επίπεδου δημόσιου χρέους, το οποίο αυξάνεται παρεμπιπτόντως, θα πρέπει να υπάρξει συνένεση για τους στρατηγικούς στόχους ε, της χώρας. Και αυτό καθίσταται όλο ένα και μεγαλύτερη ανάγκη. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση μπορούν να συνεργαστούν. Αυτό φάνηκε όταν εκπρόσωποι της αντιπολίτευση ανέλαβαν την Προεδρία της Επιτροπής ε, για τις Ευρωπαϊκές Σχέσεις και της Σχετικής ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Σταθεροποίηση της Περιφέρειας. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πρόκειται για την τελευταία εξέταση της έκθεσης για τη Σερβία στην τρέχουσα θητεία. Θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω σε όλους πώς έχει πετύχει τα τελευταία πέντε χρόνια η Σερβία. Όταν μαζευτήκαμε εδώ τον Ιούνιο του 2009 Ακόμα και συμφωνία σταθεροποίησης και εταιρικής ε, σχέσης με τη Σερβία υστερούσε λόγω έλλειψης ε, συνεργασίας της τότε κυβέρνησης με το Διεθνές Δικαστήριο. Έχουν εφαρμοστεί έκτοτε οι σχετικοί όροι και έχουν ξεκινήσει επιφέτος ο διάλογος για την προσχώρηση, οι συζητήσεις για την προσχώρηση και είμαι βέβαιος ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα στην επόμενη θητεία. Ήταν δύσκολο να πετύχουμε αυτό το σημείο και πολλές προκλήσεις ε, θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, αλλά είναι βέβαιο ότι η Σερβία οδεύει προς την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Τετάρτη θα συναντηθώ με τους κοιόντες συζητητές για να συζητήσουμε τις ε, συμβαστικές τροπολογίες που επεστάλησαν σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Κατσίν, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματο του κ. Σόπφλιν, που είναι σκιώδη του ΕΛΚ, και να παρουσιάσω τα σχολεία του. the... Καλωσορίζω την έκθεση. Είναι πλήρης και λακωνική, καλύπτει τα σημαντικά στοιχεία της, των σημαντικών εξελίξεων της Σερβίας και πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνεί με τη δήλωση ότι η Σερβία προοδεύει στην πορεία την ενταξιακή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχάσει τον τελικό στόχο. Είναι σαφές επίσης ότι η κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι η ευρωπαϊκή επιλογή είναι καλύτερη επιλογή για τη Σερβία. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι οι διαφορετικές συμφωνίες με το Κοσφοπέδιο είναι υψηλότατης προτεραιότητας και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό. Μία χαλάρωση της έντασης της Σερβίας και του Κωσυφοπεδίου είναι ο τελικός στόχος. Συμφωνούμε επίσης ότι θα υπάρξουν δυσκολίες στην επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά ότι η πολιτική βούληση για να κινηθούν οι δύο χώρες προς αυτή την κατεύθυνση είναι σαφής. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τομείς, πολλές άλλες, Πολλέ περιοχές όπου πρέπει να γίνουν σημαντικέ προσπάθειε από τη σερβική κυβέρνηση. Θα πρέπει να σημειωθούν σημαντικά βήματα στι σχέσει με, τη Σερβία με τους γειτονές της και κάποιες από τις τροπολογίες των πολιτικών μας ομάδων ε, ζητούν το άνοιγμα όλων των αρχείων καθώς και των αρχείων των κομμουνιστικών μυστικών υπηρεσιών. Το θέμα της, του, συγκεντρωτικού, του συγκεντρωτισμού στη Σερβία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο συνολικά η αυτονομία της Βοηβοδίνης έχει διαβρώσει την εξουσία της κεντρικής κυβέρνησης. Ο ανασχεδιασμός των συνόρων των περιφερειών δεν είναι κάτι το επιθυμητό. Η συνταγματική μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης είναι απαραίτητη και η σωστή χορήγηση της δικαιοσύνης είναι πολύ απαραίτητες εφόσον η χώρα θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η μείωση του δημόσιου τομέα που είναι τεράστιο βάρος για την οικονομία είναι μία άλλη πτυχή αυτού του προγράμματος. Ε, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι πολύ περισσότεροι από τους ιδιωτικού υπαλλήλου. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι ουσιαστικές και στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Η επιτυχία σε αυτόν τον αγώνα μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και επομένως να βελτιώσει και το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων της χώρας. Παράλληλα, η δημιουργία καλύτερων ε, συνθήκων ζωής θα έχουν επιπτώσεις στις μεταναστευτικές τάσεις που επηρεάζουν σοβαρά τη χώρα. Ακόμα μία φορά, συγχαρητήρια στον κύριο Κατσίν για την θαυμάσια έκθεση. Ευχαριστώ κύριο Στάνο και ο επόμενος εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Συγχαρητήρια ως πρόεδρος. Είσαστε εξαιρετικός ως προσωρινά προεδρεύων. Η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών είναι υπέρ της υποψηφιότητας της Σερβίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων. Και τα κεφάλαια 23-24 νομίζω θα πρέπει να είναι οι κύριες προτεραιότητες σαφώς σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Και όταν πήγα πρόσφατα στο Μαυροβούνιο, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τη διαφθοράς κτλ. πρέπει να είναι η κυρία προτεραιότητα. Όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά πρέπει και να πιστούν και οι ψηφοφόροι ότι αυτά τα θέματα διευθετούνται και διεκπεραιώνονται διότι και η θέση, η τοποθέτηση και των κρατών μελών είναι σημαντική για τα Δυτικά Βαλκάνια. Πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Η πρώτη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, η καταπολέμηση της διαφθοράς, το οργανωμένο έγκλημα, το ξέπλυμα χρήματος, καθώς επίσης και τα θέματα διακυβέρνησης. Ε, από τουλάχιστον δύο ε, μέλη ε, έχει ασκηθεί πίεση και όχι μόνο για το 3-2-4 ε, το άρθρο όσον αφορά την ε, κρατικοποίηση αλλά επίσης και τα θέματα των ενεργειακά θέματα του δημόσιου τομέα όπου καθυστερούν οι μεταρρυθμίσεις στη Σερβία. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει ιδιαίτερα να αποτίσουμε φόρο τιμής στα πεπραγμένα της Βαρόνης Άστον που αρχικά ήταν εκείνη η οποία ξεκίνησε αυτό τον ε, διάλογο με το Βελιγράδι. Η τροπολογία μου όμως η 26 απορρίπτει μια άμεση διασύνδεση προόδου στις διμερείς σχέσεις ε, όσον αφορά το κοσυφοπέδιο για την ε, αξιολόγηση της προόδου της Σερβίας. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και πρέπει να αφήσουμε τον χρόνο να οριμάσει ώστε τα πράγματα να προχωρήσουν. Και το κοσυφοπέδιο σε σχέση με την αναγνώριση που έχει τύχει, τις αναγνώρισης που έχει τύχει από κράτη-μέλη, σε σχέση με τη Σερβία δεν πρέπει να μεροληπτούμε. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τον κύριο Κάτσιν ε, για την έκθεσή του. Και από πλευράς της εισήγησης για το ε, Μαυροβούνιο ε, καλοχαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός Τζουκάνοβιτς του Μαυροβουνίου ήταν, είχε αναλάβει την πρωτοβουλία αυτή επίσκεψης, επίσκεψης ε, γειτονικής χώρας από την ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου. Αυτό δείχνει ότι μπορούν οι διμερείς σχέσεις ε, να προωθηθούν και να καλλιεργηθούν μεταξύ Σερβίας και Μαυροβουνίου εδώ. Ευχαριστώ. Δίνω τον λόγο στον συνάδελφο ζητώ συγγνώμη που προηγούμενα δεν ε, του έδωσα τον λόγο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ακόμα δυσκολότερος ο ρόλος ε, από ότι ο δικός σας. Ε, διότι εσείς είχατε αναλάβει να εκπροσωπήσει συνάδελφο, εγώ εκπροσωπώ την κυρία Κόπα. Πρέπει να καταδείξετε λοιπόν κατανόηση σχετικά. Πρώτον, ήθελα να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσει η κυρία ε, Κοπά τον ε, εισηγητή, κύριο Κάσιν, για την πολύ καλή έκθεσή του και υποστηρίζεται από πλευρά τη σοσιαλδημοκρατική ομάδα η διαδικασία προσέγγιση στην Ευρώπη τη Σερβία και όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Έχουμε σημαντική πρόοδο που έχει επιτελεστεί από τη Σερβία και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αυτή η ένταξη και ολοκλήρωση θα έχει ιδιαίτερα δυνατό χαρακτήρα. Επίσης σε σχέση με το Συμβούλιο ζητούμε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη διαπραγμάτευση αυτή για την ε, ένταξη της ε, Σερβίας, προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν σημειωθεί πρόοδοι. Μεγάλα βήματα έχουν γίνει σε σχέση με την ε, αρχή της εξομάλυνσης ε, των σχέσεων της Σερβίας και των τοπικών περιφερειακών εκλογών στο Κωσυφοπέδιο και σε σχέση και με την σερβική κοινότητα και τη συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές παρόλα τα γεγονότα βιοπραγιών που σημειώθηκαν στον πρώτο γύρο. Και επίσης ε, θα πρέπει να βοηθηθεί η Σερβία να ξεκινήσει τις διαδικασίες ε, ε, ένταξης. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μονομερής πίεση και όροι και προϋποθέσεις που θα τίθενται, αλλά πρέπει αμφότεροι οι εταίροι και η Σερβία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστούν. Οι διαπραγματεύσεις θα είναι μια μακρά οδός που αναμένει την ε, Σερβία και πρόοδος πρέπει να επιτευχθεί σε πολλά θέματα που εκκρεμούν όπως ε, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την καταπολέμηση της διαφθοράς ε, που ήδη αναφέρθηκαν από προλαλήσαντες όπου σημαντική πολιτική βούληση απαιτείται για να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις οι Σέρβοι. Η ανεξαρτησία των μέσων του τύπου, διαφάνεια σε σχέση με το καθεστώς ιδιοκτησίας ε, μέσων ε, ενημέρωσης, ε, μέσων του τύπου. Πρέπει να αναλάβει δράση κατά ομάδων χουλιγκάνων η Σερβία και πρέπει να προαχθεί η κατανόηση όσον αφορά και τις διαφορετικές σεξουαλικές επιλογές πολιτών. Η αρνητική διακριτική μεταχείριση των γυναικών στην αγορά εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν ε, ε, εκπροσωπούνται επαρκώς οι γυναίκες στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας παρότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις πρόσφατα που είναι θετικές. Επίσης αυτά είναι θέματα που έχει καταθέσει τροπολογίες η σοσιαλδημοκρατική ομάδα και από αυτών επικεντρώνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και πραγματικά κάνατε ό,τι μπορούσατε για να μας διαβιβάσετε αυτές τις απόψεις. Ο κύριος Στυλ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσω και εγώ την έκθεση του κύριου Κατσίν για την Σερβία. Ισορροπημένη έκθεση και η συνολική αποτίμηση είναι ότι η Σερβία έχει φτάσει στο επίπεδο που της επιτρέπει να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό οφείλεται στη βελτίωση κυρίως των σχέσεων που έχει πετύχει η τελευταία κυβέρνηση με το Κοσφοπέδιο. Πέρα από τα σχόλια του κύριου του Τάνοκ, εγώ πιστεύω ότι αυτό το γεγονός ε, στηρίζει την πολιτική κατάσταση σήμερα και γιατί να μην το αναγνωρίσουμε. Τρία σχόλια σημαντικά κατά την άποψή μου. Καταρχάς, η εφαρμογή της ε, συμφωνίας ε, Βελτίωση των σχέσεων. Αυτό θα πρέπει να παρακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια συμφωνία που έχει συνάψει η, Σερβία και η εφαρμογή αυτής της συνθήκης εξομάλυνσης των σχέσεων ε, με αυτή τη χώρα, με το κοσφοπέτη, δηλαδή, καθώς και με άλλες χώρες, είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να παρακολουθεί το κατά πόσο εφαρμόζεται. Ένα δεύτερο θέμα είναι οι αγνοούμενοι. Το είχαμε αναφέρει και σε άλλες εκθέσεις. Παραδείγματο χάρη για τη Σερβία, Ερζεγοβίνη. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε και στην έκθεση για τη Σερβία. Εγώ πρότεινα κάποιε τροπολογίες για τους αγνοούμενους. Κάποιοι συνάδελφοι ζήτησαν το... να ανοίξουν και τα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών. Εγώ θέλω να ανοίξουν και τα αρχεία του πρώην Ιουγκοσλαβικού στρατού του GNA. Γιατί εκεί είναι οι περισσότερες πληροφορίες για να δούμε πού βρίσκονται οι αγνοούμενοι. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να υπάρχει στην έκθεση. Τέλος. Το θέμα των μειονοτήτων έχει τονιστεί, αλλά υπάρχουν διάφορες τροπολογίες που έχω υποβάλει και εγώ, καθώς και άλλοι, για να τονίσουμε πιο έντονα αυτό το θέμα. μία, μία παρατήρηση που αφορά και τη Σερβία αλλά και όλες τι υπόλοιπε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης. Νομίζω ένα νέο στοιχείο το οποίο όπως είπε και η Κομισιόν θα συγκεντρώσει πολύ προσοχή και νομίζω ότι πρέπει να μην το λησμονήσει και η έκθεση. Ευχαριστώ κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι έχω ζήσει την περίοδο της ΕΛΑ από την περίοδο του Σλόμποντα Μιλόσεβιτς και εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στη Σερβία. Έχω κοινά με το σερβικό λαό και την πολιτική και σήμερα το πρωί διάβασα για μία περίπτωση ενός Αυτό διάβασα σήμερα. Αυτό είναι σοβαρό και θέλω να το θέσω. Δεν το άκουσα. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ και στην αδελφή Κατσίν δεν το έχω θέσει ως τροπολογία. Ίσως όμως καλό θα ήταν να γίνει μια συζήτηση γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό, σημαντική η συζήτηση. Εδώ και κάποιες εβδομάδες ακούω και λαμβάνω έγγραφα ότι ε, ξανά όπως την περίοδο Μιλόσεβιτς ε, υπάρχει μια συγκέντρωση εξουσίας σε ένα άτομο το άτομο αυτό φαίνεται ότι έχει ε, άνετη και χαλαρή στάση έναντι στο κοσφοπέδι. Τα αφήνουμε να περνάει αυτό. Μιλάω για τον ε, ε, κύριο Βούσιτς. Μιλάμε για τον... Ε, ο κυτρινός τύπος έχει βοήσει από σκάνδαλα και να σας πω ότι επειδή παρακολουθούσα πολύ τη Σερβία όταν ήμουν δημοσιογράφος, υπάρχει, γίνεται λόγος και μάλλον η δημοκρατία πηγαίνει προς τα πίσω, οπισθοδρομή στην Σερβία. Έχω λοιπόν μία ερώτηση να σας κάνω. Είναι υπερβολικά αυτά, αυτές οι αναφορές ή πρόκειται για τάσεις ε, ανησυχητικές για συγκέντρωση εξουσίας ε, στον αντιπρόεδρο Βούσιτς ο οποίος παρεμβαίνει στα μέσα ενημέρωση, ε, στις μυστικές υπηρεσίες, σε θέματα πολιτισμικά και δεν ακούγεται τίποτε γι' αυτόν. Κοιτάξτε, δεν ξέρω μαθαίνοντα αυτά αν θα πρέπει να ανησυχούμε. Είμαι και υπέρμαχος της προσχώρησης στη Σερβία, αλλά να μην ε, ακολουθήσει τη λανθασμένη οδό η χώρα. Να μην το γνωρίσουμε αυτό επειδή ε, το άτομο αυτό είναι διαλλακτικό σε ό,τι αφορά το κοσυφοπέδιγο. Μην γυρίσουμε λοιπόν την πλάτη σε αυτό το γεγονός. Δεν το άκουσα αυτό και θεωρώ ότι είναι κακό, κακή ένδειξη αυτή για το κοινοβουλίο μας, το γεγονός ότι δεν το έχουμε συζητήσει. Ευχαριστώ. Κύριε Πόσελτ είναι ο Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Μπέλτερ. Είναι σημαντικό παρατηρώντας τις διαδικασίες ε, και τις συνομιλίες μεταξύ της ε, Σερβίας και του Κοσμοπεδίου, να μην ξεχάσουμε, να μην παραμελήσουμε τι γίνεται και μέσα στην ίδια τη Σερβία. Αλλά ο συνάδελφος Κάτσιν θα πρέπει να παραδεχτώ, έχει καταρτήσει μια πάρα πολύ ισορροπημένη έκθεση, στην οποία αναφέρει πολλά σημαντικά στοιχεία. Πρέπει να σας πω ότι επισκέφθηκα προσφάτως την Σερβία και την επισκέπτομαι τακτικά και έχω λοιπόν αποκομίσει την αίσθηση ότι πραγματικά έχει γίνει πρόοδος. Υπάρχουν κάποια θέματα και το θέμα του κοσυφοπεδίου, τα οποία πλέον τα συζητούν με πιο ανοιχτό τρόπο, τα οποία μπορούν να συζητηθούν και με ε, αμφιλεγόμενο τρόπο. Υπάρχουν πολιτικοί δημόσια άτομα τα οποία τοποθετούνται με σαφήνεια και δηλώνουν ότι χάθηκε το κοσυφοπέδιο, άλλοι τους ε, ε, διαφωνούν μαζί τους, αλλά εν πάση περιπτώσει πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση την οποία δεν μπορούσαμε να κάνουμε και να φανταστούμε πριν από κάποια χρόνια. Άρα θεωρώ με πάσα ειλικρίνεια ότι υπάρχουν, υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Αλλά υπάρχουν και οι εξελίξεις τις οποίες έδειξε ο συνάδελφος Μπέλντερ. Και εγώ έχω δύο ομάδες ε, τροπολογιών όπως τις κατέθεσα. Η πρώτη ομάδα έχει να κάνει με κάποια στιγμή τα οποία αναφέρω και στην έκθεση για την, το κοσφοπέδιο για την οποία είμαι εισηγητής φυσικά. Δεν πρέπει να βλέπουμε την κατάσταση στο κοσφοπέδιο και στη Σερβία και να σας πω ε, ότι είμαι υπέρ της κίνησης των συνομιλιών με την Σερβία παρά το γεγονός ότι αυτό δεν είναι δημοφιλής άποψη στην ε, Γερμανία ούτε μεταξύ των συναδέλφων, ούτε μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Εγώ είμαι υπέρμαχος όμως. Αλλά Τονίζω ότι θα πρέπει να επιτύξουμε με την Σερβία επικριτική στάση όπως και με τις υπόλοιπες χώρες της υποψήφιας και η γλώσσα, η διατύπωση στις διαφορετικές εκθέσεις θα πρέπει λίγο πολύ να είναι η ίδια γιατί θέτει ένα, ξέρετε, μέτρο. Να εστιαστούμε και να κοιτάξουμε λοιπόν θέματα διατύπωσης ε, σε ό,τι αφορά θέματα την έκθεση στο Κωσυφοπέδιο για παράδειγμα. Να υπάρχει μια ισόρροπη διατύπωση, να μην ε, τα μπλέκουμε. Και κυρίως ό,τι αφορά το θέμα των μειονοτήτων. Εδώ θα θέλω να πω ότι στην Σερβία δεν είναι μόνο η Ρωμά. Ούτε μόνο η Βοηβοδίνα, όπως αναφέρεται συχνά. Υπάρχει και το Νομιπάσα, υπάρχει και το Πρέσβο. Στην κοιλάδα αυτή υπήρξε ένα ε, έντονο επεισόδιο την τελευταία εβδομάδα. Ε, ένοπλες δυνάμεις στράφηκαν κατά ενός σχολείου και επειδή έχω πάει συχνά στον Πρέσιβο, να σας πω, συνάδελφοι, ότι αν είχατε δει αυτή την ένοπλη επίθεση, δεν είναι αστυνόμοι όπως στην χώρες που γνωρίζουμε, τις πιο πολλές χώρες που γνωρίζουμε. Όχι, μιλάμε για δυνάμεις οι οποίες προκαλούν έντονο σοκ στους ε, άμαχους. Και αυτός είναι και ο σκοπός τους άλλωστε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μια έντονη κρίση και γι' αυτό λοιπόν ε, θέλω ότι ναι, να αναγνωρίσουμε τις ε, προοδούς, αλλά τα κρίσιμα σημεία, τα σημεία της κριτικής να τα τονίσουμε και αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να σας τονίσω ότι είναι, είναι επικοδομητική η στάση που κρατώ και κατά βάση συμφωνώ με αυτά που προτείνει ο συνάδελφος Κάτσιν. Ευχαριστώ κύριε Πόσελ, τον κύριο Σπλέγκοβιτς. Ευχαριστώ. Έντουαρτ, για όλα όσα είπες. Να προσθέσω κι εγώ μερικά πράγματα στην έκθεση Κατσίν. Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στα πλαίσια μιας αντιπροσωπείας στο Βελιγράδι για την ένταξη των χωρών της Νοτιολικής Ευρώπης και είδαμε σε ποιο βαθμό το πρόσφατο άνοιγμα των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σημαντικό για να αυξηθεί η σταθερότητα στη Σερβία και να βελτιωθεί η πολιτική κατάσταση, ειδικά σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της χώρας ε, και σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες των πολιτών. Μετά από όλα τα γεγονότα των οποίων γίναμε μάρτε τα τελευταία 20 χρόνια. Κάτι που ήταν πολύ σημαντικό είναι να συνεχιστεί η εφαρμογή της Συμφωνίας Εξομάλυνσης των Συμφωνιών και στις 3 Νοεμβρίου έγιναν οι πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ε, θα πρέπει να βασιστούμε στην πρόσφατη εμπειρία αξιολογώντας τη Σερβία που αποκομίσαμε από την Κροατία και νομίζω ότι μια νέα μεθοδολογία και ένα νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο θα ήταν καλό ειδικά σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση των κεφαλαίων για τη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, που θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην παγίωση των θεσμών της Κροατίας. Φυσικά η Σερβία θα πρέπει να σεβαστεί τα κριτήρια που έχουμε θέσει και τα ορόσημα που υπάρχουν, που θα είναι πολύ σημαντικά για την σωστή προετοιμασία όλων των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την οικονομία. Η σερβική κυβέρνηση προσπαθεί από ό,τι είδαμε να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα προσλαμβάνοντας ξένους ε, διακεκριμένους ε, συμβούλους και προσωπικότητες για να τις συμβουλεύσουν για τα οικονομικά. Υπάρχουν επίσης διάφορα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση τα οποία και η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει ούτως ή άλλως. Τα εφαρμόζει λοιπόν και η Σερβία στη δική της στρατηγική. Με τις σωστές αλλαγές όμως, με τις κατάλληλες αλλαγές. μουτάν μουτάντης. Και πιστεύω ότι αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν τόσο ώστε να υπάρξει σωστή οικονομική διακυβέρνηση, ο σωστός μηχανισμός και όταν χρειαστεί να εφαρμοστεί και το οικονομικό εξάμεινο και όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την οικονομική διακυβέρνηση. Επίσης, για τους γείτονες με τη Σερβία. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των σχέσεων με τους γείτονες. Είναι πολύ σημαντική διαδικασία συμφιλίωσης. Και ακριβώς γι' αυτό η Σερβία θα πρέπει να λάβει περισσότερα βήματα για να εντοπίσει τους αγνοούμενους, ειδικά εκείνους ε, που στις αρχές δεκαετίας του 90 χάθηκαν ε, στα πλαίσια της σύγκρουσης ε, με την Κροατία. Υπάρχουν πολλές οικογένειες που δεν ξέρουν τι έγιναν οι δικοί τους. Ε, πρόσφατα γιορτάστηκε η 20η επέτειος της πτώσης του Βουκοβάρ. Είναι πάρα πολύ εμβληματική η πετειος της πτωσης του βουκοβαρ ειναι αυτή για τη Σερβία. Ε, οι αγνοούμενοι, τα εγκλήματα πολέμου, θα πρέπει να συνεχίσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αγγελικές αρχές, της Σερβίας και θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια δίωξης των εγκλημάτων. Η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Οι διμερείς συμφωνίες που έχουν ήδη συναθεί θα πρέπει να εφαρμοστούν. Η προστασία των εθνικών μειονοτήτων θα πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε κυβερνητικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με βάση εμπειρίες που έχουμε από άλλες χώρες, θα πρέπει και στη Σερβία να γίνουν προσπάθειες, ούτω ώστε να χρησιμοποιηθούν σωστά τα κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, που είναι πολύ σημαντικά και θα βοηθήσουν τη Σερβία για να αυξήσει τη συμμετοχή του κοινού σε αυτή την πορεία για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βλέπω άλλους ευρωβουλευτές να θέλουν τον λόγο. Η Κομισιόν τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με άλλους ευρωβουλευτές και ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Κατσίν, τον εισηγητή. Πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ ένα πολύ ισορροπημένο σχέδιο ψηφίσματος που ούτως ή άλλως ε, συμπίπτει και με τα πορίσματα της έκθεσης πρόοδου που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2013 ήταν ιστορική χρονιά για τη Σερβία. Όχι μόνο λόγω της συμφωνίας με, πρωτοφανούς συμφωνίας με το Κοσμοπέδιο, αλλά γιατί παράλληλα η κυβέρνηση κατάφερε να δώσει νέα πνοή στις μεταρρυθμίσεις και να προσεγγίσει την περιφερειακή συνεργασία και τη σχέση με τις γειτονικές χώρες με πιο δυναμικό τρόπο. Λόγω αυτών των θετικών πολιτικών εξελίξεων σε αυτούς τους τρεις τομείς η Κομισιόν μπόρεσε να συστήσει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να το δεχτεί ούτως ή άλλως τον Ιούνιο που μας πέρασε. Έκτοτε έχουμε ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις και όπως είπε ο κύριος Κατσίν ξεκινήσαμε ήδη με την με τα κεφάλαια 23 και 24 και 32 οικονομικός έλεγχος και θα συνεχίσουμε με τις διμερείς επαφές τον Δεκέμβριο. Και εκεί θα αντιμετωπίσουμε πολλά από τα θέματα τα οποία αναφέρατε εσείς σήμερα. Καλωσορίζουμε αυτό το ψήφισμα, είναι πολύ ισορροπημένο Λέει ότι υπάρχουν και πολλές προκλήσεις στον δρόμο της Σερβίας, αλλά και τη συγχαίρει για τα θετικά που έχει κάνει. Συνοπτικά να σας πω που θεωρούμε ότι υπάρχουν οι βασικές προκλήσεις. Το κράτος δικαίου, η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς φυσικά, η ανεξάρτηση των βασικών θεσμών, η ελθοτυπία, καταπολέμηση των διακρίσεων, προστασία των μειονοτήτων και ε, ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό θα είναι, το, θα είναι όλα αυτά στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, θα είναι μακρά διαδικασία. Θα παρακολουθούμε τις μεταρρυθμίσεις της α, Σερβίας εκ του Σύνεγγης, τώρα που ξεκινήσαμε τις προτεξιακές διαπραγματεύσεις. Υπάρχει και μια άλλη πρόκληση για την κυβέρνηση της Σερβίας, κατά την άποψή μας. Το να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες, κατά την άποψή μας, και να τους μιλήσουν για τα ωφέλη από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καθ' όλη τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων θα πρέπει να υπάρχει αυτή η επαφή. Γι' αυτό η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ε, που συνεδρίασε τον Νοέμβριο ήταν, είναι πολύ καλός ε, τρόπος για να, έρθουν σε επαφή, να έρθουμε σε επαφή με το Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών της Σερβίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στην πρωταξιακή διαδικασία. Συνολικά υποστηρίζουμε αυτό το ψήφισμα. Και για να απαντήσω το ερώτημά σας, αν λαμβανόταν ποτέ μια απόφαση για μια διακυβερνητική διάσκεψη πριν από τον Ιανουάριο η Κομισιόν θα ήταν έτοιμη για να παίξει το δικό της ρόλο, ούτως ώστε να παραστεί σε αυτή τη διάσκεψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα να συνοψίσει ο εισηγητής αυτή τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. De facto, πραγματικά, πρόεδρε, από πλευρά της Επιτροπής Εξωτερικών και όσον αφορά την σκιώδη εισήγητη από πλευράς ε, ΕΛΚΑ έχουν τα πράγματα σημαντικά βελτιωθεί και αυτό είναι πολύ θετικό. Μέσα σε ένα τέτοιο πνεύμα θα προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε μια ισορροπημένη έκθεση όσον αφορά τη Σερβία και νομίζω ότι τα καταφέραμε όπως τονίσατε όλοι σας στις παρεμβάσεις σας. Όμως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και αναφέρατε κάποιες λεπτομέρειες εξάλλου. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα όλες αυτές τις μικρολεπτομέρειες από πλευράς μας. Ο κύριος Τένοκ ανέφερε την διαφθορά ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Συμφωνώ μαζί του. Ανέφερε ιδιαίτερα και τη μεταβατική περίοδο ή την μετάβαση όσον αφορά τα θέματα του άρθρου 359 που δεν υφίσταται πλέον και που μετατέθηκαν στο 3 2, 3, 4 ως άρθρο τα σχετικά θέματα. Το πρόβλημα είναι η κατάχρηση άρθρων από πλευράς ε, της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυτά ως πρόσχημα. Είναι κάτι που θα πρέπει <clears throat> οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να κατονομάσουμε τα θέματα όσον αφορά τους μαφιόζους ε, που ε, έχουν τους επιχειρηματίες ως ομήρους και δυσκολεύουν τα πράγματα πολύ περισσότερο σε σχέση με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η καταπολέμηση αυτού του είδους της διαφθοράς για να επιτευχθεί χρειάζονται σημαντικές προσωπικότητες και ο κύριος Μπέντερ εξέφρασε κάποια παράπονα σε σχέση με το σθένος κάποιων προσωπικότητων. Χωρίς ε, στεναρή βούληση, χωρίς εξουσία και στεναρή στάση δεν είναι είναι δυνατόν να γίνει τίποτα. Δεν θέλω όλα να τα ευλογήσω όσα συμβαίνουν σε σχέση με τη Σερβία. Θέλω μόνο να πω πόσο σημαντικό είναι το ότι στρέφονται σε αυτό το τεράστιο έργο που έχει βαθιές ρίζες στο θέμα της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος στη Σερβία. Και από την άλλη πλευρά οι σχέσεις καλής γειτονίας έχει, ε, έχουν, οι σχέσεις καλής γειτονίας έχουν τεράστια σχέση. Και θέλω να αναφέρω και τον θετικό ρόλο που διαδραματίζει η Σερβία στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Είναι πολύ πιο καρποφόρα τα πράγματα και γόνιμα από ό,τι στο παρελθόν. Όταν κάποιοι από τους πολιτικούς ηγέτες προσπαθούσαν να αυτοπαρουσιαστούν ως <clears throat> έχοντας ε, στενούς δεσμούς με την ε, προηγούμενη Προεδρία και την προηγούμενη κυβέρνηση και αυτό ήταν ένα πρόσχημα να τηρούν μια απόλυτα αντίθετη θέση και τοποθέτηση από αυτά τα οποία απαιτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα, σε σχέση με την ιδιαίτερη προσοχή για τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν ως προς αυτά τα θέματα, σημαντικό όμως είναι να υπογραμμίσουμε και κάτι, ότι ο, διάλο, διάλογος σε σχέση με τους αγνοούμενους είναι μια αναγκαία προϋπόθεση μεταξύ των αρχών της ε, Σερβίας και της Πρίστινα στο Κωσυφοπέδιο. Αυτό δείχνει ότι αντιμετωπίζουν ε, τις πιο βαθιά ριζωμένες, ε, ας το πω έτσι, προβληματικές καταστάσεις και πρέπει αυτό να θεωρηθεί θετικό, όχι μόνο μόνο για αυτούς αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Ο κύριος Μπέντερ έκανε κάποιες ε, αναφορές και είπε <clears throat> ότι υπάρχει κάποιο υπόλοιμα <clears throat> των ε, δράσεων και των, ε, της κληρονομιάς του Μιλόσεβιτς που ίσως κάποια, από κάποια στοιχεία αυτού του κληροδοτήματος συνεχίζονται όπως παλιότερα υπό τον Μιλόσεβιτς. Θα έλεγα ότι αυτό όμως πολιτικά δεν είναι δίκαιο να το πει κανείς θεωρώ ότι όλες ε, οι πολιτικές, όλα τα πολιτικά κόμματα μεταμορφώθηκαν, ε, άλλαξαν, μεταβλήθηκαν και μάλιστα εκβάθρων. Και σε σχέση με το ηγέτη του, ε, του Σοσιαλιστικού Κόμματος θα συναντηθούμε για πολλωστή φορά, στις Βρυξέλλες και το Δεκέμβριο θα έχουμε και μια συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό. 20 συναντήσεις μέσα ένα χρόνο είναι ένα επίτευγμα που πραγματικά πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το εκτιμήσουμε πολύ θετικά έχουν μεταβεί στη Νέα Υόρκη και έχουν επιστρέψει και χρησιμοποίησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να προαγάγουν ε, τις επαφές ε, και να ε, μπορέσουν να επανορθώσουν τα ασφάλματα όσον αφορά το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει πραγματικά να τύχουν προσοχή και σε σχέση και με την κυρία Άστον πρέπει να αναφέρονται. Διότι χωρίς την ενεργό συμμετοχή της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου δεν θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και όλα αυτά τα πράγματα. Μπορούμε τώρα να κάνουμε υποθέσεις. Έχουν έναν πρωθυπουργό ή έχουν κάποιους σκιώδεις πρωθυπουργούς, αναπληρωτές πρωθυπουργούς. Ναι, φυσικά υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό και όλο και ενδυναμώνεται περαιτέρω. Και παρότι υπήρχε, ένα υπήρξε ανασχηματισμός της κυβέρνησης πριν από κάποιους μήνες, όλο και περισσότερο καθίσταται πρόδειλο ότι σε σχέση με τις ε, ε, κοινοβουλευτικές εκλογές ε, που θα διεξαχθούν σχετικά σύντομα θα έχουμε αυτή την εξέλιξη. Δεν θέλω να τοποθετηθώ σχετικά, αλλά θα υπάρξουν σαφώς πρώιμες, πρόορες εκλογές στη Σερβία και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ενδεχόμενο, αυτό το γεγονός. Να προετοιμαστούμε, να το αντιμετωπίσουμε. Ο κύριος Πόσελτ έκανε λόγο για μειονότητες. Ειδικότερα ανέφερε την κατάσταση στο νότο της Σερβίας. Ναι, φυσικά η Σερβία έχει χωροφύλακες εκεί και έχουν ε, πάρα πολύ μεγάλη εξουσία και μπορεί πολύ σημαντικά να σηματοδοτούνται κάποια πράγματα από αυτές τις δράσεις. Όμως, ο διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και Πριστίνα πιστεύω ότι θα δημιουργήσει θετικά παρεπόμενα και για το, τους Σέρβους τους ίδιους ε, και για τους ε, Αλβανούς ε, ε, όσον αφορά τις δύο αυτές περιοχές. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν ενώπιον των εξελίξεων, μελλοντικών εξελίξεων και πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς αυτές τις εξελίξεις το 2014. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι φυσικά υπάρχουν πάντα φόβοι για τα όσα συμβαίνουν στη Σερβία και τις κατευθύνσεις ε, που ακολουθούν. Αν είναι μια γραμμική προς τα εμπρός ε, προοδευτική, ας το πω σε εξέλιξη, αν είναι θετικά όλα ή όχι. Το πιο όμως σημαντικό είναι να διοργανωθεί αυτή η διακυβερνητική διάσκεψη το δυνατόν ταχύτερα και να ανοίξουν και τα κεφάλαια 23 και 24. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων θα είναι σε, θέμα, σε θέση με να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα πολύ ευαίσθητα θέματα και θα έχει εργαλεία και μέσα στα χέρια της για να επηρεάσει τα πράγματα ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο θετικό πλαίσιο και εμείς θα μπορέσουμε από την άλλη πλευρά να ε, τοποθετηθούμε με ιδιαίτερα, θα, ας το πω ε, αυστηρό πνεύμα για αυτές τις ε, εξελίξεις ως ε, αδέκαστοι κριτές. Πιστεύω ότι σε σχέση με την ε, συμφωνία για τη συμβαστική τροπολογία θα ψηφίσουμε στις 5 Δεκεμβρίου αυτή τη συμβαστική τροπολογία. Θα είναι πολύ σωστή η στιγμή να αποσταλεί ένα μήνυμα προς το Συμβούλιο, να υπομειστεί το Συμβούλιο τις δικές του ευθύνες ε, για να αποφασίσουν προς τα που θα κινηθούν σε σχέση με τη διακυβερνητική διάσκεψη είναι σημαντικό να δράσουν νωρίτερα και όχι να καθυστερήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτό ολοκληρώνει τη συζήτησή μας για το σημείο στην ημερήσια διάταξη υπαριθμών 6. Και χωρίς καθυστέρηση ξεκινάμε με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η έκθεση πρόοδου για το 2013 για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο Ρίτσαρτ Χάουιτ είναι ο εισηγητής μας. Του δίνω μέσα τον λόγο. Παρακαλώ κύριε Χάουιτ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ασυνήθιστο να, έχουμε να έχουμε άπλετο χρόνο μπροστά μας. Είναι περίεργο αυτό το προνόμιο και πολύ ευχάριστο για μια φορά στην ΑΦΕΤ, ε, γιατί έχουμε χρόνο για τα θέματα που μας απασχολούν. Είναι η τρίτη φορά που έχω την τιμή να παρουσιάσω ως εισηγητής ε, το σχέδιο έκθεσής μου για τη χώρα αυτή και το κάνω με μεγάλη χαρά. Την ξέρω τη χώρα, τους ανθρώπους, τους θεσμούς της, πολύ καλά. Είναι με πολύ σημαντική χώρα. Καλό είναι να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Ε, πιστεύω ότι θα συνεχίσει την προσπάθειά της ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η έκθεσή μου απεικονίζει όλα αυτά τα στοιχεία. Παρά τα προβλήματα, παρά τις προκλήσεις, παρά τις επικρίσεις που θα ακούσω στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο γενικά, το σημείο 1 στην πρώτη πρόταση λέει ότι ανεπιφύλακτα θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τεθεί μια ημερομηνία για την έναρξη των ε, ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη χώρα αυτή. Και ελπίζω ότι και φέτος όπως και πέρυσι θα παραμείνει ως έχει αυτή η φράση, χωρίς τροπολογίες, γιατί είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεύτερον, προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και μπορεί εδώ μπορεί να, πολλά από αυτά που λέει η έκθεση μπορούν να τροποποιηθούν πριν φτάσουν στην Ολομέλεια. Αλλά θέλω να σταλεί ένα έντονο μήνυμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο, γι' αυτό δημοσιεύουμε τώρα την έκθεση, ότι ο κίνδυνος ε, υπαναχώρησης είναι απτός λόγω των ε, γεγονότων της 24ης Δεκεμβρίου του, της περσίνης χρονιάς, που ήταν δύσκολη χρονιά, ε, και συμφωνώ ότι ήταν μια χαμένη χρονιά. Αλλά αν θυμάστε, στα συμπέρασμα του, του Συμβουλίου του 2012, το Συμβούλιο λέει στην παράγραφο 2 ότι συμφωνεί με την άποψη της Κομισιόν ότι η απόφαση για έναρξη των διαπραγματεύσεων στην επόμενη Προεδρία ε, σημαίνει ότι η Κομισιόν πρέπει να ετοιμάσει όλο το προπαρασκευαστικό ε, έργο για να γίνει ε, πραγματικότητα αυτό. Αυτό το είπε το περασμένο Δεκέμβριο και δεν θα ήθελα να υπαναχωρήσουμε σε σχέση με αυτά τα συμπεράσματα φέτος. Εν συνεχεία, ε, συμφωνώ με τον Επίτροπο Φίλε όταν παρουσίασε την έκθεση πρόοδου φέτος που είπε ότι οι ανησυχίες που υπάρχουν στο Συμβούλιο και αλλού για τη χώρα δεν τους επιτρέπουν να ορίσουν ακόμα μία ε, ημερομηνία. Ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα κεφάλαια 23 και 24 για τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφού τα ελέγξουμε πρώτα. Ε, καταλαβαίνω ότι εκεί είναι οι περισσότερες ανησυχίες για όσους έχουν επικρίσεις για τη χώρα. Εγώ υποστηρίζω αυτό που είπε η Κομισιόν. Πάμε στο όνομα του ονόματος τώρα. Ακόμα μια φορά. Θέλω να πω επίσημα ότι θα υποβάλω μια οριζόντια τροπολογία σε όλο το κείμενο που θα αφήσει μία ονομασία και μια αναφορά στο, στο επίθετο Μακεδονία. Και όλες τις άλλες ονομασίες θα τις αντικαταστήσει με το όνομα που ε, και όλες τις άλλες αναφορές που λένε η χώρα, αυτή η χώρα κτλ. Γιατί? Γιατί δεν θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει μέσο θέατρο πολέμου, α πούμε, για το όνομα. Και τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω ότι το πετύχαμε. Θα το ξανακάνω αυτό, ε, προτείνοντας ένα όνομα λοιπόν. Τώρα για το όνομα αυτό καθεαυτό, φυσικά η έκθεσή μου ε, θέλει, λέει ότι πρέπει να σημειωθεί η πρόοδο, αλλά κάτι παραπάνω λέει επίση, ε, συμφωνώ με την Κομισιόν, ότι αν δεν υπάρξει πρόοδο για την ένταξη τη χώρα, θα επηρεαστεί η αξιοπιστία της ε, ενταξιακής διαδικασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης στο σχέδιο κειμένου λέω ότι η αποτυχία εδώ και 20 χρόνια του πλαισίου του ΟΗΕ να σημειωθεί ε, πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για το όνομα ε, ρίχνει σκιά και αμφιβολίες για την αξιοπιστία αυτής της διαδικασίας. Ελπίζω να ακούσετε αυτά τα λόγια. Δύο άλλα ε, θέματα για το όνομα που βάζω φέτος. Πρώτον, έχουμε τους Έλληνες που τώρα θα αναλάβουν όσον Σονούπο την προεδρία τους επόμενους 6 μήνες από τις αρχές του 2014. Είχα κάποιες ιδιωτικές συζητήσεις με αυτούς και νομίζω ότι και η Κομισιόν το έκανε, το ξέρω. Δεν θέλω να εκφράσω ψευδείς ελπίδες, είναι περίπλοκο το θέμα, αλλά προσωπικά θα ήθελα δημόσια να πω ότι επίσημα πιστεύω, ελπίζω ότι η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η δέσμευση που έχει η Ελλάδα προς όλη την περιφέρεια θα βοηθήσει ούτω ώστε να σημειωθεί πραγματικά πρόοδος. Δεύτερον, θα έχετε συναντήσει πολλοί από του, τον κύριο Αμέτη που είναι ε, μέλος της ε, κυβέρνησης εθνασπισμού και που ανήκει στην, ε, και εκπροσωπεί την αλβανική μειονότητα. Κάνει διάφορες διεθνείς επισκέψεις ούτως ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα του ονόματος και αποφάσισα στο σχέδιο της έκθεσης να αναφέρω ότι για την αλβανική κοινότητα, αν δεν επιληθεί το όνομα και αν δεν εξασφαλιστεί η ευρωατλαντική ατζέντα, κάτι που θέλουν περισσότεροι στη χώρα, όταν βλέπω την... Όταν βλέπουν την Αλβανία στην έκθεση πρόοδου που έχει προχωρήσει και αν συγκρίνουν ε, αυτή την πρόοδο με την αποτυχία για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ε, θα υπάρχει θέμα. Ε, και το λέω αυτό έτσι με μεγάλη προσοχή και ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Δεν ήθελα να σχολιάσω απλώς την έκθεση πρόοδου, αλλά να πω και κάτι παραπάνω, κάποια καινούργια στοιχεία, ούτως ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα. Υπάρχουν δύο καινοτομίε φέτος που ήθελα να τονίσω για πρώτη φορά. Πέρυσι μίλησα στο ψήφισμά μου για το κόστος της μη διεύρυνσης για τη χώρα. Φέτος θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω και να μιλήσω για την κυβέρνηση της χώρας και να απαιτήσω από την Κομισιόν να μας δώσουν μια ποσοτική ανάλυση για το κοινωνικό και οικονομικό κόστος που θα προκύψει από τη συνέχιση της αποτυχίας ε, ε, για την ένταξη της χώρας, για τη χώρα λοιπόν, για την περιοχή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω να ανταποκριθεί θετικά η Κομισιόν σε αυτή την πρόταση Και ελπίζω και ο Υπουργό Εξωτερικών όταν έρθει στι Βρυξέλλε μέσα στη βδομάδα να αντιδράσει θετικά. Επίση, έχω κάνει και μια σύσταση ότι η χώρα θα πρέπει να αναγνωριστεί με, από την Κομισιόν ως μια χώρα με λειτουργική οικονομία. Φυσικά, όπως άλλες χώρες στην περιοχή έχει υψηλή ανεργία και έχει πολλά άλλα προβλήματα, αλλά η πρόοδος που έχει σημειώσει σε ό,τι αφορά την οικονομία της αγοράς είναι αναφυσβήτητη. Και είναι δικαιολογημένο να πούμε προς την Κομισιόν ότι θα πρέπει ε, να τον αναγνωρίσουν και να, δώσουν, ε, να, να αναγνωρίσουν φέτος. Τώρα, για τα γεγονότα της 24ης Δεκεμβρίου του 2012 έχουν συζητηθεί πολλές φορές στην ΑΦΕΤ, πολλές και άλλες φορές βέβαια. Αλλά για να σας πω, πιστεύω ότι βρισκόμαστε τώρα. Μέσα αυτή τη χρονιά ετοιμάστηκα να εκφράσω έτσι πολύ έντονες, με πολύ έντονα χρώματα να σχολιάσω το τι έγινε και δημόσια. Άκουσα τα διάφορα, τους διάφορους συμμετέχοντες, ε, φορείς, ε, κόμματα κτλ. Και το σκέφτηκα πολύ προσεκτικά και το ζήγησα, το ζήγησα αυτό. Και είπα επίσημα ότι αυτό που συνέβη εκείνη τη μέρα αμφισβητεί τη δημοκρατική νομιμότητα της χώρας. Το είπα έτσι. Ξέρω πολύ καλά ότι είναι πολύ βαριά αυτή η δήλωση. Και το λέω, γιατί κατά την άποψή μου ισχύει, αλλά και γιατί ότι πρέπει να είμαστε πιο μαλακοί με τη χώρα. Την 1η Μαρτίου όμως, ο κύριος Μπούτσακ και εγώ ζητήσαμε να γίνουν διαμεσολαβητές μεταξύ των δύο μερών. Τότε η αντιπολίτευση μάλιστα είχε μποϊκοτάρει την διαδικασία, αλλά τελικά αυτή η προσπάθεια ε, πέτυχε. Και φέτος στο ψήφισμά μου εκφράζω την ικανοποίηση. Ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο, αλλά κυρίως ε, τα ενδιαφερόμενα μέρη τα συγχαίρω. Ε, δημιουργήθηκε και μια εξεταστική επιτροπή και παρά τις μεγάλες προκλήσεις μπόρεσαν να φτάσουν σε συνενετική συμφωνία μετά από λίγους μήνες. Ο κ. Βανούτ είναι ο εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τα μέρη σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι κάνει μια θαυμάσια δουλειά και νομίζω ότι θα μπορέσει να συνεχίσει. Υπάρχει τώρα μια δέσμευση από τα μέρη στη χώρα να υπογράψουν μια συμφωνία για να θέσουν την διατλαντική σχέση και την ευρωπαϊκή σχέση ψηλά στην ατζέντα. Θέλω αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί και αυτό το μνημόνιο επίσης σύνδεσης να εφαρμοστεί. Αυτό λένε ορισμένοι ότι δεν χρειάζεται τελικά να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν τα πάντα της συμφωνίας. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια πρώτη προθεσμία, η οποία όμως δεν γίνεται να εφαρμόσει κάθε στοιχείο της σύστασης μέχρι τη συνοκορυφή του Δεκεμβρίου. Και θέλω μέχρι το Δεκέμβριο ε, να, εφαρμοστεί, να εφαρμοστούν όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Και τελικά θέλω να εφαρμοστεί πλήρω βέβαια στη συμφωνία. Μίλησα αρκετά. Τώρα θέλω να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία της έκθεσης, ορισμένα ε, συμπίπτουν με αυτά που είχα γράψει στο παρελθόν. Θέλω όμως να μιλήσω για τις τρεις συναντήσεις που έγιναν μεταξύ του Βούλγαρου Πρωθυπουργού και του Πρωθυπουργού της Σκοπίων τους τελευταίους εννέα μήνες ε, σε καλό πνεύμα συνεργασία και ελπίζω οι Βούλγαροι εδώ θα συμφωνήσουν ε, ότι έχουμε σε μια έτσι φρασιολογία που θα αναγνωρίζει αυτό το γεγονός. Επίσης, επιμένω ότι όλες οι συστάσεις των συστάσεων των αποστολών παρακολούθησης των εκλογών της ε, ΟΑΣΕ ο ΙΝΤΙΡ να εφαρμοστούν. Η αποκέντρωση πηγαίνει προς την λάθος κατεύθυνση, όχι προς τη σωστή, μας ανησυχεί αυτό. Επίσης υπάρχει ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος στην, στο θέμα της εκπαίδευσης, να συμμετέχουν στον ατόν περισσότεροι. Ξέρω ότι κάποια θέματα εδώ ανησυχούν τους ευρωβουλευτές για την ε, ελευθεροτυπία και την ε, ελευθερία έκφρασης. Εκεί δεν κρατιέμαι, τα λέω ανοιχτά τα πράγματα. Υπάρχουν ξεκάθαρα πράγματα. Ε, επίσης για το φόβο που υπάρχει στη χώρα για επιλεκτική δικαιοσύνη. Και επίσης υπάρχει ανάγκη για να σημειωθεί περισσότερο πρόοδος στα θέματα της δίωξης των ε, υποθέσεων διαφθοράς, αλλά δίωξης όλων των ε, ενόχων. Επίσης για τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων και του κέντρου που υπάρχει για τους ομοφιλόφιλους ε, στα Σκόπια. Υπάρχει συγκεκριμένη παράγραφος για την καταδίκη της βίας εναντίον των ομοφιλοφίλων ανδρών και γυναικών και φιλομεταβατικών στη χώρα θα γίνει και μια στρογγυλή τράπεζα με εκπροσώπους της, ε, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιών. Υπάρχουν δύο ε, γερμανικές οργανώσεις που θα με βοηθήσουν. Εντελώς ανεξάρτητα από την Κομισιόν. Και διάφορες συστάσεις ε, που είχα αναφέρει πέρυσι έχουν εφαρμοστεί. Ιδίως ό,τι αφορά το δεύτερο πρόγραμμα δαπανών του IPA και θα ήθελα να υπάρξει ένα ελάχιστο ποσοστό το οποίο ε, να δαπανάτε όχι μέσω του κυβερνητικού προϋπολογισμού αλλά να δίδεται σε αποκεντρωμένους φορείς και επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια πιο ανεξάρτητη και πλουραλιστική κοινωνία τελευταίο, παρότι υπάρχει και χωριστή έκθεση ε, για αυτό το θέμα, υπάρχει το θέμα της απελευθέρωσης από την υποχρέωση θεωρήσεων. Το συζήτησα με τον εισηγητή της έκθεσης, αλλά έχω γράψει δύο λόγια ότι η Επιτροπή μας θέλει να παραμείνει το σημερινό καθεστώς απελευθέρωσης από την υποχρέωση θεωρήσεων για τη χώρα αυτή. Ελπίζω να θεωρείτε ότι η έκθεσή μου είναι και πλήρης και δίκαιη. Έχω ε, λάβει υπόψη διάφορες τροπολογίες και ελπίζω να ακούσω και άλλες. Ευχαριστώ. Κύριος Κούκαν, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Τώρα μιλώ εξ ονόματος του Σκιώδη του ΕΛΚ για την Μακεδονία λέει ο Θα ήθελα να πω πόσο εκτιμώ καταρχάς την δουλειά του κυρία Χόουιτ και την δέσμευσή του για το θέμα αυτό της ευρωπαϊκής ε, ένταξης της Μακεδονίας. Έχουμε ε, μπροστά μας ένα καλό σχέδιο έκθεσης με κάποια πολύ σημαντικά και ουσιώδη μηνύματα. Συμφωνώ με τη γενική κατεύθυνση της έκθεσης και επίσης υποστηρίζω την έκκληση προς το Συμβούλιο να οριστεί η ημερομηνία για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Μακεδονία χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Επίσης, ε, συμφωνώ σε ό,τι αφορά την αγανάκτηση που υπάρχει σε ό,τι αφορά την επανάληψη τα τελευταία τέσσερα χρόνια του ίδιου μηνύματος. Αυτή η έκθεση σίγουρα θα δώσει έναυσμα για συζήτηση πέρα από την Επιτροπή μας και πιστεύω ότι χρειάζεται τέτοια συζήτηση για να κινηθούν προς τα εμπρό τα πράγματα. Η σύσταση υπερσυνή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλάμβανε την ιδέα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την ένταξη και αυτό θα έπρεπε λοιπόν να συμβάλλει στη δημιουργία των όρων και των συνθήκων στην εξέβρεση λύσης για το όνομα και να βελτιωθούν οι καλές σχέσεις γειτονίας. Αυτή η ιδέα προτάθηκε και φέτος και νομίζω ότι η εξέταση της ε, περιορισμένης προόδου εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τεθεί υποδοκιμή. Θεωρώ ότι θα προωθήσει την επίλυση του θέματος στο Κοινοβούλιο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι με την ένταξη και την προσχώρηση της Μακεδονίας αλλά έχουμε και τα όρια της αξιοπιστίας για την ευρωπαϊκή διαδικασία ενοποίηση στην περιφέρεια. Και υπό την έννοια αυτή είναι ακριβές να υποδείξουμε τους κινδύνους και το κόστος ενδεχόμενης δρόμηση της χώρας. Κάποια μηνύματα εμφανίστηκαν στις αρχές του έτους όταν και βιώσαμε πολιτική κρίση. Αυτό ξεπεράστηκε μεταξύ άλλων και λόγω της αποστολής ε, Φιούλε με τον συνάδελφο ε, Μπούζεκ ε, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδεικνύει αυτό πόσο ευάλωτη είναι η πώς θα μπορούσε να γίνει η πολιτική κατάσταση στη χώρα. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη και να συνεχίσουμε επικοδομητικά την ανάπτυξη της χώρας. Συμφωνώ να τονιστεί η σημασία της εφαρμογής των συστάσεων του Κοινοβουλίου και της ε, σχετικής ε, ερευνητική επιτροπής του Κοινοβουλίου και τη σημασία της διατήρησης πολιτικού διαλόγου μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβερνητικού κόμματος. Αυτό είναι σημαντικό θέμα σε ό,τι αφορά και την ευρωπαϊκή ατζέντα που θα πρέπει να παραμείνει στρατηγική προτεραιότητα της χώρας. Συμφωνώ επίσης με τον επικρατικό τόνο της έκθεσης σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα στην ελευθεροτυπία και την ελευθερία έκφρασης περαιτέρω στο κράτος δικαίου και τα θέματα που άπτονται του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς θα πρέπει να συνεχιστούν να αντιμετωπίζονται. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί πιο πολύ προσοχή σε θέματα εφαρμογής και ε, εφαρμογής και εκτέλεσης του πολιτικού, των πολιτικών συμφωνιών σε ό,τι αφορά και τον πολιτικό και προταξιακό διάλογο. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Χόουιτ και ανυπομονώ και προσμένω την μετέπειτα συνεργασία μας, την πολιτική μας συνεργασία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι, λέει ο κύριο Στάμακ. Δεν είχα ζητήσει το λόγο, αλλά πολύ ευχαρίστω παίρνω το λόγο να συγχαρώ τον σοσιαλιστή συνάδελφο και τον εισηγητή Ρίτσαρτ Χάουιτ από το ECR κανονικά ξέρετε είμαστε από πολύ διαφορετικές ε, άκρες του πολιτικού φάσματος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ταυτίζεται η άποψή μας σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της διαδικασίας ε, ένταξης της Μακεδονίας. Είμαι ένας από τους μεγαλύτερους φίλους της Μακεδόνας και συναντώ και κάποιους πολιτικούς εδώ στι αυτή την εβδομάδα. Έχω μεταβεί πολλές φορές στη χώρα, καταλαβαίνω την αγανάκτηση της κυβέρνησης ε, σε ό,τι αφορά τη διαρκή, το πληρακή μπλοκάρισμα, σε ό,τι αφορά το, την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Δέκα χρόνια πώς έχουν περάσει. Δεν μπορώ να τα μετρήσω πλέον ε. και συνέχεια βάζει βέτο η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, βάσει και μόνο του θέμα του ονόματος, το οποίο είναι ακατανόητο για οποιονδήποτε μη Έλληνα. Είμαι Ελληνόφιλος, ε, ε, σε γενικέ γραμμέ σε όλα τα υπόλοιπα θέματα. Αλλά παρά όλα αυτά, να πω ότι την έκθεση, είναι ισορροπημένη. Σας συγχαίρω για την προσπάθεια που κάνετε. Ο κύριος Πόσολτ έθεσε προηγουμένως μια ερώτηση και έκανε ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά το να συμμετάσχει η Μακεδονία στη συζήτηση για την Αλβανία. Υπήρχε ένα σημαντικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά σχόλια του πρώην Πρόεδρου Μπαρίσα, το οποίο προκάλεσε μεγάλη αποσταθεροποίηση στην περιφέρεια, στην περιοχή, αλλά ευτυχώς αυτό έχει υποχωρήσει πλέον και δεν ακούμε, δεν παρουσιάζονται περαιτέρω προβλήματα. Επίσης, υποδείχθηκε ότι τα δύο βασικά, οι δύο βασικές ομάδες ε, πολιτικές στο Κοινοβούλιο της Μακεδονίας έχουν πλέον συνάψει ειρήνη και ακολουθούν μια πολιτική ε, εθνικής συνένεσης για τις φιλοδοξίες της Μακεδονίας. Ε, ασφαλώς το θέμα δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ. Προφανώς είναι γραφτισμένη η Μακεδονία ε, σε ό,τι αφορά την πρόοδο για το θέμα αυτό και πάλι λόγω της Αθήνας, λόγω του ονόματος, ελπίζω να ασκηθεί μαζική πίεση και στην Αθήνα και στη Μακεδονία για να βρουν μια λύση αμοιβαία αποδεκτή για το θέμα το όνομα, προκειμένου να ευωδώσουν και αυτές οι προσπάθειες. Ελπίζω λοιπόν κάποιος να βρει ένα όνομα που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, όλες τις πλευρές και να μπορέσει να περάσει και από ένα δημοψήφισμα στην ίδια τη Μακεδονία. Πέραν τούτων, να εγκομιάσω τις προσπάθειες της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Σας ελπίσουμε λοιπόν του χρόνου να μπορέσουμε να πούμε κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά τις προπτικές της Μακεδονίας και σε ό,τι αφορά και την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόκ, σε ό,τι αφορά την ελληνική συμμετοχή. Ο κύριος Στήρ ja Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα ήθελα να καλωσορίσω. Είναι καλοδεχούμενη αυτή η έκθεση. Είναι ισορροπημένη και έχει με θετικό τρόπο συνταχθεί. Πρώτα απ' όλα θέλω να καλωσορίσω, να χαιρετήσω το σημείο, το εδάφιο 1, όπου ζητείται από το Συμβούλιο να καθοριστεί μια ημερομηνία για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αλλά και άλλα εδάφια στην έκθεση αυτή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για την ανάγκη να ενισχυθεί το κράτος δικαίου και φυσικά να ανοίξει το κεφάλαιο το θέμα της ελευθερίας των μέσων του τύπου, της ενημέρωσης. Θα πρέπει κάτι να προσθέσουμε για την ανάγκη να υπάρξουν αλλοδαπές επενδύσεις και για την ενίσχυση της διαφάνειας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δημόσιες αγορές και δημόσιες προμήθειες. Θα συμφωνούσα με τον εισηγητή και θέλω να το τονίσω. Στην παράγραφο 24 υπάρχει ανάγκη να σχολιάσουμε κάποια πράγματα. Τον τρόπο για παράδειγμα με τον, τον τρόπο με τον οποίο εγκρίθηκε, υιοθετήθηκε το νομοθέτημα για τις εκτρώσεις. Δεν είναι νομίζω το σωστό σημείο να αναφερθεί να συζητηθεί αυτό το θέμα το οποίο δεν πήγε όπως θα έπρεπε όμως σε όλα τα άλλα θέματα για αυτή την έκθεση θα πρέπει να πούμε ότι αυτά θα βρεθούν στο επίκεντρο μόνο αν δοθεί μια ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων για την Μακεδονία. Και το πιο σημαντικό είναι η έκκληση προς το Συμβούλιο να διαραγεί, να σπάσει ο φαύλος κύκλος που έχει επιβληθεί από την Ελλάδα με το πάγωμα των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι όπως οι συνάδελφοι τόνισαν, θα ήθελα και εγώ να επενέσω <clears throat> τις προσπάθειες του εισηγητή που επένδυσε τεράστιες προσπάθειες στην έκθεση αυτή. Πόσες φορές επισκέφθηκε αυτή τη χώρα και ξεκίνησε διάλογο και συνέχισε τον διάλογο για να προαχθούν συγκεκριμένα θέματα. Θα ήθελα λοιπόν να πω, κατά κάποιο τρόπο <clears throat> συμμετείχα και εγώ σε διάφορες συζητήσεις ε, σε σχέση με τα θέματα της έκθεσης που αφορούν τους γείτονες της Μακεδονίας και έχω την εντύπωση ότι κάπως τα έχω ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Είναι μια αίσθηση déjà vu και όσον αφορά το ψήφισμα και για την αντίδραση στην ε, Μακεδονία και λέει η κυβέρνηση εντάξει αξίζουμε να ξεκινήσουμε να ξεψίσα δεν πρέπει να αισθανόμαστε οποιασδήποτε ενοχές, ε, δεν είμαστε εμείς οι φταίχτες, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Ε, έτσι εξελίσσονται τα πράγματα στην πολιτική ζωή. Φυσικά υπάρχουν επικρίσεις, αλλά φυσικά επενώ εγώ τον εισηγητή, αλλά οι κανονικές αντιδράσεις είναι διαφορετικές. Λένε είναι όλα εντάξει με εμάς. Ε, όμως λόγω του θέματος της ε, ονομασίας ε, της χώρας μας ε, τα πράγματα παγώνουν και δεν προχωρούν. Και εδώ βρίσκεται πρόκληση για μας που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έγινε η προσπάθεια να επεξηγηθούν αυτά τα πράγματα επανειλημμένα. Είναι ενδιαφέρον, δεν υπήρξαν παρεμβάσεις Ελλήνων συναδέλφων. Όταν όμως ερχόμαστε στο κύριο θέμα κολλάνε τα πράγματα. Πάλι αποτελματώνονται. Πώς είναι δυνατόν η ονομασία, ένα όνομα να παρακολεί την επίτευξη προόδου δεν ναι. βλέπω κι εγώ τίποτα το διαφορετικό. Γιατί αυτή η κυβέρνηση εδώ και αρκετά χρόνια έχει μια εθνικιστική ημερήσια διάταξη. Δεν είδατε τι έγινε στο κέντρο των Σκοπίων με όλα αυτά τα μεγάλα μνημεία, γάλματα, ανδριάντες ε, ε, που ε, ξεκίνησε η κυβέρνηση και ανέγειρε η κυβέρνηση και λέγεται ότι δεν είναι δυνατόν ε, να γίνεται αυτό έναντι γειτόνων. Αυτό όμως δείχνει πόσο έχει τύχει χειραγώγηση η ιστορία περνώντας πίσω στη μεσαιωνική περίοδο, τη βυζαντινή περίοδο και στην σύγχρονη πάλι μετά εποχή και με την Βουλγαρία, παρότι προσπαθούμε να ασκήσουμε επικρίσεις και να πούμε γιατί διώκεται τους ε, Βουλγάρους οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι Βούλγαροι και όμως παρόλα αυτά τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα με αυτά τα θέματα. Εντάξει, και εγώ συμφωνώ, έχουν κολλήσει τα πράγματα, αλλά δούμε τι βρίσκεται πίσω από όλη αυτή την κατάσταση. Και σε σχέση και με τις διαπραγματεύσεις πέρσι, τι συνέβη. Η άλλη κυβέρνηση ήταν εκείνη η οποία είχε υιοθετήσει κάποιες ε, θέσεις. Τώρα έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Είναι κάποια θεμελιώδη πράγματα τα οποία θα μπορούσαν εύκολα να ε, ε, υλοποιηθούν από την ε, πλευρά της Μακεδονίας. Τι έχουμε, τρεις φορές ε, συναντήσεις, τρεις φορές όπου η μακεδονική πλευρά συνεχίζει να ε, προωθεί εντός εισαγωγικών διαλόγους και συναντήσεις χωρίς όμως να σημειώνεται καμία πρόοδος, χωρίς να γίνεται τίποτα. Όταν έχουμε ιστορικές προσωπικότητες σε σχέση με την ιστορία η θέση ήταν από πλευράς μας επικοδομητική από πλευρά σου όταν ότι εντάξει ας αφήσουμε αυτή την, ε, αυτό το ζήτημα, ας το ε, θέσουμε στο περιθώριο. Όμως η ε, μακεδονική πλευρά αρνείται να υιοθετήσει μια πιο επικοδομητική θέση. Ποιος θέλει λοιπόν και σε τι οφείλεται αυτό. Τώρα το αν θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις ή όχι, τρεις φορές και ίσως θα μπορούσαμε και 30 φορές να συναντηθούμε. Όμως αισθανόμαστε, διαισθανόμαστε ότι με αυτή την κυβέρνηση εκεί στα Σκόπια δεν υπάρχει καμιά βούληση να καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό. Όσον αφορά τον συμβιβασμό επί του ονόματος, ας παρέμβουν οι Έλληνες και ας πούν τις δικές τους τις απόψεις. Όμως εθνικιστικές απόψεις εξακολουθούν να είναι πολύ σταθερές Κάποιοι οι οποίοι υιοθέτησαν και οικοδόμησαν ε, την ιστεροφημία τους ε, με τοποθετήσεις κατά των Βουλγάρων κατά το παρελθόν, κατά τις τελευταίες 4-5 ε, δεκαετίες έχουν ακόμα επιρροή. Και εκείνοι οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε υιοθέτηση νέων θέσεων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους αντιμετωπίζουμε ακριβώς ένα πρόβλημα βλέπουμε σε σχέση με τους πολίτες μας. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις σε σχέση με τη Βουλγαρία, όμως οι θέσεις αυτές δεν αλλάζουν. Διότι αυτό θα μπορούσε ίσως στο μέλλον να περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα αν οξυνθεί. Γι' αυτό είπα ότι θα έπρεπε να συνεχίσουμε να επεξηγούμε και να διευκρινίζουμε περί τίνος πρόκειται και να λέμε ότι σε σχέση με τους Έλληνες, τους Μακεδόνες, τους Βουλγάρους δεν υφίστανται προβλήματα μεταξύ τους. Όμως υπάρχουν κάποιες πολιτικές θέσεις και τοποθετήσεις που υπονομεύουν τα πράγματα και διαρκώς δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ αυτών των λαών. Ευχαριστώ. Thank you, Chair. I'll try to be... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομο. Πιο σύντομο από ό,τι θα φαντάζεστε, για ένα πολύ απλό λόγο. Οι θέσεις που εξέφρασαν ο συνάδελφος Κύριλοφ από τη Βουλγαρία απόλυτα συμπίπτει με τη δική μου, αλλά θα προσθέσω κάτι σημαντικό. Σημαντικές λεπτομέρειες. Αν η Αλβανία είχε Πάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κοινοβούλιο. Να μην είχε προκαλέσει έκπληξη η σερβική θέση, η ελληνική θέση, η βουλγαρική θέση να συνέπιπτε σε κάποια από τα ανοιχτά θέματα, εκκρεμή θέματα. Οι Σέρβοι έχουν θέμα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ελβανία έχουν ε, θέματα με την ιστορία, οι Έλληνες με την ονομασία και οι Βουλγαροί. Γιατί, γιατί γίνεται αυτό στην ε, γωνία της, των Βαλκανίων αυτή. Γιατί αντιμετωπίζουμε, όπως είπε ο Ευγένη Κυρίλοφ, αντιμετωπίζουμε μια, ένα νέο έθνος, ένα πολύ νέο κράτος, το οποίο ε, δημιουργήθηκε τον Αύγουστο, τον Αύγουστο του 1944 και το έθνος και το κράτος. Άρα, τι θα κάνουμε στη συνέχεια, πώς ασφαλώς θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειες της μακεδονικής ε, κοινωνίας και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι αξίζουν την υποστήριξη, την προσοχή μας και την τεχνογνωσία μας για να προετοιμαστούν για την προσχώρηση στην Ένωση, αλλά για να είμαστε και επίμονοι και συνεπείς σε ό,τι αφορά τις συστάσεις μας. Καταρχάς, θα πρέπει να είμαστε λογικοί, να μην ε, προκαλούμε τους γείτονες. Αυτή η ιδέα να ξεκινήσουν, να ανοίξουν τα κεφάλαια και ιδιαίτερου το 23 και το 24. Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα πληρούν τους όρους που προβλέπονται στα κεφάλαια στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αν δεν πληρούν τους πιο απλούς όρους των παραγράφων που ήδη έχουν ενταχθεί στα προηγούμενα ψηφίσματα και τις προηγούμενες εκθέσεις. Μία από τις παραγράφους αυτές ορίζει ότι πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να συμμετάσχουν σε κοινέ ε, εορτασμούς κοινών εορτασμών. Τον Οκτώβριο ε, προκάλεσαν ε, ομάδα Αλβανών Βουλγάρων στην περιφερειά τους ότι οργανώθηκε ένα σεμινάριο λόγω της επαιτίου του 1913 κατά των Σέρβων. Μποϊκοτάρισμα ήταν η το απάντηση των ε, θεσμικών οργάνων τους στα Σκόπια. Κάποιες μέρες αργότερα η επίσημη Ακαδημία, η Μεκατονική, διοργάνωσε εναλλακτικό σεμινάριο. Αν ακολουθήσουν λοιπόν αυτό το δρόμο, προφανώς δεν ε, εκπληρώνουν τους όρους και τις δεσμεύσεις που έχουν κάνει προς το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τα ψηφίσματα που ήδη έχουν εγκριθεί. Παραγράφους γνωστές στα ψηφίσματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι ανοίγοντα τα κεφάλαια αυτά θα καλύψουν όλα αυτά τα θέματα. Τελευταίο σημείο. Στο σημείο 15 αναφέρεται το θέμα του πολιτικού μητρώου, του αστικού μητρώου. Βοηθήστε με λίγο. Τι εννοούμε. Μιλάμε για μια εναλλακτική λύση για την απογραφή. Θα καταργήσουμε την διαδικασία της απογραφής και θα εξαρτηθούμε από τι, από μια καταγραφή στα αστυνομικά τμήματα, στους Δήμους. Αυτό δεν να σας πω περίεργο με πάσα ειλικρίνεια, ας πούμε ότι η απόγραφη δεν μπορεί να γίνει στη Μακεδονία γιατί θα είμαι διπλωματικός για οικονομικούς λόγους. Α, αλλά να πούμε, να μιλήσουμε για ένα μητρό, αυτό θεωρώ ότι δεν λειτουργεί. Σας ευχαριστώ να είμαστε πιο συνεκτικοί. Εκτός μικροφώνου σχόλια του Πρόεδρου. Δεν ξέρω, πρόεδρε γιατί το λέτε αυτό. Βρίσκω ότι πραγματικά θα έπρεπε να σταματήσει η επίκριση της Μακεδονίας, η επικρίση στη Μακεδονία. Κάθε χώρα έχει τις ελλείψεις της, κάθε χώρα έχει τις προόδους που έχει σημειώσει. Η Μακεδονία έκανε μεγάλες προόδους, έχει το καλύτερο δίκαιο προστασίας μειονοτήτων στα Βαλκάνια και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ήταν ένα από τα πρώτα κράτη η Μακεδονία που πήραν το το καθεστώς υποψήφιας ε, ε, χώρας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό εγκρίθηκε τότε. Δεν μπορεί λοιπόν να πει κανείς ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Ε, δεν οφείλεται στην πρόοδο της Μακεδονίας, οφείλεται στο θέμα της ονομασίας. Το γνωρίζουν όλοι. Το γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο επί πολλά χρόνια με μεγάλη πλειοψηφία ζητούσε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Μακεδονία. Και το λέω με κάθε σαφήνεια. Αν το Δεκέμβριο το Συμβούλιο δεν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Μακεδονία, αλλά τις ξεκινήσει με τη Σερβία, ε, τότε λοιπόν θα δημιουργηθεί εντύπωση και θα ενδυναμωθεί η εντύπωση στα Βαλκάνια ότι δεν είναι κοινότητα δικαίου με αντικειμενικά κριτήρια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι μια ασίδωτη, αυθαίρετη κοινότητα, όπου κάποιος που τροχοπεδεί τα πράγματα με αρνησή κυρία μπορεί να επιβάλλει τις θέσεις του είτε αυτές οι θέσεις είναι δικαιολογημένες είτε όχι. Αυτό είναι το επικίνδυνο μήνυμα σε αυτή την περίπτωση προς τη Μακεδονία. Φυσικά πρέπει να είναι σεβαστά τα κριτήρια, αλλά τα κριτήρια υλοποιούνται καλύτερα από τη Μακεδονία από ότι σε σχέση με τις περισσότερες χώρες με τις οποίες ασχοληθήκαμε απόψε και με τις οποίες ασχολούμεθα ο ήθιστε στα Βαλκάνια με τις χώρες αυτές. Και το λέω ξεκάθαρα, είναι σκάνδαλο, σκανδαλώδες το πώς αντιμετωπίζουμε αυτή τη χώρα εμείς. Έχω πάρα πολύ μεγάλες ανησυχίες για αποσταθεροποίηση της Μακεδονίας. Κύριε Κυρίλοφα, αυτά τα οποία είπατε είναι το άκρο ναότον του κινησμού. Το να λέτε δηλαδή ότι ε, απλά και μόνο σημειώνεται η περίπτωση αυτή, αντίθετα βρίσκονται σε απόγνωση και τίποτα δεν μπορεί να γίνει γιατί πρόκειται για αυθαίρετη στάση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά και το ΝΑΤΟ με την αρνήση κυρία κάποιων. Και εν συντομία τρεις παρατηρήσεις. Όπως και ο συνάδελφος πιστεύω και εγώ το θέμα των εκτρώσεων δεν ανήκει, δεν πρέπει να εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Δεν ανήκει στο πλαίσιο νομοθετικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανήκει στην επικουρικότητα ως θέμα. Τα ιστορικά θέματα δεν μπορούν έτσι με μονοκοντιλιά να επιληθούν. Παράδειγμα, η Τσεχία, η δημοκρατία της Τσεχίας κρίμα που ο Τσέχος συνάδελφος δεν είναι εδώ, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων είχε ανεγείρει μνημεία υπέρ του, Ντε, του Μπένες, με τα διατάγματα Μπένες και Τρία εκατομμύρια Σουδητών Γερμανών απέλασε, εξετόπισε ο Μπένες μεταξύ αυτών ε, και οι πρόγονοί μου, οι παππούδες μου, οι συγγενείς μου και για τα θέματα των Σουδητών Γερμανών ε, υπάρχουν ιστορικές ρίζες όμως αυτός ο διάλογος είναι εφικτός μόνο αν υπάρχει γειτονική εταιρική σχέση και συνεργασία και είμαι υπέρ αυτής και τέλος η εξωτερική πολιτική της Μακεδονίας είναι ιδιαίτερα επικοδομητική Θέλω να υπενθυμίσω την διαδικασία που από πλευράς Προέδρου Ιβάνοφ ξεκίνησε όπου οι πρόεδροι των, ε, της Μακεδονίας, της Αλβανίας, του Κωσυφοπεδίου και Μαυροβουνίου συνέρχονται εκ περιτροπής κατά το πρότυπο των χωρών Βίσεγκραντ. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα όπως έγινε με κάποιες παρεμβάσεις, μόνο με επικρίσεις της Μακεδονίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ θερμά. Είναι μια διαρκώς επαναλαμβανόμενη ιστορία αυτή που διαρκεί ε, συνεχώς. Εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται και εμπλέκονται και εκείνοι οι οποίοι διαρκώς ε, οργίζονται σε σχέση με κάποιους γείτονες υπήρξε συζήτηση σε σχέση με τους Έλληνες, τώρα υπάρχει θέμα υποσυζήτηση με τους, ε, σε σχέση με τους Βουλγάρους και τους Έλληνες και υπάρχουν και θέματα και με την Αλβανία. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Πρέπει κάποια πράγματα να κατονομαστούν. Κύριε Χάουιτ, σας δίνω τον λόγο σύντομα παρακαλώ. <clears throat> Και υπό το επόμενο έχουμε ένα σημαντικό σημείο, υπό το 10 για τις ε, ε, τις συστάσεις ε, όσον αφορά την εκδήλωση για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Είναι όλα όσα ανέφερε ο κύριος Πόσελ πολύ σωστά. Είναι καλές οι συμφωνίες, αλλά ακούγονται διαρκώς ανησυχίες για την εφαρμογή τους στην πράξη, στην πρακτική ζωή, καθημερινή ζωή. Και υπάρχουν εδώ αυτές οι πτυχές. Και ίσως θα έπρεπε πιο, με μεγαλύτερη σαφήνεια να τοποθετηθούμε για αυτά τα θέματα. Κάπως αποκρύπτονται κάποια πράγματα ή αποσιωπούνται και για την κατάσταση όπως δημιουργείται η διακρύβωση του τι συμβαίνει με, με την πλειοψηφία στην Μακεδονία θα πρέπει ιδιαίτερα έντονα να τύχει της προσοχής μας. Ένα τρίτο του πληθυσμού είναι μειονότητες που δεν ανήκουν σε αυτή την ταυτότητα των εντοσαγωγικών Μακεδόνων, Σλαβομακεδόνων. Είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να αντιμετωπιστεί. Έχετε τον λόγο κύριε Χάουιτς. Θα ολοκληρώσω σε τρία λεπτά Χαίρομαι ιδιαίτερα που κάναμε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ κύριε Κλουκάν για την ε, συνεργασία μας. Νομίζω ότι αυτό σε πολύ τη συγκεκριμένη πολιτική, το συγκεκριμένο τομέα. Δεν ε, σχολίασα συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τη χειρονομία του κυρίου Φιούλη και σε ό,τι αφορά το θέμα ε, του ονόματος και για την διαπραγματεύση. Σύμφωνο απόλυτα και το, να, να μπει αυτό στο πρακτικά. Συμφωνώ και με αυτό που είπατε για την επιστοδρόμηση σε θέματα αξιοπιστίας και το γεγονός ότι το λέτε εσείς. Αυτό νομίζω ότι δίνει ένα χαρακτηριστικό ε, μήνυμα σε όσους μας ακούν σε ό,τι αφορά τον κύριο και Είπατε ότι μας χωρίζει ούτε ένα συγκαρόχαρτο γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά, ταυτίζονται οι απόψεις μας. Ε, θα ήθελα να πω ότι καταλαβαίνω το θέμα του ονόματος. Όταν λέει ο κόσμος ότι είναι ακατανόητο το θέμα αυτό, εγώ πρέπει να σας πω ότι το καταλαβαίνω και το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ε, βαθιά ε, ριζωμένες απόψεις που μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε και ήμουν πάντα πολύ προσεκτικός αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση και στις δύο πλευρές, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε το βάθος των συναισθημάτων μας. Θα ήθελα να πω ότι εγώ το έχω κάνει σε ό,τι αφορά την παραγράφο 24 για την αναπαραγωγική υγεία. Ήμουν πάρα πολύ προσεκτικό στη διατύπωση για να μην σχολιάσω αν ο νόμος ήταν καλός ή κακός. Καταλαβαίνω τι λένε οι συνάδελφοι ότι αυτό δεν είναι δικαίωμα του κοινοβουλίου μας και θεωρείται... Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ προσεκτική η διατύπωση του 24 τι λέω ότι θα πρέπει το κοινοβούλιο της χώρας να ακολουθήσει τις διαδικασίες τις κοινοβουλευτικές και δεν έχει γίνει αυτό. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς η δημοκρατία, η κοινοβουλευτική δημοκρατία θα πρέπει να ενδυναμωθεί. Άρα θεωρείτε ή μπορεί να μην θεωρείτε ότι ο τρόπος είναι σωστός. Αλλά το θέμα είναι ο τρόπος που πέρασε το θέμα αυτό. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κύριλοφ για τις καλά σου, τα καλά σας λόγια και συμφωνώ σε ό,τι αφορά την επαφή με τον, τον κόσμο, τους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λέτε ότι η κυβέρνηση διατείνεται ότι είναι όλα καλά. Να είμαστε δίκαιοι. Δεν το λέει αυτό η κυβέρνηση, για να είμαι ειλικρινής. Κατανοούν τις προκλήσεις, υπάρχουν ανταλλαγές, γίνονται συζητήσεις σε ό,τι αφορά... Συγγνώμη πρόεδρε που ώρα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα ότι οι προκλητικές ενέργειες είναι πραγματικά επιζήμιες. Το αναφέρω διαρκώς αυτό στη χώρα και στους ε, συνομιλητές μου, το λέω ασφαλώς και στους συναδέλφους εδώ. Θα έλεγα σε ό,τι αφορά το πνεύμα των συναντήσεων και την πρόοδο που έγινε και να σας πω τι μου είπε και ο βούλγαρος πρέσβης στα Σκόπια. Ούτε αυτός είπε ότι είναι όλα τέλεια, αλλά θεωρώ ότι αποτυπώνει το πνεύμα που επικρατεί. Θεωρώ ότι υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ της βουλγαρικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης στα Σκόπια για το ποια α, περιστατικά, ποιοι εορτασμοί θα πρέπει να υπάρξουν. Θα πρέπει λοιπόν ε, και στις δύο πλευρές να βρουν κάποιους κοινούς εορτασμούς και μετά να εξελιχθεί η κατάσταση. Και τι λέω στους Βουλγάρους συναδέλφους, πέρσι με τεράστιο ρυθμό Βούλγαρων ε, ε μερών, είχα, τα πάρα πολύ τα Βούλγαροι, ήταν πραγματικά δυσανάλογη αυτή η εκπροσώπηση. Να είναι επίσης επικοδομητική διατύπωση, να πούμε τι θέλουμε με θετικό τρόπο, με αισιόδοξο τρόπο, όχι να καταδικάζουμε μόνο, αλλά ασφαλώς αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και ιδιαίτερως και Είμαι βεβαίως ότι είστε διατεθειμένοι να το κάνετε αυτό σε ό,τι αφορά την, τα αίτια και την ιδέα ότι δεν εφαρμόζονται οι όροι. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι απλά αυτά που το ζητούμε να εφαρμόσουν. Θεωρώ ότι είναι περίπλοκα. Είναι περίπλοκα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τους όρους αυτούς. Τρία τελευταία ζητήματα. Κύριε Πόσελτ, συμφωνώ απόλυτα αυτά που λέτε για τα θέματα ιστορίας και καλωσορίζω αυτά που είπατε σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, το παράδειγμα στο Κομινόβο όπου υπάρχει θα θυμάστε από τις προηγούμενες εκθέσεις μας ότι ζητήσαμε από τις τοπικές επιτροπές να εφαρμόσουν την συμφωνία πλαίσιο και να τη θέσουν, να την καταστήσουν λειτουργική. στις τροπολογίες φαντάζομαι θα τεθούν διάφορα θέματα σε ό,τι αφορά την Συμφωνία της Οχρίντας και τη δεύτερη φάση εφαρμογής αυτής και προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση και να, ξεκινήσουν, να ξεκινήσει η εφαρμογή των ε, όρων αυτών. Συμφωνώ λοιπόν με την άποψή σας στο θέμα αυτό και αυτό θα το σκεφτούμε στο τελικό κείμενο του Κοινοβουλίου. Έχετε την υποστήριξή μου σε ό,τι αφορά τα θέματα που αναφέρετε. Ευχαριστώ λοιπόν και εσάς και όλους τους συναδέλφους που συνεργάζονται μαζί μου για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ θερμά. Έχουμε την προθεσμία 10 Δεκεμβρίου 18.00 το βράδυ. Αν συμφωνείτε, ολοκληρώνεται η συνεδρίαση επ' αυτού. Και χαίρομαι που μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι η Επίτροπος Γεωργίευα <clears throat> μπόρεσε να έρθει σε μας. Χαίρομαι για το ότι σε αυτή τη συνεδρίαση θα έχουμε εκπροσώπους και της Επιτροπής Ανάπτυξης ε, ανάμεσά μας και την κυρία Εύα Ζολή. Μια κοινή συνεδρίαση με κοινή πρωτοκαθεδρία, προεδρία από πλευρά της ε, κυρία Εύα Ζολή, τις ευθύνες σας ε, για την χρηματοοικονομική βοήθεια και συνδρομή, δίνοντας απάντηση στα ζητήματα που αυτή τη στιγμή απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και δουλειά από εσά με τους τυφώνες στην, στις Φιλιππίνες, με τα όσα τεκταίνονται στην κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, για να αναφέρω μόνο κάποια από τα πολλά θέματα καθίσατε σαφές όταν βλέπουμε και πόσοι στη στην Συρία μυριάδες ε, έχουν υποστεί πλήγματα, λιμοκτονούν, πόσοι βρίσκονται εκτοπισμένοι εκτός ε, Συρίας και πόσοι είναι οι εκτοπισμένοι εντός Συρίας. Είναι τεράστιες οι ανάγκες για την ανθρωπιστική βοήθεια και όλα αυτά είναι θέματα τεράστιας εμβέλειας ε, και θέματα χρηματικής συνδρομής επίσης, χρημάτων, κονδυλίων, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είμαι ευγνώμων για όλους αυτούς τους λόγους που μπορείτε να μας παρουσιάσετε αυτή την κατάσταση και τα προβλήματα τα οποία αναφύονται και που υπάρχουν ανάγκες να δράσουμε και τι μπορεί να γίνει. Αλλά επίσης και είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια να δοθεί, αλλά και να υπάρξει πολιτική σταθεροποίηση, να αντιμετωπιστεί η αποσταθεροποίηση. Είναι διτό το πρόβλημα και έχει και στρατιωτική πτυχή. Και έτσι λοιπόν οι δύο μας επιτροπές ε, παρακολουθούν ε, ιδιαίτερα το έργο το οποίο αναπτύσσεται. Θα ήθελα ε, να παρακαλέσω να παρέμβετε εσείς παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Κυρία Επίτροπε, με μεγάλη χαρά σας ε, υποδεχόμαστε στην κοινή συνεδρίαση αυτή ΑΦΕΤ και Επιτροπής Ανάπτυξης για τη Συρία και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Στην Επιτροπή Ανάπτυξης τον Αύγουστο κάναμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Έκτοτε βέβαια έχει επιδεινωθεί η κατάσταση και στις δύο χώρες και περιμένω λοιπόν να σας ακούσω με ανυπομονησία για να δούμε που βρισκόμαστε σήμερα. Είμαι πολύ ανήσυχη από τις δυσκολίες που υπάρχουν, αν όχι, από την, αδυναμίες για τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις να έχουν πρόσβαση στη Συρία και να δώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Σε ορισμένε ε, περιοχές της χώρας χρησιμοποιείται ο λοιμός ως πραγματικό όπλο. Τώρα, αυτό που ονομάζουμε ξεχασμένη κρίση ε, στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Από τότε που οι αντάρτες σε λέκα ε, την περασμένη άνοιξη ανέτρεψαν την κυβέρνηση, έχει επανέλθει στην επικαιρότητα. Και η χώρα και τα 5 εκατομμύρια φτωχών κατοίκων ε, έχουν να αντιμετωπίσουν, εκτός από τη φτώχεια, την τεράστια ακυβερνησία και το τρομακτικό ανθρωπιστικό πρόβλημα. Ξέρω, κυρία Επίτροπη, ότι είσαστε εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσετε στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο την κρίση αυτή. Από τότε που έγινε το πραξικόπημα στο τέλος του περασμένης χρονιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε στις περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες για να προσπαθήσει να σταθεροποιήσει τη χώρα και την κυβέρνησή της. Δυστυχώς οι προσπάθειες αυτές δεν άρχισαν και ο ΙΕ, η Γαλλία, οι Ηνωμένε Πολιτείε όλοι ε, αναγνωρίζουν τον άμεσο κίνδυνο γενοκτονίας. 20 χρόνια μετά την Ρουάντα Πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε μια νέα γενοκτονία στην Αφρική και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια πολιτική λύση. 6.000 κιανόκρανοι μπορούν να μεταβούν στην Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία. Η Γαλλία έχει περισσότερους στρατιώτες και θα μπορούσε να στείλει 1.000 με 1.500 στρατιώτες. Αν αυτές οι παρεμβάσεις μας επιτρέψουν να βγούμε από την πολιτική και ασφαλιστική κρίση, δεν λύνουν παρόλα αυτά το πρόβλημα στη ρίζα του, που είναι η τεράστια φτώχεια. Ε, υπάρχει ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη χώρα αυτή. Πρέπει να ε, ενισχύσουμε την ε, βοήθειά μας για να υπάρξει ε, σταθερή δημοκρατική κατάσταση και για μια χώρα που είναι η εκατοστή, ογδοικοστή σε, στον κατάλογο φτώχεια σε 187 χώρες. Η πολιτική ε, κρίση είναι έντονη, η ανθρωπιστική κρίση είναι έντονη. Οι σημερινές ευρωπαϊκές δυσκολίες δεν πρέπει να μας κάνουν να κλείσουμε τα μάτια στις ανθρωπιστικές κρίσεις που υπάρχουν στις Φιλιππίνες, στο Νεπάλ, από όπου μόλις επέστρεψα, στη Συρία, στην Κεντροαφρικανική ε, Δημοκρατία. Ε, στο, στην τελευταία χώρα υπάρχει πέρα από την ανθρωπιστική κρίση και κίνδυνο γενοκτονία. Πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει για να την αποφύγουμε. Γιατί είναι κατεπήγον το πρόβλημα. Κυρία Γεωργίευα, σα καλωσορίζω και είμαι πεπισμένη ότι αυτή η συζήτηση θα είναι επικοδομητική. Κυρία Γεωργίευα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπρόκ, ευχαριστώ κυρία Ζολή που παρουσιάσατε το θέμα αυτό που κάνετε την εισαγωγή για την κρίση στη Συρία και την κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Μιλάμε για δύο χώρες, για δύο συγκρούσεις που διαφέρουν από πολλές απόψεις. Στη Συρία έχουμε μια ανθρωπιστική καταστροφή, την πιο δραματική των τελευταίων δεκαετιών, το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης δίνουν μεγάλη έμφαση σε αυτό που συμβαίνει στις, στη Συρία και από την άλλη έχουμε μια άλλη χώρα, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, που είναι το σύμβολο της ξεχασμένης κρίσης. Για να πω ξεχασμένη χώρα. Αυτές οι δύο χώρες όμως και αυτές οι δύο κρίσεις μοιάζουν πολύ παρόλα αυτά σε ό,τι αφορά την κλίμακα της, του προβλήματος, στην περίπτωση της Συρίας Έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα τα οποία έχουν επηρεαστεί και χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Στην περίπτωση της ε, Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, από τα 4,6 εκατομμύρια του πληθυσμού, ε, μπορώ να πω ότι και τα 4,6 επηρεάζονται από την ε, κρίση. Και υπάρχει πιθανότητα να αποσταθεροποιηθεί ολόκληρη περιοχή και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Επίσης μπορούμε να διδαχτούμε πολλά και στι δύο περιπτωσει ε, από το τι συμβαίνει αν δεν δράσουμε εγκαίρω ω διεθνής κοινότητα. Πριν πω στι λεπτομέρειες των δύο αυτών ε, προβλημάτων, μια και ανέφερε ο κύριος Μπρόκ της Φιλιππίνες και τον α, ε, τυφώνα Χαϊάν, θα ήθελα να σας πω πολύ σύντομα ότι πραγματικά η κατάσταση είναι δραματική η φυσική καταστροφή, ήταν απίστευτη, αλλά όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έδρασε έγκαιρα, γενναιόδωρα και με πραγματικά συντονισμένο τρόπο. Πήγα στις Φιλιππίνες, ε, στο Τακλομπάν, στις 16 Νοεμβρίου, μία εβδομάδα μετά τον τυφώνα και φτάσαμε με ένα μικρό, μικρό ελικόπτερο, πετάξαμε πάνω από τις ε, πληγήσεις περιοχές. Ήταν απίστευτο το θέαμα και έβλεπε τη διαφορά ανάμεσα στην, στο, στις περιοχές που δεν τις επηρέασε ο τυφώνας και τις ε, περιοχές που πλήγησαν από τον τυφώνα. Ήταν η διαφορά ανάμεσα στον παράδεισο και στην κόλαση. Ό,τι ακριβώς έκανε το τσουνάμι, ό,τι έκανε ο σεισμός στην Ναϊτή. Αισθάνθηκα συμπόνια για τον κόσμο γιατί το αποτύπωμα της καταστροφής είναι τόσο μεγάλο που να, το να δοθεί βοήθεια σε όλους δεν ήταν καθόλου εύκολο. Επίσης αισθάνθηκα ότι ως Ευρωπαίοι δείξαμε ακόμα μια φορά πόσο αλληλέγγυοι είμαστε με άλλα έθνη στις πιο δύσκολες στιγμές που περνούν. Το Σάββατο, την επόμενη του τυφώνα, πήγε μια ομάδα. Η πρώτη ομάδα αξιολόγησης ε, από το εξωτερικό που πέταξε στις Φιλιππίνες και αποφασίσαμε δύο μέρες μετά, την Κυριακή, ε, για χορήγηση κονδυλίων. Η πρώτη απόφαση. Επίσης, μια ομάδα βελγική πολιτική, πολιτικής προστασίας ε, πήγε στο Τακλομπάν τρεις μέρες μετά τον τυφώνα. Η πρώτη διεθνής ομάδα που έδωσε ιατρική βοήθεια και καθαρισμό του νερού. Εν συνεχεία Πήγε και μια γερμανική ιατρική ομάδα που εντάχθηκε εκεί. Έχουμε δώσει παραπάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ βοήθειας, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 15 κράτη-μέλη έχουν δώσει και βοήθεια σε είδος και ομάδες ούτως ώστε να βοηθήσουν να συντονίσουν την βοήθεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ήταν η πρώτη φορά που ανταποκριθήκαμε μετά τη δημιουργία του Συντονιστικού Κέντρου Επίγουσας Βοήθειας και η ικανότητα να συντονίσουμε την ευρωπαϊκή βοήθεια είναι πάρα πολύ ορατή. Αποφύγαμε το, τον κίνδυνο το να βοηθήσουμε κάποιου δύο φορές και κάποιους να τους ξεχάσουμε εντελώ. Εσείς προέρχεστε από διαφορετικές χώρες. Θέλω να πω σε όλους τους Ευρωπαίους ότι είμαστε πραγματικά εκεί που μας χρειάζονται. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Ας πάω τώρα όμως ε, στο θέμα μας, που είναι η Συρία και η κεντροαφρικανική δημοκρατία, για το πολιτικό πλαίσιο. Ξέρετε ότι έχουμε μια ημερομηνία για το Γενέβα 2, 22 Ιανουαρίου. Και ευελπιστούμε ιδιαίτερα από πλευρά τη κοινότητά μα ότι αυτό θα οδηγήσει στο να ανοίξει μια δίωδο για την ειρήνευση. Όμω από την άλλη πλευρά είναι απόλυτα σαφές ότι ακόμα και αν στεφτεί με επιτυχία η Γενέβη 2 την επόμενη κιόλα ημέρα, οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις και συνέπειες θα είναι τόσο σοβαρές και τέτοια εμβέλειας που θα οδηγηθούμε μέσα στο 2014 και ακόμα στο 2015 μέχρι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανθρωπιστικές συνέπειες αυτής της κρίσης. Και ιδιαίτερα ανησυχούμε για τρία θέματα, για τρεις άξονες. Το πρώτο θέμα είναι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης εντός της ίδιας της Συρίας, αποδυναμώνοντας ε, τον πληθυσμό που έχει υποστεί τόσα πλήγματα, αλλά καθιστώντας και τόσο δύσκολο τόσο περίπλοκο και δυσχερές το να παρασχεθεί, να δοθεί ανθρωπιστική σύνδρομη. Εξακολουθεί και είναι μείζον πρόβλημα η πρόσβαση, η προσπελασιμότητα στη Συρία. Και εμεί ε, πιστεύουμε ότι αν δεν υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την πρόσβαση στον πληττόμενο ε, πληθυσμό της Συρίας, όχι μόνο περισσότεροι πολίτες ε, θα πληγούν, αλλά και περισσότερα παιδιά και πολίτες θα αποβιώσουν τελικά και η η δυνατότητα αυτή θα έπρεπε να μπορέσει να εξεταστεί από αυτό το πρίσμα μέσα σε ένα επιταχυμένο και διευρυμένο πλαίσιο. Και πρέπει να δοθεί η βοήθεια, η συνδρομή στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, τις ε, γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους. Για το θέμα των παιδιών ακριβώς. Τώρα <clears throat> αντιμετωπίζουμε μια φρικτή αποτροπιαστική πραγματικότητα Δηλαδή σε σχέση με τα όσα είχαμε δει να ε, συμβαίνουν στην ε, Σομαλία. Μία ολόκληρη γενεά δηλαδή εξοντώνεται, ε, έχει καταδικαστεί και η απώλεια των, των παιδιών που σκοτώνονται από τις σφαίρες αλλά επίσης αντιμε... πεθαίνουν από οι άσημες ασθένειες αλλά και από την ίδια την πείνα και χάνουμε εδώ τεράστιες ευκαιρίες σε μια χώρα που συνήθιζε να έχει ελεύθερη πρόσβαση προς πελασιμότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα. 97% των αγοριών, 96% των κοριτσιών μπορούσαν να πηγαίνουν στο σχολείο παλιότερα. Τώρα 2,5 εκατομμύρια παιδιά δεν πάνε πια στο σχολείο. Και μεταξύ των προσφύγων ο αριθμός έχει αυξηθεί, έχει αυξηθεί σε 2,2 εκατομμύρια. Δύο τρίτα των παιδιών σε σχολική ηλικία βρίσκονται εκτός σχολείων έρημα και ανησυχούμε πάρα πολύ για τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης ε, ιδιαίτερα σε άλλες χώρες, γειτονικές χώρες, ε, στον Λίβανο και την Ιορδανία. Και ο κίνδυνος που υπάρχει να αποσταθεροποιηθούν αυτές οι χώρες με ενδυνάμει τρομακτικές επιπτώσεις για τους πολίτες αυτών των χωρών, τους Λιβανέζους και τους ε, κατοίκους της Ιορδανίας, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο ευρύτερα. Κάνουμε λοιπόν υπολογισμούς και λέμε ότι η αύξηση των προσφύγων στην περίπτωση της κατάρρευσης του Λιβάνου θα μπορούσε πραγματικά ο Θεός να ε, οδηγήσει να μην φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Προσευχόμαστε να μην γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο και υπάρξει τέτοια κατάρρευση, τότε ο κίνδυνος ενός τεράστιου μεταναστευτικού ρεύματος από αυτή τη χώρα προς την Ευρώπη πραγματικά εντείνεται. Και προς τη δική μου χώρα, την Βουλγαρία, υπάρχει μεταναστευτικό ρεύμα και υπάρχει σημαντική αύξηση προσφύγων που περνούν τα σύνορα την Παρασκευή. Αποκινούμε τον, τον ύπατο εκπρόσωπο για τους πρόσφυγες των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουτέρες, διασφαλίσαμε ότι θα έπρεπε να κινητοποιηθεί όλη η δυνατότητα συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από την ύπατη αρμοστία των ΗΠΑ για τους πρόσφυγες για να αντιμετωπίσουμε τις ε, πιο έντονες ανάγκες. Τι βλέπουμε κάνοντας ε, υπολογισμούς ε, και σκιαγραφώντας το τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον. Δεν είναι δυνατόν να πω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Δεν υπάρχουν θετικές προοπτικές. Δεν υπάρχουν βελτιώσεις ε, σχετικά. Έχουμε μια σταδιακή επιδίνωση. Δηλαδή τα όσα έχουν ήδη σημειωθεί και είναι ήδη αρνητικά επιδεινώνονται με βραδείς ρυθμούς βέβαια. Όμως μπορεί να έχουμε και ταχύτερη, ταχύτατη επιδείνωση λόγω απρόβλεπτων εξελίξεων για παράδειγμα στην ίδια τη Συρία, εντός Συρίας ή όπως προανέφερα το τι θα μπορούσε να συμβεί με τον Λίβανο. Αν δεν αντέξει ο Λίβανος και δεν μπορέσει να υποστεί αυτή την αυξημένη πίεση από τα αυξημένα αυτά μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα. Τι θα συνέβαινε. Λοιπόν βλέπουμε τεράστιες ανάγκες ανθρωπιστικές υπάρχουν και θα υπάρχουν για το 2014. Τίθεται το ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Οι δράσεις μας επικεντρώνονται σε τέσσερις άξονες ο πρώτος ε, άξονας. Να συνεχίσουμε να συλλέγουμε τα κονδύλια εκείνα που είναι αναγκαία να βοηθηθούν οι πολίτες στην ίδια τη Συρία και στις γειτονικέ χώρες. Διαθέσαμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή της ε, σύνδρομης. Περίπου το ίμιση για τους εντός Συρίας ε, ευρισκόμενους και το άλλο ίμιση για εκείνους που ευρίσκονται στις γειτονικές χώρες και έχουν εκτοπιστεί εκεί. Επίσης συμπεριλαμβάνεται η σύνδρομη, η υποστήριξη για τις ε, λιβανέζικες και ιορδανικές κοινότητες ε, που, είναι, ε, που έχουν υποδέχονται τους πρόσφυγες αυτούς και καταβάλουν προσπάθειες να τους περιθάλψουν. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Στις 18 Δεκεμβρίου θα έχουμε μια συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, μια συνεδρίαση που έχει στόχο να κινητοποιήσει όλους, εμάς και άλλους, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες κατά το 2014 που θα είναι αυξημένες. Και δεύτερον, επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στην ε, προσπάθεια να υπάρχει προσπελασιμότητα, πρόσβαση σε αυτούς τους πληθυσμούς. Βρισκόμαστε ως προπομπή, ως πρωτοπόροι, διεκδικώντας και απαιτώντας ε, εκείνοι που μπορούν να ανασκήσουν επιρροή στους ε, αντιμαχόμενους, να ασκήσουν αυτή την επιρροή τους, για να υπάρξει δυνατότητα πρόσβαση προσπελασιμότητας στα άτομα τα οποία έχουν τέτοιες ανάγκες έχουμε μια δήλωση αλλά δεν υπάρχει ένα δεσμευτικό ακόμα πλαίσιο ε, ψηφίσματος που να διασφαλίζει αυτή την πρόσβαση. Και πρέπει να γίνει αυτό, διότι τα χρήματα δεν βοηθούν κανέναν αν δεν υπάρχει πρόσβαση στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δεν μπορεί κανείς να φτάσει σε αυτούς, η βοήθεια δεν φτάνει σε αυτούς. Πρέπει να δούμε επίσης, ε, να βρούμε τρόπους για να επιτύχουμε πιο αποτελεσματικό συντονισμό για την παροχή της ε, βοήθειας αυτής ε, με τα Ηνωμένα Έθνη και την ευρύτερη ανθρωπιστική κοινότητα αλλά και αυτό το οποίο αποκαλούμε υψηλή ομάδα υψηλών αξιωματούχων η υψηλή ομάδα ε, υψηλών αξιωματούχων που συναπαρτίζεται από εκπροσώπους από τις χώρες της περιοχής, από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να καταβληθούν συλλογικές προσπάθειες με συντονισμένο τρόπο για να είμαστε αποτελεσματικοί. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της αύξησης και έντασης ε, της εμπλοκής μας, και σε σχέση με την ε, εκπροσώπησή μας που είχε το, τα γραφεία μας είχαν κλείσει στη Δαμασκό και πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούμε Έχουμε μπροστά μας το πρόβλημα μιας χαμένης γενεάς, το πρόβλημα αυτών των παιδιών που εξοντώνονται. Από κοινού με την UNICEF, UNICEF ξεκινήσαμε μια πρωτοβουλία να μην χαθεί αυτή η γενεά, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, να βοηθηθούν τα παιδιά, αλλά και να εργαστούμε υπέρ της δικής μας ασφάλειας για να είμαστε ειλικρινείς. Διότι η ριζοσπαστικοποίηση, η ε, ακραία αυτή ε, κατάσταση που δημιουργείται στην ε, Συρία δεν είναι κάτι το οποίο θα διασφαλίσει μελλοντικές προοπτικές αλλά υπονομεύει τις προοπτικές για την ασφάλεια. Βασιζόμαστε πάντα στην δική σας υποστήριξη διότι θα είναι πραγματικά μια πολύ σκληρή μάχη αυτή που θα πρέπει να δώσουμε και μια πραγματικά ε, θα πρέπει να διαβούμε ε, άνυδρη και έρημη χώρα για να τα καταφέρουμε. Και όπως αναφέρθηκε από την κυρία ε, Ζολή, ε, με την πρώτη φορά και με τον ε, Υπουργό ε, Εξωτερικών της Γαλλίας κύριο Φαμπιούς είχαμε αναλάβει πρωτοβουλίες αλλά και στο παρελθόν επίσης μια άλλη φορά είναι μια ας το πω έτσι σύραξη που ε, λησμονήθηκε επί υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα και αγνοήθηκε από την παγκόσμια κοινότητα. Αυτό το οποίο ήταν μια κρίση στην αρχή, μια, το ξέσπασμα μιας κρίσης έγινε μια τραγωδία με πραγματικά τραγικές ε, ε, διαστάσεις ε, και έχει καταστρέψει και ματοκυλήσει τη χώρα. Αυτό που είδα είναι ένα τσουνάμι λαιλασιών και βιοπραγιών πολίτες ε, Σύριοι που κρύβονται ε, στα δάση στους θάμνους ε, που βρίσκουν για να κρυφτούν από τους, τις ανταρτικές δυνάμεις που επιτίθενται εναντίον τους. Και υπάρχουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε πάρα πολύ ευρία κλίμακα. Απαγωγές, δολοφονίες, βιασμοί, κακοποιήσεις και στην περιοχή του Μπαγκή για παράδειγμα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Υπάρχει ίσως ε, κάποια έννοια ε, τάξης, ε, εκτός όμως της πρωτεύουσας Μπαγκή έχουν όλα διαλυθεί. Δεν πληρώνονται μισθοί επί μήνες. Υπάρχουν, ας το πω έτσι, υπάρχει προσφυγή των πάντων στο ίδιο το Μπαγκή. Ε, και οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο υπό την αιγίδα ανθρωπιστικών οργανώσεων. Θέλω να επενέσω ε, την ανθρωπιστική κοινότητα διότι πραγματικά παρέχει τη συνδρομή της σε πάρα πολύ ευάλωτες ομάδες ανθρώπων. Παρόλους τους κινδύνους ε, που είναι πραγματικά έντονοι και ιδιαίτερα επικίνδυνοι και δολοφονούνται τα μέλη των οργανώσεων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας εκεί. Και όταν βλέπουμε ποιος είναι ο πυρήνας του προβλήματος, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι απίστευτα επικίνδυνα. Πρώτον, αυτή η χώρα για πρώτη φορά βιώνει διαθρησκευτικές ε, ταραχές και δολοφονίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Φαμπιούς έκανε λόγο για γενοκτονία που είναι ένας πραγματικός κίνδυνος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Μια χώρα όπου συμβίωναν οι άνθρωποι, συνυπήρχαν χωρίς βία ειρηνικά, τώρα έχει διχαστεί μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών και οι περισσότεροι από τους στρατιωτικούς ηγέτες είναι μουσουλμάνοι, πολλοί από αυτούς είναι αλλοδαποί και όλα αυτά η διαθρησκευτική αυτή σύραξη όταν ξεκινήσει μια φορά και ξεσπάσει το γνωρίζουμε από άλλες χώρες, είναι απίστευτα δύσκολο να αναχαιτιστεί και να ακυρωθεί. Το σενάριο λοιπόν αυτό της απόλυτης καταστροφής δεν είναι πλέον υπόθεση εργασίας για αυτή τη χώρα της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας. Τι κάνουμε και τι πρέπει και μπορεί να γίνει. Κινητοποιηθήκαμε ιδιαίτερα έντονα με δραματικό τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει ανθρωπιστική χρηματοδότηση και τώρα δεν είναι πλέον πρόβλημα κονδυλίων ή χρημάτων. Είναι το θέμα της παρουσίας ε, ατόμων επιτόπου με ικανότητες και δεξιότητες να παράσχουν βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Το υπαρχόν ένα πρόβλημα είναι όμως το πρόβλημα της ασφάλειας. Η ασφάλεια μπορεί να ανοικοδομηθεί μόνο με σημαντική αύξηση των ειρηνευτικών δυνάμεων, ενόπλων στρατιωτικών δυνάμεων σε αυτή τη χώρα. Δυνάμεων που θα προστατέψουν τον πληθυσμό αυτής της χώρας από τρόπες πράξεις ε, και πλήγματα πρέπει να έχουν πρόσβαση για να μπορέσουν να παρέμβουν σε ανθρωπιστική βάση αυτοί οι άνθρωποι για να βοηθήσουν τους πληθυσμούς εκεί. Είναι τεράστια σημασία να υπάρξει μια πολιτική διεργασία που θα οδηγήσει σε εκλογές και στην εξομάλυνση της κατάστασης σε αυτή τη χώρα. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να υπάρξει μια ε, εμπλοκή της διεθνούς κοινότητας καθημερινά επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό για τη διεθνή κοινότητα να εμπλακεί, να υπάρξει ένας οδικός χάρτης που θα προβλέπει εκλογές, κοινοβουλευτικές εκλογές ε, το 2015. Και τρίτον, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ε, να μην αυταπατώμεθα επιτρέψαμε <clears throat> η κεντροαφρικανική δημοκρατία να γίνει ένα ορφανό, ένα ε, παιδί το οποίο δεν το πρόσεχε κανείς. Και βλέπουμε ότι η τοποθέτηση αυτή, αυτή η προοπτική πρέπει να αλλάξει. Να αλλάξει ώστε να εμπλακούμε μακροπρόθεσμα και να δεσμευτούμε για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη. Όπως είπε η κυρία Ζολή, η ανάπτυξη, η δυνατότητα ανάπτυξης είναι η καλύτερη δυνατότητα να αποτραπούν καταστροφές, σειράξεις. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τονίζοντας ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θα ήθελα να πω ότι δεν έχει χαθεί ακόμα το θέμα, η υπόθεση αυτή αυτής της χώρας. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και να αλλάξουμε τα πράγματα, να ανατρέψουμε τη σημερινή κατάσταση και να τροποποιήσουμε την κατάσταση των πραγμάτων στο μέλλον. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι μπορώ να σας πω ότι έχουμε δεσμευτεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση και η συνεργασία με την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, μια και το ανέφερα, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω λέγοντα ότι με βάση του πώς εμείς δρούμε και θα δράσουμε με βάση θέματα σειράξεων και συγκρούσεων, πρέπει να καθορίσουμε με κάθε σαφήνεια ποια είναι η θέση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην ευρύτερη, ε, σφαιρικότερη αυτή, ε, στο σφαιρικότερο σκηνικό το οποίο εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλήξαμε στο ότι πρέπει να βρεθεί δυνατότητα εμπλοκής ε, και να βοήθειασε και εκ των έξω η ανθρωπιστική βοήθεια <clears throat> δεν πρέπει να θεωρείται ότι παρέχεται σε ένα ξεχωριστό πλανήτη αλλά επίσης βρισκόμαστε ε, εκτός αυτού του πλαισίου γιατί δεν λαμβάνονται αποφάσεις για την ανθρωπιστική δράση με βάση κάποιο σκεπτικό ε, πολιτικής ε, μεροληψίας ή ιδιοτέλειας. Είμαστε αμερόληπτοι και μπορούμε έτσι να μπορούμε να δρούμε σε περιοχές που κανείς άλλος δεν πάει. Στο βορρά του Μαλή για παράδειγμα ή στις χώρες της Υπέθρου, στις περιοχές της στην κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία ή στη Συρία την ίδια, εντός της ίδιας της Συρίας. Πάμε εκεί όπου δεν πάει κανείς. Και επιπλέον είμαι απόλυτα πεισμένη <clears throat> ότι εγώ δεν θα είμαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου, δεν θα είμαι επίτροπος με αυτό το χαρτοφυλάκι του χρόνου, αλλά είμαι πεισμένη ότι αυτή η προσέγγιση εντός και εκτός, εντός και εκτός υποστήριξης και δράσης είναι αυτό το οποίο μπορεί να, έχει δίνει αποτελέσματα για μας ως υπηαδύναμη. Ευχαριστώ. the of την επόμενη φορά λοιπόν θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη αυτά και θα πρέπει να μιλήσουμε με την κυβέρνησή σας. <laughs> Yeah. The case is the Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι έτοιμη να συζητήσω με την βουλγαρική κυβέρνηση για να κρατήσουμε την κυρία Γεωργίευα στο πόστο της. Σας ευχαριστώ κύριε Γεωργίευα για όλες τις ε, προσπάθειές σας και επιτρέψτε μου να σταθώ λίγο στη χώρα που γνωρίζω καλύτερα, τη Συρία. Έχω δύο-τρεις ερωτήσεις να σας θέσω. Πρώτον, κάτι που μπορεί να σας φανεί χαζό, αλλά αφορά τις στατιστικές των θανάτων και ασθενειών μεταξύ των εκτοπιστέντων και των προσφύγων. Πριν τρεις εβδομάδες πήγα στη Συρία και στο Λίβανο και ρώτησα την ύπατη αρμοστία προσφύγων για τις στατιστικές, κυρίως για την πολιομιελίτιδα και για τις στατιστικές για θανάτους και στη Συρία αλλά και στο Λίβανο. Μας είπαν ότι Κοιτάξτε, είμαστε πνιγμένοι στη δουλειά και δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε στατιστικές. Είναι τρομερό αυτό. Ε, πρέπει να πω ότι φτάνει ο χειμώνα και θα σκοτώσει τόσους ανθρώπους όσους και ο πόλεμος και οι βόμβες. Πρόκειται για μια τέτοια ανθρωπιστική βοήθεια που ακόμα και οι στατιστικές του τι θα συμβούν είναι ε, δύσκολο να τις λάβουμε υπόψη μας. το τι θα συμβεί. Το ίδιο μου είπαν και οι γιατροί χωρίς σύνορα ότι αυτό θα συμβεί παρά τις ανθρωπιστικές καταστροφές, θα να πω ότι έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε τα νούμερα για να βλέπουμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Γιατί θα μπορούσε να μας εντυπωσιάσει η εξέλιξη αυτή. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο ότι η ανθρωπιστική διάσταση δεν είναι πολιτική. Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις άξονες. Καταρχάς είναι ο χημικός αφοπλισμός, με το Γενέβη 2 έχουμε μια μικρή ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει, το ελπίζουμε. Και τρίτον είναι αυτή η διάσταση η ανθρωπιστική. Για αυτό το τρίτο σημείο, την τρίτη διάσταση. Εσείς και η ομάδα σας έχετε δυνατότητα σήμερα να πάρετε θεωρήσεις για, τις, για τη Συρία. Πόσο μπορείτε να δουλέψετε εκεί και για την πρόσβαση που είναι τεράστια δυσκολία. Ποιο μα τρενάρει, ποια είναι η τροχοπέδη, λόγω τη κατάσταση, λόγω τη κυβέρνηση ή λόγω των ανταρτών. Υπάρχουν δύο ομάδε ανταρτών διαφορετικέ στη Συρία και όταν θέλουμε να πάμε σε μια περιοχή όπου βρίσκονται αυτοί, πρέπει να μιλήσουμε και με τους δύο. Αυτό είναι το ερώτημα και ένα τελευταίο ερώτημα, μια και έρχεται ο χειμώνα, στη χρηματοδότηση που προβλέπετε, μέχρι ποιου σημείου δώστε μας μια εκτίμηση, έτσι. Μέχρι ποιο σημείο μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες. Όταν πήγα πιο παλιά, συζητούσαμε για τις οικογένειες που θα βοηθήσουμε και ποιες θα ξεχάσουμε γιατί δεν είχαμε αρκετά χρήματα. Και είδα οικογένειες να μαλώνουν, να τσακώνονται, ενώ δεν είχαν τίποτα μέσα στα στρατόπεδα ε, για την ανθρωπιστική αυτή βοήθεια Μιλάμε για απτά στοιχεία, έτσι, για απτά πράγματα. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για όλα όσα κάνετε. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο κυρία Γεωργίευα για τις προσπάθειές του και για το ότι ήρθε εδώ να μας παρουσιάσει την κατάσταση επιπλέον. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, να κάνω δύο ερωτήσεις σύντομες. Η πρώτη, Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι η μέγιστη χορηγή βοήθειας ε, για την Συριακή τραγωδία. Θα ήθελα να ξέρω ποιες άλλες χώρες καταβάλουν προσπάθειες και ιδιαίτερα αν οι αραβικές χώρες για παράδειγμα που είναι τόσο πλούσιες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία ή τα Εμμυράτα, Αραβικά Εμμυράτα βοηθούν και εκείνα τα κράτη να ανακουφιστεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία. Δεύτερον, μια ερώτηση ίσως πιο πέρα από τις ανθρωπιστικές ανησυχίες που εξέφρασε η Επίτροπος για τις Αρμοδιότητες. νέο κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσία που έχει δημιουργηθεί για την καταστροφή των χημικών όπλων και ένα νέο κλίμα που έχει δημιουργηθεί στη διεθνή κοινότητα με τη συμφωνία ή ε, τις διαπραγματεύσεις στη Γενέβη που προχωρούν με το Ιράν. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν για να βοηθηθεί Πρώτον, ώστε αυτή η συνάντηση στη Γενέβη σε σχέση με τη Συρία να μπορέσει να στεφτεί με επιτυχία και τον Ιανουάριο να μπορέσει να δώσει αποτελέσματα όπως λέγεται και να διευκολυνθούν τα πράγματα για αυτά τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε. Και δεύτερον, για την πρόσβαση, την προσπελασιμότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας εντός Συρίας. Αυτό το νέο κλίμα μεταξύ των, νέων, των υπερδυνάμεων μπορεί να βοηθήσει για αυτές τις προσπάθειες. Όχι μόνο στη διάσκεψη της Γενέβη για να μπορέσει αυτή να ολοκληρωθεί, αλλά και να έχουμε πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στα άτομα που πλήττονται τόσο πολύ στη Συρία. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Σας ευχαριστώ κύριε Επιτρόπε, κυρία Σχάκε και για την ε, καλή σας δουλειά και τη θερμή σας ε, δουλειά. Όπως πάντα, πείτε μας, ε, μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το πιο βασικό εμπόδιο για απόφαση του ψηφίσματο, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ε, πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Επίσης, ε, μπορείτε να μας πείτε τι σας απασχολεί κυρίως ε, σε ό,τι αφορά αυτούς που εργάζονται στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία, σε ό,τι αφορά τα περιστατικά ακραίας βίας και τρίτον, τι περιμένετε από τη Γενέβη σε ό,τι αφορά το ανθρωπιστικό επίπεδο ή μήπως έχετε και άλλες προσδοκίες. Ευχαριστώ. Κυρία Αργεντίνη Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το in but out, κυρία Γεωργίευα. Καλή αυτή η αρχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή όμως αυτή η αρχή, γιατί θέλουμε να ζητήσουμε λύσεις, όχι να παραμείνουμε στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια. Θα προσπαθήσω όμως να τηρήσω αυτή την βασική αρχή ότι δεν θα πρέπει να είναι πολιτική η ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί όταν καταστεί πολιτική δεν μπορεί να επιτελέσει το σκοπό της. Διάβασα ότι επισκεφθήκατε στη Βουλγαρία προσφάτως ε, Σύρους πρόσφυγες. Ε, μιλήσατε για... με Κούρδους, για παράδειγμα, εθνικής καταγωγής Κούρδους. Πείτε μας, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίσει την κρίση στη Συρία σε ό,τι αφορά τον σύνδεσμο μεταξύ Σύρων και Σύρων που φιλοξενούνται σε γειτονικέ χώρες. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε επίσης την τοποθέτηση των Παλαιστινίων Σύρων προσφύγων που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, τρομακτικές καταστάσεις, αύξηση βλέπουμε των Παλαιστίνιων Σύρων που προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κεντροαφρικανική δημοκρατία τώρα. Είπατε ότι θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της κατάστασης και ότι μπορέσουμε να κινηθούμε προς ε, τις εκλογές, προς μια φυσιολογική κατάσταση. Είναι εκπληκτικό αυτό γιατί αυτή η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες επί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Σαλάκα είδαμε πρόσφατα εισήλθε στην πρωτεύουσα και είδαμε πως τα στρατεύματα της Αφρικανικής Δημοκρατίας της ε, Αφρικανικής Ένωσης, συγγνώμη, ε, έκπληκτα και δεν μπόρεσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι μια χώρα που περιτριγυρίζεται από αποτυχημένα κράτη. Και προσφάτως, ναι, ναι, ναι, πρόεδρε, ολοκληρώνω. Πού πιστεύετε ότι βασίζεται αυτή η ιδέα, ότι θα μπορούσε να υπάρχουν εκλογές και μια φυσιολογική υποτυπωδός κατάσταση αρχές του 2015. Αναρωτιέμαι. Ευχαριστώ, κύριε Σάφκιν. Πρόεδρε, μου δέντε το λόγο πριν από τον κύριο Τάνοκ. Φοβερή στιγμή. Σχόλιο εκτό μικροφώνου του Πρόεδρου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Όταν συζητάμε τα θέματα αυτά, πάντα λέω ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμεί πληρώνουμε. Είμαστε payers, όχι players, όχι Φορεί, δηλαδή. Πόσο όμως μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε μόνο ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς να λέμε στα άτομα τα εκάστοτε ότι πρέπει να σταματήσουν. Γιατί άμα το κάνουν δεν πρέπει να συνεχίσουμε να πληρώνουμε. Κοιτάξτε, εμείς ε, το δικό μου το εκλογικό κοινό έχει ε, αγανακτήσει και είναι βέβαιοι ότι βέβαια σε αυτό ισχύει και για άλλους. Πρέπει να υπάρχει ένα quid pro quo ότι αν δεν σταματήσετε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να συνεχίσουμε να σας δίνουμε χρήματα. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Η κυρία Ζολή. I want to thank you very much. Σας ευχαριστώ, κυρία Γεωργίεβα, για την παρουσίαση αυτή της κατάστασης. Τι πιστεύετε για τα κράτη-μέλη που δεν παρακολουθούν ε, τις οδηγίες μας για, τις, ε, για τους πρόσφυγες και ανοίγουν τα σύνορά τους. Για τη Γαλλία που πήρε 250, 250 πρόσφυγες όταν έχουμε 2,5 εκατομμύρια. Ενώ η Γερμανία 6.000, η Σουηδία πήρε 17.000 ενώ είναι λιγότερο από 10 εκατομμύρια. Δεν παραβιάσουμε τις δικές μας οδηγίες για το άνοιγμα των συνόρων μας ενώπιον αυτής κατάστασης. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να μείνω και να επιμείνω στην κατάσταση των προσφύγων, προσφύγων από την Παλαιστίνη. Οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες είναι ήδη εξόριστοι στη δική τους χώρα, από τη δική τους χώρα στη Συρία αυτή τη στιγμή με τις ε, πληροφορίες που έχω βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση για να γίνουν δεκτοί σε οποιαδήποτε χώρα. Δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Παλαιστίνη, δεν μπορούν να επιστρέψουν στο Ισραήλ, δεν τους δέχονται στην Αίγυπτο, έχουν δυσκολίες να πάνε στην Ευρώπη. Γιατί, Γιατί δεν τους θεωρούν ότι έχουν το καθεστώς προσφύγων. Είναι εξόριστοι και δεν είναι πρόσφυγες σαν τους άλλους. Μέσα στη σοβαρότητα αυτής της κατάστασης που πλήττονται όλοι, αυτοί οι εξόριστοι των Παλαιστινίων είναι η σοβαρότητα χειρότερη ίσως περίπτωση και θα θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω βουλγαρικά. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κυρία Γεωργίευα για τις λεπτομέρειες εξηγήσει και για τη σαφή παρουσίαση του προβλήματος της κρίσης στη Συρία και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Είναι πολύ περίπλοκα αυτά τα θέματα και από τη μία χρειαζόμαστε ανθρωπιστική βοήθεια για το λαό της Συρίας προφανώς, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ και σε, άλλα, σε άλλες πτυχές του προβλήματος. Θα ήθελα να μιλήσω για τους πρόσφυγες της Συριακής κρίσης. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε Πώς γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να συντονίζει την οδύσσια των προσφύγων αυτών στο δρόμο προς άλλες χώρες, στο δρόμο που έχουν πάρει για να πάνε σε άλλες χώρες. Πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους πρόσφυγες, πώς θα τους βοηθήσουμε να καταρτιστούν, να εκπαιδευτούν, να φροντίσουν την υγεία τους. Πώς θα βοηθήσουμε τις χώρες οι οποίες επηρεάζονται από τη μεταναστευτική αυτή ροή, από την ροή αυτή των προσφύγων. Είναι κάτι που ξέρουν όλοι, ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν και τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Στις 22 Ιανουαρίου, κυρία Γεωργίευα, Μία αντιπροσωπεία από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ με ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες θα επισκεφτεί τη Βουλγαρία. Και θα πάμε στα σύνορα με την Τουρκία. Θα μπούμε στην Τουρκία επίσης και θα επισκεφτούμε τα στρατόπεδα προσφύγων. Τι θα μας συμβουλεύατε ε, για να επικεντρωθούμε, σε τι να επικεντρωθούμε. Ε, σε τι πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα. Και δεύτερον, μιλήσατε για μια ήπια δύναμη. Μπορούμε να ασκήσουμε ήπια ισχύ εναντίον αυτών που χρησιμοποιούν όπλα. Μπορεί αυτοί να, υποχωρήσουν. Και όταν μιλάω για πίεση μεγάλη και για ισχυρά όπλα, ε, δεν εννοώ μόνο φυσικά την κυβέρνηση, αλλά και τη Ρωσία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε την τραγωδία που εξελίσσεται στην περιοχή, που διαδραματίζεται στην περιοχή. Ευχαριστώ. Η Συρία είναι ένα αποκαρδιωτικό ε, και αξιολύπητο θέαμα ε, ε, στον τύπο μας, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μιλάμε για ελεύθερου σκοπευτέ που στοχεύουν και χτυπάνε παιδιά. Επίσης υπάρχουν ισχυρισμοί ότι ο βιασμό χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου. Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ε, από ό,τι συνέβαινε δύο-τρία χρόνια πριν στην Αφρική. Επομένως η κατάσταση είναι πραγματικά καταθλιπτική. Ο ρόλος της Κίνας και ε, Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι επίσης μια τραγωδία. Ε, γιατί δεν επιτρέπουν ε, την διεθνή κοινότητα να βρει μια λύση. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω ε, αφορά το ρόλο των λεγόμενων φιλικών κρατών και μια υποψήφια χώρα μεταξύ αυτών της Τουρκία, του Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, που δίνουν όπλα και λεφτά στου εξτρεμιστές τζιχαντιστές. Και το, το Ιράκ ας πούμε και του Λιβάνου. Μιλήσατε για την αποσταθεροποίηση ε, του Λιβάνου, αλλά δεν μιλήσατε για την αποσταθεροποίηση που προκαλείται στο Ιράκ, όπου τώρα, ε, λόγω του ότι μπαίνουν όπλα από τη Συρία, ας πούμε, υπάρχει αποσταθεροποίηση. Επίσης, οι χριστιανοί πρόσφυγες από το Ιράκ, που ήρθαν πριν από μια δεκαετία, πήγαν στη Συρία, νομίζοντας ότι θα βρουν εκεί, ε, σε αυτό το μη θεοκρατικό καθεστώς, ας πούμε, όπως το Ιράν, ε, κάποια προστασία. Και τώρα κινδυνεύουν πάλι να σφαγιαστούν από αυτούς τους εξτρεμιστές τζιχαντίστες. Τι πίεση ασκούν τα κράτη-μέλη σε χώρες, όπως αυτές που ανέφερα, για να σταματήσουν να οπλίζουν αυτές τις ακραίες ε, τζιχαντιστικές ομάδες. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Και θα ήθελα να παρουσιάσω ένα προβληματισμό, μια σκέψη. Το σχολίαζε πιο πριν ο συνάδελφος. Κάνουμε λόγο για τα παιδιά, για παιδιά που έχουν ε, αποβιώσει σαν συνέπεια των πολεμικών πράξεων. 800 ε, εκτελέστηκαν, 400 ήταν θύματα ελευθέρων σκοπευτών και έχουμε και δεκάδες ε, που δολοφονήθηκαν ε, και βασανίστηκαν. Είναι συγκεκριμένα θέματα αυτά. Ποιες συγκεκριμένες δράσεις αναλαμβάνουμε εμείς ε, και πρωτοβουλίες έναντι των ανήλικων, για τα ανήλικα παιδιά. Κάνατε λόγο για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την UNICEF. Θα ήθελα να ξέρω τι συγκεκριμένα γίνεται. Επίσης να μας ενημερώσετε για τον έλεγχο μιας οδού για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μεταξύ Μασκού και Χόμς ε, στην περιοχή Κουαλαμών. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται σε σχέση με την παροχή βοήθειας ε, λόγω του ελέγχου των ε, κυβερνητικών σε αυτή την δίωδο. Από την άλλη πλευρά για την κεντροαφρικανική δημοκρατία δεν μπορούμε παρά να συγχαρούμε και να επενέσουμε τη δράση σας σε μία από τις πιο δραματικές κρίσεις που ωστόσο όμως από την συνάντηση που είχαμε τον, η Επιτροπή Ανάπτυξης μπορεί να μας πει ποια σχέδια ανάπτυξης σχεδιάστηκαν για την την αποκατάσταση και παγίωση, εμπέδωση της κρατικής εξουσίας. Εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βοηθήσαμε να γίνει γνωστή η κατάσταση εκεί. Το εγγράψαμε στις ημερήσεις διατάξεις μας, στις εργασίες μας με τους Αφρικανούς εταίρους μας. Αλλά έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά δεν επαρκούν. Υπάρχουν δυσκολίες ε, και γνωρίζετε ότι παρόλες τις δυσκολίες μπορείτε να βασίζετε σε εμά ε, για την υποστήριξη που μπορούμε να δώσουμε για την επίτευξη μεγαλύτερων αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ που μου δίνει το λόγο, κύριε Χάουιτ. Σε ό,τι αφορά τα αραβικά κράτη, να πάω λίγο παραπέρα από την κυρία Σάκη και από τους υπόλοιπους ε, ομιλητές. Τι μόχλευση προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ό,τι αφορά τα χρήματα που δαπανούμε, σε ό,τι αφορά και τους άλλους δωρητές, σε ό,τι αφορά την τήρηση των δεσμεύσεων. Πριν από κάποιες εβδομάδες αναφέρθηκε ότι το UNHCR παίζει σημαντικό ρόλο και έγινε μια σημαντική συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς πήγε λοιπόν αυτή η συνάντηση για την ανθρωπιστική πρόσβαση τώρα. Ακούσαμε τι είπατε για τα ψηφίσματα. Μεγάλη όμως απόσταση υπάρχει από τα ψηφίσματα και την πραγματικότητα από το τι γίνεται στο επιτόπου. Πείτε μας λοιπόν, στην πράξη υπάρχει ένα ολόκληρο κοινό που παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση. Τι γίνεται λοιπόν με την ε, ανθρωπιστική αυτή βοήθεια, πώς μπορεί να καταστεί πιο αποτελεσματική σε ό,τι αφορά επίσης τους Παλαιστινίους προσφύγους. Προσφάτως ακούσαμε ότι η Αλκάιντα τους απασχολεί πιο πολύ από κάθε τι άλλο σε ό,τι αφορά την ειρηνική τους επιβίωση. Δεν προσπαθώ να σας κάνω να προβείτε σε πολιτικά πολιτικές δηλώσεις, αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε, όπως είπε και ο συνάδελφος, από πού προέρχεται η απειλή στη Συρία. Σχολιάστε σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, το λόγο έχει επίτροπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Και πιο πολύ για το γεγονός ότι καταδεικνύεται τη δέσμευσή σας και αυτό είναι απαραίτητο δεδομένη της δραματικής ε, κρίσης στην Συρία αλλά και σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία στο, στην καρδιά της ε, Αφρικής σε μια ευάλωτη και δεύτερη περιοχή. Να προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Οματοποιώντας τες και οι συνάδελφοι εδώ θα ε, βεβαιωθούν ότι δεν θα ξεχάσω τίποτε. Για να μην απαντάω σε κάθε έναν ξεχωριστά, δεν έχουμε και πολύ χρόνο άλλωστε. Καταρχάς, για το ερώτημα του τι γνωρίζουμε για τις εξελίξεις στη Συρία. Αν θέλετε να κλείσετε το μικρόφωνο, ρωτάει η κυρία Ντεκάιζερ, ζητάει η κυρία Ντεκάιζερ στον πρόεδρο. Okay. Okay. Perhaps it, it is being picked up by my, my mic. Ο κύριος Χόιτ λέει ο πρόεδρος, ίσως έχει μικρόφωνο ανοιχτό. So first on what is what what we know about the Καταρχάς, λοιπόν, τι ξέρουμε για τις εξελίξεις ε, στην ε, Συρία, στο ιστορικό της Συρίας. Ε, πόσο καλά και ακριβή και καλά είναι τα στατιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τις πιο δραματικές κατηγορίες του πληθυσμού, σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες εκείνες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η έλλειψη τέτοιων στοιχείων τι σημαίνει ότι τα στοιχεία που συλλέγουμε δυστυχώς δεν είναι ούτε πλήρη ούτε ακριβή απαραίτητα γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι έχουμε 18 περιπτώσεις πολιομιλίτιδας, αλλά δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν περισσότερες ε, τέτοιες περιπτώσεις ε, που δεν έχουν αναφερθεί, επειδή ολόκληροι πληθυσμοί βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει απαραίτητα πρόσβαση. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μηχανισμό συντονισμού των πιο βασικών οργανώσεων που παρέχουν βοήθεια στο ιστορικό της Συρίας αλλά και στις γειτονικέ ε, περιοχές προκειμένου να σχηματίσουμε μια όσο πιο ολοκληρωμένη εικόνα γίνεται για τον πληθυσμό που αντιμετωπίζει κινδύνους σε ό,τι αφορά τα είδη κινδύνων και επίσης σε ό,τι αφορά τη βοήθεια που διοχετεύεται και μέσα από ποιες οδούς διοχετεύεται. Η... Εμάς στην Επιτροπή μας αναφέρθηκε, κοιτάξτε, προσπαθούμε να ε, συνενώσουμε και να συντονίσουμε τους βασικούς εταίρους για την πιο συστηματική συλλογή πληροφοριών για τα προβλήματα και για τα βήματα που γίνονται για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά σε μια συνάντηση που θα τις οποίες θα προεδρεύσω στις 18 Δεκεμβρίου και θα ακολουθήσει και ακρόαση στο Κοινοβούλιο με τους βασικούς φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας, θα εξετάσουμε ακριβώς τα θέματα αυτά. Άσφαλος μας ανησυχεί ιδιαίτερος ο κίνδυνος που πλήττει τους πλέον ευάλωτους και ενδεχομένως να ε, ε, επιμολύνει και την υπόλοιπη περιοχή. Πανδημία πολυμελίτιδας και άλλες πανδημίες το υγειονομικό σύστημα στη Συρία έχει καταρρεύσει. Ένα παράδειγμα να σας δώσω κάποιες παραμέτρους και μόνο που καθορίζουν το ότι δεν υπάρχει πλέον υγειονομικό σύστημα σε μια χώρα που ήταν σχετικά καλή σε ό,τι αφορά τις ε, κοινοφιλείς υπηρεσίες. 15.000 γιατροί έχουν φύγει από τη Συρία. 92% των ε, ασθενοφόρων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έχουν καταστραφεί δύο τρίτα τουλάχιστον των υγειονομικών εγκαταστάσεων σε διαφορετικούς ε, βαθμούς ε, έχουν καταστεί τελείως ε, άχρηστες. Και αν δεν υπήρχε η ανθρωπιστική κοινότητα για να παράχει, παρέχει, παρέχει, παρέχει υπηρεσίες, θα ήταν τραγική η κατάσταση. Θα υπήρχε ασφαλώς και υπάρχει κίνδυνος υπάρχει κίνδυνος διάρειας μεταξύ των ε, παιδιών ή άσημων ασθενειών, επειδή υπάρχει η ασημων ασθενειων επειδη υπαρχει μολυνση του πόσιμου νερού. Τώρα να απαντήσω το, τι κάνουμε ιδιαίτερα για τα παιδιά. Το θέσατε το ερώτημα αυτό. Η εταιρική σχέση που έχουμε συνάψει με την UNICEF μας έχει οδηγήσει στο να ορίσουμε τέσσερις βασικές δράσεις σε ό,τι αφορά τα παιδιά λεπτομερέστατα σε ό,τι αφορά, βάση, σε ό,τι αφορά προσέγγιση βάση της χώρας, της και για τη Συρία και για το εξωτερικό της Συρίας. Ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν ειδική παροχή βοήθεια για τα παιδιά, σε θέματα ε, εμβολιασμού, θέματα ε, σύντησης των πιο ευάλωτων παιδιών, επίσης προστασία και εκτός της Συρίας για να προστατεύσουμε τα παιδιά από την βία και κατά της πορνείας και λυπάμαι που χρησιμοποιώ αυτή την φρεχτή λέξη σε ό,τι αφορά την προστασία των παιδιών από κυκλώματα σκλαβιάς, ουσιαστικά εργασίες με πολύ πολύ χαμηλούς μισθούς. Κατά τρίτον, πρόσβαση στην εκπαίδευση. Είναι πολύ βασική αυτή η πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα παιδιά στο εσωτερικό της Συρίας αλλά και στις γειτονικές όμορες χώρες. Και κατά τέταρτον, οι νεολαίες στη Συρία, τα νέα αυτά άτομα που θα κληθούν να ανοικοδομήσουν τη Συρία όταν τελειώσει αυτή η κατάσταση. Και ο κίνδυνος της ε, ριζοσπαστικοποίησης των ατόμων αυτών. Σε αυτούς τους τομείς λοιπόν έχουμε διαμορφώσει μέτρα τα οποία έχουν αξιολογηθεί γύρω στο 1 δισεκατομμύρια δολάρια για τους επόμενους 18 μήνες. Αυτό χρειάζεται προκειμένου. Και στην επόμενη συνάντηση θα συζητήσουμε το θέμα αυτό ενδελαχέστερα σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα για τα παιδιά. Να δούμε Ποιο μπορεί να κάνει και τι. Πώς μπορούν να δεσμευτούν και οι διάφορες οργανώσεις παροχής ε, βοήθειας. Να περάσω τώρα σε ένα δεύτερο, σε μια δεύτερη ομάδα ερωτήσεων. σε ό,τι αφορά τη συλλογή πόρων και στην κατανομή των ευθυνών. Τι κάνουμε από πλευρά της Ευρώπης. Δύο πράγματα. Αφενός, δίνουμε ένα παράδειγμα, αλλά και χρησιμοποιούμε το παράδειγμα αυτό για να ασκήσουμε πίεση στους άλλους να διαδραματίσουν το ρόλο τους και και με ορατό τρόπο και με διακριτό τρόπο αλλά και με πιο διακριτικό τρόπο προσπαθώ να απευθυνθώ στις χώρες του Πρεσικού κόλπου, στη Ρωσία, στην Κίνα να τις καλέσω όλες αυτές τις χώρες προκειμένου να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην παροχή βοήθειας προς τη Συρία και στις γειτονικές χώρες. Κάποιες φορές ε, είναι επιτυχής αυτή η δραστηριοποίησή μου, κάποιες άλλε όχι. Να σας πω ένα παράδειγμα επιτυχέ με το Κουβέιτ. Καταφέραμε το Κουβέιτ να δραστηριοποιηθεί πολύ πιο έντονα και μάλιστα με διαφανή τρόπο μέσω του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε την αίσθηση ότι δεν ε, εισακούομεθα. Να σας βεβαιώσω όμως ότι θα συνεχίσουμε να ζητούμε κινητοποίηση σε χώρες της περιφέρειας. Είμαστε ηγετικοί, ξέρετε, φορείς, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα χρήματα, αλλά και σε ό,τι αφορά το να προλαμβάνουμε τι θα συμβεί. Είμαστε οι πρώτοι που κινηθήκαμε και παρήχαμε βοήθεια και είπαμε ότι δεν βοηθούμε αρκετά από τους πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες. Να σας ε, ευχαριστήσω που αναφέρετε το Ιράκ, γιατί το Ιράκ αντιμετωπίζει μεγάλο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά 200.000 ε, πρόσφυγες που έχουν λάβει από τη Συρία και σε ό,τι αφορά την ε, ροή όπλων που προέρχεται από την σύραξη στη Συρία. Ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι είναι η ύψη της σημασίας να βοηθήσουμε τις χώρες που αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, αντίκτυπο από τη σύγκρουση αυτή. Κινητοποιήσαμε τον προϋπολογισμό από το Ταμείο Γειτονία για τις χώρες αυτές. Και... Κινητοποιήσαμε κονδύλια, ασκήσαμε πίεση ώστε να υπάρξει υπευθυνότητα και υπεύθυνη εμπλοκή σε αυτή την περιοχή του κόσμου από πλευράς μας. Και είδαμε τα ωφέλη αυτού του είδους δράσης και άσκησης πίεσης. Και μια και είμαι και αναφέρομαι στο θέμα των επιπτώσεων στις γειτονικέ χώρες γύρω από τη Συρία, ας απαντήσω στις παρεμβάσεις των δύο Βουλγάρων Ευρωβουλευτών αλλά και άλλων που έθεσαν και έθιξαν το θέμα της επίπτωσης αυτής της κρίσης στην ίδια την Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνουν όλα αυτά όσον αφορά ροές προσφύγων, κινδύνων. Ποιες είναι οι απαντήσεις από πλευράς Για τώρα, προς το παρόν, μέχρι σήμερα η ροή προσφύγων προς την Ευρώπη από τη Συρία βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα δεδομένου του πληθυσμού των ε, προσφύγων από αυτή τη χώρα συνολικά. Σήμερα έχουμε περίπου 55.000 Σύριους στην ε, Ευρώπη, έναντι 2,3 εκατομμυρίων προσφύγων από τη Συρία στις γειτονικές χώρες γύρω από τη Συρία. Όμως η τάση ποια είναι. Η τάση είναι και επιτρέψτε μου να το πω αυτό ξεκάθαρα, ανοιχτά και ε, ανυπόκριτα. Όταν επενδύουμε για να βοηθήσουμε τη Συρία, τους πολίτες της Συρίας και τους γείτονες της Συρίας. Επενδύουμε επίσης στη μείωση των κινδύνων ενός προ, ε, κύματος προσφύγων από εκεί προς την Ευρώπη. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη δήλωση. Τώρα όμως υπάρχουν αρκετοί που έρχονται, προσέρχονται στην Ευρώπη και έχουμε μια πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί. Διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση αυτών των ετούντων άσυλο. Κάποιες χώρες είναι πιο ανοιχτές. Η Σουηδία. Αναφέρατε τη Σουηδία, αλλά ουσιαστικά και η Γερμανία. Η Γερμανία επιπρόσθετα σε αυτού ε, που άνοιξαν τι θύρε του ε, για του πρόσφυγε, 14.000 ε, πολίτε τη Συρίας δέχτηκε η Γερμανία. Για την επανένωση οικογενειών, άλλων που προσήλθαν στη Γερμανία για προστασία. Αυτή η σημαντική όμω διαφορά στην προσέγγιση από χώρα σε χώρα του προβλήματο των ετούντων ασύλων, των προσφύγων συνολικά, είναι ένα ζήτημα το οποίο εγώ πιστεύω πρέπει να αντιμετωπιστεί και να επιληθεί. Δεν είναι βέβαια δική μου δουλειά. Είναι τη Επιτρόπου Σεσίλια Μάλστρομ που πρέπει εκείνη να επιληθεί και των Υπουργών Εσωτερικών ε, του Συμβουλίου, των κρατών μελών να δράσουν. Όμως το λέω αυτό, μια και αναφερόμαστε σε διαφορετικό επίπεδο για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, σας λέω, δεν υπάρχει τρόπος να αποφευθεί η αύξηση του, της ροής των προσφύγων από τη Συρία στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να αποφευθεί αυτό. Η πίεση στις γειτονικέ χώρες είναι τόσο δραματικής μορφής, ώστε οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι όροι και προϋποθέσεις ε, για τη διαβίωση αυτών των προσφύγων στις γειτονικέ χώρες επιδεινώνονται. Για κάποιους από αυτούς τους πρόσφυγες είναι απάνθρωπες αυτές οι συνθήκες. Τι κάνουν λοιπόν. Αν εσείς βρισκόσαστε σε ένα πρότυπο κατάστασης, ε, σε μια τέτοια με συγχωρείτε, κατάσταση όπου τα παιδιά σας θα αντιμετώπιζαν κίνδυνο να αποβιώσουν, τι θα κάνατε. Θα τρέχατε να ξεφύγετε, να αποδράσετε, να βρεθούν ε, τα παιδιά σας, οι οικογένειές σας σε ασφάλεια. Αυτό είναι το θέμα που όλο και περισσότερο θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση από τις ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του προβλήματος των προσφύγων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το έμαθα αυτό εξετάζοντας τα πράγματα. Πέρυσι είχαμε περίπου 100.000 πρόσφυγες ετούντες άσυλοι που πήραν, χορηγήθηκε άσυλο σε αυτούς. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. 60% από αυτούς πήγαν σε πέντε χώρες. Γερμανία και Σουηδία που προαναφέρθηκαν, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Βέλγιο. Αυτές ήταν οι πέντε αυτές χώρες. Και ένας πολύ μικρός αριθμός πήγαν σε χώρες που δεν είχαν παράδοση σχετική και δεν είχαν εργαστεί για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των ετούντων άσυλο σε, αυτό, σε αυτά τα επίπεδα. Έτσι λοιπόν, σε σχέση με αυτό το ζήτημα, είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμός, περισσότερο συντονισμένη προσπάθεια από την Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε μια κρίση που θα μας συνοδεύει και θα ε, έχει δραματικές διαστάσεις και στο μέλλον. Πώς να βοηθηθούν τώρα αυτές οι χώρες για την υποδοχή των προσφύγων. Έχει μέσα και εργαλεία η Ευρωπαϊκή Ένωση και παροχή βοήθειας και παροχή βοήθειας για την επιτήρηση των συνόρων με καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο παρέχεται αυτή η βοήθεια στη Βουλγαρία για την επιτήρηση των συνόρων της για παράδειγμα. Αλλά το μεγαλύτερο κέρδος θα ήταν μια κοινή πολιτική, μια κοινή προσέγγιση από τις ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια πιο ισοδίκαια ε, προσέγγιση και κατανομή επιμερισμό των προσπαθειών για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πολύ δύσκολο, πολύ σκληρό, δύσκολο αυτό το πρόβλημα. Μια και στις χώρες μας, σε πολλές από τις χώρες μας Πέντε χρόνια ύφεση και κρίσης ε, έχουμε περάσει με αύξηση της ανεργίας ε, των Ευρωπαίων πολιτών στις χώρες που έχουν πληγεί υπάρχει όλο και μεγαλύτερη εχθρότητα από πλευρά των πολιτών μας στις χώρες μας έναντι των προσφύγων, αλλοδαπών, μεγαλύτερη ξενοφοβία. Είναι γεγονός αυτό. Το πώς θα δημιουργηθεί μια κοινή πολιτική μέσα σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι εύκολο ερώτημα να απαντηθεί. Όμως είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ούτως ή άλλως, το δυνατόν ταχύτερα. Και πάλι βλέποντας ε, και πιο πέρα για αυτά τα θέματα, τώρα είναι η χρονική στιγμή. Τώρα είναι η χρονική στιγμή να δράσουμε. Δεν πρέπει να πιαστούμε απροετοίμαστοι και ανέτοιμοι. Το καλό είναι ότι υπάρχει μια task force, μια ομάδα κρούσης που εργάζεται για αυτά τα θέματα και συντονίζει. Είναι καλό να θυμόμαστε και να σκεφτόμαστε ότι μετά από την κρίση της Ιουγκοσλαβίας, της κατάρρευσης της Ιουγκοσλαβίας, δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο, ένα σχέδιο δράσης στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση μαζικών ροών προσφύγων. Είναι σημαντικό να ε, χτίσουμε σε αυτά τα θεμέλια και με βάση αυτή την πείρα να προχωρήσουμε. Επειδή όμως είμαι υπερήφανη που είμαι Ευρωπαία, πρέπει να προσθέσω κάτι. Καμιά φορά αφήνουμε να καθοριστούμε εμείς και η ταυτότητά μας από άλλους με τους χειρότερους όρους και με όρους που κυλιδώνουν και υποτιμούν αυτό που είμαστε και κάνουμε. Η Ευρώπη είναι πιο ανοιχτή για την υποδοχή προσφύγων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ήπειρο μεταξύ των ε, βιομηχανικών χωρών. Είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί εμείς οι Ευρωπαίοι. 80-90% προσφύγων πάνε από μια φτωχή χώρα σε μια άλλη φτωχή χώρα που είναι η γειτονική τους χώρα. Από τους 10-20% ε, που απομένουν 74% πάνε στην Ευρώπη μαζικά. 65% έρχονται, προσέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν μας καθορίζουν και λένε ότι είμαστε το φρούριο, το οχυρό της Ευρώπης, δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό για μας τους Ευρωπαίους. Δεν, αντα, δεν αντανακλά την πραγματικότητα της Ευρώπης. Αλλά η, δική μου, ας το πω αρμοδιότητα ε, και η δική μου εικόνα δεν μπορεί να συμπίπτει με αυτή την αρνητική εικόνα που δίνεται καμιά φορά. Δεν μπορώ να πω ότι ταυτίζομαι με τέτοιου είδους προσδιορισμούς. Μία άλλη πτυχή για τα θέματα προσφύγων και να πω στον κύριο Ευρωβουλευτή ε, σε σχέση με την ε, Βουλγαρία τον ε, Ιανουάριο είναι πολύ σημαντικό να δει κανείς πώς συνεργάζονται περισσότερο αυτές οι χώρες μια και αφορά ένα κοινό ζήτημα μεταξύ τους, ένα ευρωπαϊκό κοινό ζήτημα. Τι μπορεί να γίνει για να υπάρξει μεγαλύτερο αποτέλεσμα μεγαλύτερος εξοπλισμός, περισσότερες δυνατότητες για τον καθορισμό τριών κατηγοριών πολιτών που περνούν τα σύνορά μας. Αυτούς που είναι πραγματικοί, αυθεντικοί πρόσφυγες θέλουν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους, πρέπει να προστατευτούν. Οι άλλοι είναι οικονομικοί μετανάστες, δεν ε, διαφεύγουν από ένα πόλεμο, δεν είναι λοιπόν πρόσφυγες, δεν έχουμε καμιά υποχρέωση ε, να τους προστατέψουμε έναντι των άλλων. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος μικρός αριθμός ε, που μπορεί να αποτελούν, να έχουν ένα κίνδυνο ασφάλειας. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ξεχωριστά αυτές τις τρεις κατηγορίες με το σωστότερο τρόπο, όχι να τις αναμειγνύουμε και να τις συγχαίουμε και να μην έχουμε θετικά αποτελέσματα στις πολιτικές μας να διαφοροποιούμαστε. Και φυσικά όταν κάνουμε λόγο για πρόσφυγες, επιτρέψτε μου να πω, ολοκληρώνοντας αυτό το τμήμα των θεμάτων, με τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες να ολοκληρώσουμε. Πράγματι, η πιο ευάλωτη, εύτρωτη κατηγορία είναι εκείνη, επειδή είναι διπλά, διτά πρόσφυγες οι Παλαιστίνοι και έχουν πάρα πολύ περιορισμένες επιλογές. Ή μένουν στη Συρία όπου ουσιαστικά από, ε, προσελκύονται και στρατολογούνται από τις ε, ε, αλληλοσπαρασόμενες ομάδες σε αυτή την εθνοσύραξη ή πάνε στο Λίβανο όπου επιτρέπεται με να εισέλθουν αλλά κάτω από φρικτές συνθήκες να περάσουν στο Λίβανο ή αναζητούν τρόπους να περάσουν στην ε, ε, Ευρώπη. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί με την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους ε, πρόσφυγες και την συνεργασία μας για την συνδρομή σε σχέση με τους πρόσφυγες και αυτά τα άτομα. Είναι όμως άτομα που έχουν πληγεί με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο. Επόμενο θέμα. Τι γίνεται με το γεωπολιτικό περιβάλλον. Ποιες είναι οι προσδοκίες μας, τι αναμένουμε από την ε, συνδιάσκεψη Γενέβης 2 των ειρηνευτικών ε, διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων. Πώς μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, να ενεργοποιηθούμε πιο αποτελεσματικά. Για τη Γενέβη 2 λοιπόν, προφανές είναι ότι πρέπει να αναζητήσουμε, να προχωρήσουμε στη Γενέβη 2 με ένα ανοιχτό πνεύμα και να υποστηρίξουμε με αυτόν τον τρόπο ενεργά την ειρηνευτική διαδικασία. Όμως δεν είναι δεδομένο ότι όταν θα συνέρθουν τα εμπλεκόμενα μέρη θα καταφέρουν να καταλήξουν γοργά σε μια συμφωνία ειρήνευσης. Δεν είναι δεδομένο. Και αν καταλήξουν σε μια συμφωνία ειρήνευσης δεν θα είναι εύκολο να υλοποιηθεί αυτή ενδεχόμενα. Εντάξει, μέσα σε αυτό η προοπτική σε σχέση με το Ιράν διαγράφεται ίσως, είναι μια θετική εξέλιξη για τη Συρία, το πρόβλημα της Συρίας επειδή είναι μια δύναμη, μια ισχυρή, ε, ένας ισχυρός παράγοντας ε, ε, το Ιράν έναντι της Συρίας. Και αν θέλουμε να είναι μια δύναμη, μια ισχύς που θα ασκήσει την επιρροή της θετικά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τα πράγματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό, αναμένουμε να το δούμε πώς θα μπορέσει να γίνει. Για την πρόταση ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών, γιατί υπάρχει στεναρή βούληση να εγκριθεί και να προαχθεί. Ο κύριος Χόουτ είναι εκείνος ο οποίος το είπε ότι το ίδιο το ψήφισμα δεν αξίζει δεκάρα αν δεν υλοποιηθεί χειροπιαστά. Είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του. Διότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο των ε, χημικών όπλων και πρέπει να ε, δράσουμε αποτελεσματικά. Λοιπόν, ωραία, λέει η κυρία ε, Γεωργίευα. Θα επιταχύνω για να, να ολοκληρώσω. Θα πατήσω τον γκάζι για να πάω πιο γρήγορα. Λοιπόν, επιταχύνω. Το θέμα ποιο είναι. Έχουμε μία αντιμετώπιση χημικών όπλων <clears throat> ως απειλή, αλλά δεν τη χάνουν της ίδιας αντιμετώπισης τα νέα όπλα και εκείνα τα οποία φωνεύουν διαρκώς όλο και περισσότερους αμάχους. Είναι λοιπόν πολύ ε, άδικο να σκοτώνονται οι άμαχοι. Το ίδιο όμως άδικο είναι να χρησιμοποιούνται και χημικά όπλα. Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία όπου το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ δεν καταδίκασε τις δολοφονίες των πολιτών, των αμάχων και των ε, υπαλλήλων και συντελεστών των ανθρωπιστικών ε, οργανώσεων που δολοφονούνται εκεί. Όμως όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα για την πρόταση ψηφίσματος και πρέπει να υλοποιηθεί το ψήφισμα. Αυτό μας φέρνει στους μεγάλους παίκτες αυτού του θέματος. Πρέπει να τεθούν τα ζητήματα αμφωτέρωθεν. Ποια θα είναι η πίεση και τι σημαίνει να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση και προσπελασιμότητα να υπάρχει δυνατότητα να έχει θεωρήσεις διαβατηρίων οι υπάλληλοι και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο σε πολύ ευρύτερη κλίμακα. Ναι, είδαμε μικρές βελτιώσεις, αλλά πόρο απέχουν από το αναγκαίο πλαίσιο. Πρέπει να υπάρξει δυνατότητα εφοδιοπομπών, ανθρωπιστικής βοήθειας. Μπορούμε να έχουμε ένα οδικό χάρτη που θα καθορίζει τις διαδρομές για αυτές τις εφοδιοπομπές. Θα πρέπει διαζώσεις ξεκάθαρα να τοποθετηθούμε και να λέμε όταν σκοτώνονται άμαχοι γυναίκες παιδιά, άμαχοι. Αυτό θα έχει επιπτώσεις. Θα τιμωρηθούν, θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι αρμόδιοι και θα ε, υποστούν τις ε, ε, ποινές που πρέπει να επιβληθούν. Μέχρι σήμερα γίνονται πολύ λίγα. Ευελπιστώ λοιπόν να δούμε ότι θα υπάρξει μια αλλαγή της δυναμικής μεταξύ των, της στάσης των μελών της ασφάλειας, ε, ε, Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ας περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις που θα σημειωθούν, τι θα γίνει στη Γενέβη όταν ε, ξεκινήσει ο γύρος Γενέβης 2. Τώρα, ξέχασα κάτι για τη Συρία. Ωραία, ας περάσω τώρα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία λοιπόν. Το κύριο ερώτημα εδώ είναι <clears throat> γιατί πιστεύω ότι υπάρχει κάποια ευκαιρία, μια ελπίδα για την κεντροαφρικανική ε, δημοκρατία και δεν εγκαταλείπω τις ελπίδες μου. Είναι μια σχετικά μικρή χώρα. Που ακόμα δεν έχει περάσει σε, μια, σε ένα πλήρη θρησκευτικό πόλεμο. Εάν έχουμε ειρηνευτικές δυνάμεις παρούσες, θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την ειρήνη στον πληθυσμό. Εκεί που είναι σήμερα οι δυνάμεις αυτές, ε, οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές από τις περιοχές που δεν έχουμε ειρηνευτικές δυνάμεις. Υπάρχει θέμα λοιπόν κινητοποίησης, αλλά κινητοποίηση πρέπει να γίνει τώρα. Το δεύτερο, που μου δίνει ελπίδα είναι ότι οι όμορες χώρες είναι πολύ ασταθείς. Αλλά το Τσάντ, το οποίο έπαιξε περίεργο ρόλο απέναντι στην κεντροαφρικανική δημοκρατία, είναι αποφασισμένο να βοηθήσει. Και άλλες αφρικανικές χώρες που ανησυχούν για την περίπτωση του να γίνει χώρα αυτή μια νέα Σομαλία με τον κύριο Φαμπίου και με τη Βαλερία Άμος κάναμε μια συζήτηση για την κεντροαφρικανική δημοκρατία στη Νέα Υόρκη. Και οι αφρικανικές χώρες είδαμε, ε, η Μπραζαβίλ το, του Κόγκο και το Τσάντ προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα. Συναντήθηκα με προσωπικότητες από την περιοχή και έχω την αίσθηση ότι πιστεύουν πως αν αφήσουμε μόνη τη χώρα θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά αν η διεθνής κοινότητα ανασκουμποθεί, θα ανατραπεί η κατάσταση και θα έχουμε θετική εξέλιξη όπως το Μαλί. Δεν πρόκειται να είναι εύκολη κατάσταση. Δεν πρόκειται η ειρήνη να έρθει μόνο μιας, αλλά οι προοπτικές των εκλογών ε, τον Ιανουάριο του 2015 δεν είναι μία φαντασιοπληξία. Εάν δεν βάλουμε ειρηνευτικές δυνάμεις γρήγορα στην ε, χώρα, τότε μπορεί να χάσουμε άπαξ και διαπαντός ε, το ενδεχόμενο σταθεροποίησης. Όταν ταξιδεύεις στη χώρα, διαπιστώνεις ότι η καλοσύνη είναι στην κουλτούρα του λαού. Ε, υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών, αλλά δεν μιλάμε για μια κατάσταση που έχει ξεφύγει τελείως. Δεν μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ας ανθρώπους που συγκρούονται. Σας ευχαριστώ όλους που με ανεχτήκατε. Μίλησα 27 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Ήμουνα αρκετά αναλυτική, αλλά τα θέματα είναι τεράστια, το διακύβευμα είναι φοβερό και άξιο της προσοχής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε, που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας ε, μαζί μας. Όχι μόνο τις σκέψεις σας, αλλά και τις γνώσεις σας, το όραμά σας και τις ανησυχίες σας. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε για να συνεχίσουμε με ψήφισμα και να προτάσουμε αυτό το θέμα και να προσπαθούμε να αναζητήσουμε λύσεις. Ο πίνακας που μας τη για τη Συρία και για την κεντροαφρικανική δημοκρατία είναι πραγματικά ζωφερός. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους και καλό σας βράδυ.